Καλημέρα σας. Αν θέλετε, καθίστε για να ξεκινήσουμε. Διότι έχουμε μια κάπως ε, φορτωμένη για τον πρόεδρο ημερήσια διάταξη, με πολλούς σπουδαίους ομιλητές. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους. Παρακαλώ καθίστε. Uh, because, um, it be δεν θα να βιαστούμε. Δεν με ακούτε. You can't hear me. Um, you can, yes. Uh, there is interpretation. Ωραία. Υπάρχει διερμηνία εξ όσων γνωρίζω σχεδόν σε όλες τις γλώσσες που ελπίζουμε ότι θα μιληθούν. Χρησιμοποιήστε λοιπόν τα ακουστικά σας και βρείτε το κανάλι που θέλετε να ακούτε. Θα δουλέψουν σκληρά οι διερμηνείς σήμερα το πρωί, ως συνήθως γιατί το πρόγραμμά μας είναι εντατικό. Σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής της Προστασίας των Καταναλωτών και της Εσωτερικής Αγοράς στην ακρόασή μας σήμερα το πρωί. Είναι η δεύτερη ακρόαση που οργανώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια για την τυποποίηση και νομίζω πολλοί από εσάς συμμετείχατε και στην πρώτη από αυτές. Όταν είδαμε για άλλη μια φορά τις προδιαγραφές και τα πρότυπα, εν αναμονή μια της νομοθετικής πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόταση που επικαιροποίησε το νομοθετικό πλαίσιο για την τυποποίηση. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να δούμε τις λεπτομέρειες αυτών των εξέλιξεων. Και εδώ καλωσορίζω την πολύ σκληρά εργαζόμενη αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας, την κυρία Λαρακόμη, που είναι η για την Επιτροπή μας για το πρόγραμμα των προδιαγραφών εδώ υπάρχουν και πολλοί σκεώδεις εισηγητές, η κυρία Σαλτεμόζε, η κυρία Ρίλε, ο κύριο Μέκ, η κυρία Μάγερ και επίσης καλωσορίζω και τον κύριο Κύριεκ, ο οποίος εκπροσωπεί την Επιτροπή Βιομηχανία και τον κύριο Προύστ που ετοιμάζει γνωμοδότηση για την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Και οι δυο είστε καλοδεχούμενοι, ενώ από τα εθνικά κράτη, επειδή έχουμε πολλέ ομιλίε και παρεμβάζει το θέμα αυτό, έχουμε επίση πολλού συμμετέχοντε. Λοιπόν, θα περιμένουμε να ακούσουμε τι συνεισφορέ όλων. Τώρα, να θυμίσω ότι εδώ περνάμε και στο διαδίκτυο και από την προηγούμενη ακρόασή μα ξέρουμε ότι πολλοί είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για τι προδιαγραφέ και τα πρότυπα και πολλέ επιτροπέ ανά τον κόσμο, εκτό τη Ευρώπη, παρακολούθησαν, άκουσαν την ακρόασή μα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους όσους, όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο και σας ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας για την ανάπτυξη των προτύπων γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι που απασχολούνται σε φορείς που εξετάζουν την τυποποίηση ανά την Ευρώπη και τον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ακρόαση και θα καλέσω τον κύριο Γκυρέκ και τον κύριο Προύστ να μας Κάνω κάποια σχόλια, σύντομα σχόλια, τη δική τους άποψη για το θέμα. Να καλωσορίσω την κύριο Κρέσπο, την κυρία Μπρίκμαν και την ομάδα της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι όλοι μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε κι εσείς. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο και μετά θα περάσουμε στην ακρόαση αυτή καθ' αυτή καλωσορίζοντας και τους ε, εξαιρετικούς μας ομιλητές. Πρώτα απ' όλα, ε, ευχαριστώ όλους για τις ομιλίες που μας έδωσαν, τους οποίες έχετε στους φακέλους σας. Έχετε και τα βιογραφικά σημειώματα όλων των ομιλητών, λογικά. Δεν θα τους παρουσιάσω λοιπόν έναν έναν, αλλά διαβάστε τα γιατί είναι όλοι εξαιρετικοί επαγγελματίες. Απλώ να πω σε όλου ότι καλό θα ήταν να σεβαστούν το χρόνο ομιλία του. Ξέρω ότι είναι κάπω περιοριστικό αυτό, αλλιώ δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε του πάντε. Χωρί καθυστέρηση λοιπόν, θα καλέσω τη Λάρα να ανοίξει την ακρόαση. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Καλημέρα σε όλου. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση και εκ των προτέρων ευχαριστώ τον καθένα από εσά για την παρουσία του και για τη συνεισφορά, τη σημαντική συνεισφορά που ελπίζουμε ότι θα ακούσουμε από εσά κατά την ακρόαση αυτή. Όπως σωστά θύμισε ο Πρόεδρος, αυτή είναι μια δεύτερη ακρόαση σε σχέση με την ακρόαση που είχε οργανώσει ο συνάδελφος Κοζούσνικ. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την παρουσίαση κάποιων πτυχών που ξεκινούσαν από την Πήγαζε μάλλον από την έκθεση πρωτοβουλίας. Εδώ σε αυτήν την διακοινοβουλευτική συζήτηση θα οδηγηθούμε στην ε, υιοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί θα έχουμε έναν κανονισμό αρκετά ευαίσθητου χαρακτήρα και πολύ χρήσιμο. Διότι θα οδεύει, ελπίζουμε, στη σωστή κατεύθυνση και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή μέρα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και για τη δημοκρατία. Με τις πολιτικές εξελίξεις όπως τις βιώνουμε πρόσφατα και όπως τις βιώνουν πολλοί από αυτούς τους συναδέλφους αποδεικνύει ότι πρέπει να είμαστε στην υπηρεσία των πολιτών. Την, ε, τους πολίτες της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν όπως βλέπετε επιλέξαμε και αφήσει που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών, τις δραστηριότητες που ο καθένας από εμά διεξάγει καθημερινά. Θέλουμε λοιπόν διάλογος να υπάρξει μεταξύ μας και είμαι πεπισμένη ότι θα είναι χρήσιμος. Ελπίζω ότι με την διοργάνωση της ακρόασης που προτείναμε θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις σημαντικές πτυχές για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του πώς ε, εξελίσσεται η τυποποίηση, ποιες διαδικασίες εμπλέκονται εδώ και ποιες βελτιώσεις είναι απαραίτητες πώς θα γίνει το σύστημα πιο γερό. Ήδη έχουμε επιτελέσει σημαντικό έργο εδώ. Ω κοινοβούλιο έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα με μια έκθεση πρωτοβουλία η οποία εγκρίθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Γκοζούσνικ και όσους και όδους εισηγητές συμμετείχαν διότι βοήθησαν να είναι πολύ συγκεκριμένη έκθεση και σκόπιμη και εύστοχη. Βλέπουμε όμως ότι πολλά από τα ζητήματα τίθενται ξανά ε, και μάλιστα πολλοί από τους ε, νέους εισηγητές στη δεύτερη φάση εξέτασης της τυποποίησης συμμετέχουν εκ νέου. Πρόθεσή μου εδώ είναι να συνεργαστούμε στενά μεταξύ μας, όπως και στο παρελθόν, αυτό να συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον. Θα εκπροσωπηθούν προφανώς όλες οι πολιτικές ομάδες και όλες οι πολιτικές ε, δυναμικές. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό για να υπάρχει συνένεση και να υπάρξει ένα τέτοιο αποτέλεσμα στην Ολομέλεια που να ικανοποιήσει όλους μας. Επίση, σημειώνω με ικανοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επεξεργασία του πακέτου αναθεώρησης για την τυποποίηση έλαβε υπόψη τη πολλέ από τι προτάσει που προήλθαν από το Κοινοβούλιο. Αυτό προφανώς μας κάνει όλους υπερήφανους και σας ευχαριστούμε. Εδώ λοιπόν ε, δουλειά μας είναι να εντοπίσουμε ποια σημεία θα μπορούσαν να βελτιωθούν στην πρόταση της Επιτροπής. Βεβαίως το σημείο από το οποίο ξεκινάμε είναι εξαιρετικό, αλλά θα μπορούσαμε να δούμε πώς θα υλοποιηθεί ακόμη καλύτερα. Θα έλεγα λοιπόν να ακολουθήσουμε εδώ μια ρεαλιστική προσέγγιση κοντά στην πραγματικότητα που να μας επιτρέψει να δούμε ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα ώστε η όλη διαδικασία να γίνει πιο εύχρηστη και καλής ποιότητας. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής τυποποίησης είναι πολύ σημαντική. Το γνωρίζουμε όλοι. Η αναθεώρηση αυτή σήμερα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της ε, γενικότερης οικονομικής κρίσης. Πρέπει λοιπόν να είμαστε και ταχείς αλλά πρέπει να επιδιώξουμε να πετύχουμε και τον στόχο κλειδί για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η εσωτερική αγορά έχει ανάγκη να απελευθερωθεί από φραγμούς που την παρεμποδίζουν και πρέπει να τονωθεί επίσης. Για να απλουστευτεί χρειάζονται αρκετές προτάσεις και για την ανάπτυξη εδώ το είδαμε αυτό και με το Single Market Act και με άλλες προτάσεις και με αυτή την έκθεση έχουμε μια νέα ευκαιρία. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις της Ευρώπης. Θα πρέπει να λάβει υπόψη τις χρονικές, τους χρονικούς περιορισμούς, θα πρέπει να είναι ταχύ λοιπόν και να είναι και γραμμικό, να ανταποκρίνεται και στις τεχνολογικές αλλαγές που αντιμετωπίζουμε. Εδώ δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειες σε αυτή την παρουσίαση. Θα είμαι σύντομη, διότι δεν θέλω να αφαιρέσω και χρόνο από τους ομιλητές μας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα λάβω υπόψη αυτό που μου λέει και ο πρόεδρος εδώ δίπλα μου. Καλύτερα να έχετε εσείς περισσότερο χρόνο για να παρουσιάσετε τις δικές σας ομιλίες, τις δικές σας συνεισφορές και τις απόψεις σας. Ας αρχίσουμε λοιπόν επισήμως την ακρόαση. Σας εύχομαι σε όλους καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Δίνετε ένα καλό παράδειγμα και στους ομιλητές με τη συντομία σας. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Γκίρετ και από τον, Γκέρετ και από τον κύριο Πράουτ αν θέλουν να κάνουν κάποια σχόλια εξ ονόματος των επιτροπών τους για ένα-δύο λεπτά. Φυσικά θα έχετε τη δυνατότητα να παρέμβετε αργότερα. Ο κύριος Γκίρετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για αυτή την ακρόαση που εστιάζει σε θέματα τυποποίηση στη βιομηχανία. Χωρίς τυποποίηση η βιομηχανία δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν μας ενδιαφέρει η ποιότητα των προϊόντων, θα πρέπει να προωθηθεί η ποιότητα μέσω της τυποποίησης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την προστασία των καταναλωτών. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε μεταλαμπάδευση βελτίστων πρακτικών και να εξασφαλίσουμε και μία συνένεση για όλους αυτούς οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία αυτή. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ταχεία ανάπτυξη στις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις τεχνολογίες ε, στον πυρηνικό τομέα, στη βιοτεχνολογία. Όλοι αυτοί οι τομείς είναι σε ραγδαία ανάπτυξη. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επομένως αποδίδει μεγάλη σημασία στο να υπάρξει η συνεργασία των κρατών μελών για να μπορέσουν να υπερπηδηθούν τα εμπόδια σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα και να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν ε, συμβατές συμβατά πρότυπα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα προϊόντα σε κάθε κράτος μέλος να μπορούν να λειτουργήσουν και να γίνονται αποδεκτά και στις αγορές των άλλων κρατών των μελών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι διάφανη, δημοκρατική και θα χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα και αμεροληψία. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και σεβασμός όλων των προτύπων. <clears throat> Γιατί τα πρότυπα τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά από τη βιομηχανία απλώς δεν θα εφαρμοστούν στη συνέχεια. Αυτό απαιτεί λοιπόν την συμμετοχή όλων των φορέων και των κρατών μελών. Εξάλλου, η χρήση των προτύπων αυτών στην αγορά σημαίνει και μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές. Η Ευρώπη, λοιπόν, ε, είναι πρωτοπόρος σε διάφορα προϊόντα, όπως είναι φαρμακευτικά προϊόντα, χημικά προϊόντα, προϊόντα για την κατασκευαστική βιομηχανία κτλ. Αυτή η διαδικασία όμως είναι σε κίνδυνο γιατί υπάρχει και η μετακίνηση των επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θεμελιώδους σημασία τα πρότυπα για να εξασφαλιστεί ότι ακόμα και η μετακίνηση των επιχειρήσεων δεν θα θυγεί η διαδικασία της ε, βιομηχανίας στην ε, Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν να ιδιέπονται οι αγορές ανεξάρτητα από όπου γίνεται η παραγωγή, από τις ίδιες αρχές και τα ίδια πρότυπα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να προωθήσουμε τη διαδικασία εναρμόνισης στην Ευρώπη και έτσι να χρησιμοποιήσουμε όλο το δυναμικό το οποίο μπορεί να προκύψει μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Η τυποποίηση και η παροχή διπλωμάτων ευαισθητεχνίες είναι δύο θεμελιώδη εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και στις εργασίες της Κομισιόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσετε. Ελπίζω να μην μίλησα πολύ γρήγορα και να μην ε, δημιούργησα προβλήματα στους διερμηνείς. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ήσασταν πάρα πολύ σαφείς και είναι τσακάλια οι διερμηνείς μας. Ο κύριος Προύστ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την ε, Επιτροπή σας και ιδιαίτερα την εισηγήτρια που με προσκαλέσατε για να λάβω το λόγο, την ευκαιρία αυτού του διαλόγου σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έναν κανονισμό που αφορά την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Η τυποποίηση έχει άμεσο αντίκτυπο για την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, τι διεθνεί συναλλαγέ και ελπίζω η συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μα να είναι αποτελεσματική. Ελπίζω επίση ότι θα συναντήσω ξανά την εισηγήτρια ώστε να υπάρξει απόλυτο συντονισμό μεταξύ των εργασιών των δύο επιτροπών μα. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την πρόταση κανονισμού, που από όλε τι πτυχέ φαίνεται ικανοποιητική, όμω από την άποψη του διεθνού εμπορίου θα μπορούσε να επιδεχτεί και των βελτιώσεων. Θα Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η διεθνή ε, διάσταση λύπη, απουσιάζει σχεδόν απόλυτα από την πρόταση αυτή. Δύο λοιπόν ε, συλλογιστικέ θα πρέπει να μα απασχολήσουν. Πρώτα απ' όλα η θέση που δίνεται στα διάφορα φόρουμ και κονσόρσια στον ε, τομέα των ΤΕΙΣΕ κυρίω. Επίση, τι γίνεται με τι αρχέ του ΠΟΕ στην αναγνώριση των ειδικών διαπιστεύσεων και την χρήση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών στι διεθνεί αγορέ για να παραμείνουμε σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε σχέση με τα διάφορα φόρα και κονσόρσια, πρέπει να προσπαθήσουμε στο κείμενο αυτό να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που προτείνονται στο παράρτημα 2 από τα διάφορα διεθνή φόρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι το συγκεκριμένο άρθρο παροτρύνει τις μεγάλες επιχειρήσεις να συνεργάζονται μεταξύ τους για, τεχνικές, ε, για τεχνικά πρότυπα που θα πρέπει να περνούν από διεθνή φόρα και κονσόρσια και όχι από τι κλασικέ διαδικασίε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσει μεταξύ των κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων, των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οργανώσεων καταναλωτών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν τίθεται θέμα θέμα του ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων τυποποίηση και των υπόλοιπων διεθνών φορέων. Μπορεί οι προδιαγραφέ να γίνουν κάποια στιγμή δύσκολε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει μα. Έτσι δημιουργούνται δύο μεγάλε, μάλλον οι δύο μεγάλε πολιτικέ ε, ομάδε πολλέ φορέ ε, οργανώνονται σε ευρύτερα πλαίσια ώστε να επιβάλλουν τη δική τους άποψη και αυτό αποτελεί τροχοπέδι. Θα πρέπει λοιπόν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μην υποχρώνονται από κάποιον εκτός ένωσης γίγαντα στο να επιβάλλουν κανόνες που δεν μπορούν να τις ε, υλοποιήσουν. Επίσης, το παράρτημα 2 έχει να κάνει και με τους κανόνες του ΠΟΕ που ισχύουν για την αναγνώριση των τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των ΤΕΙΣΕ, δηλαδή πάλι σε σχέση με τα φόρα και τα κονσόρσια. Αυτό ε, γύρει πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί η Επιτροπή θεωρεί ότι ο τομέας των ε, ΤΙΚ θα πρέπει να είναι ένα τομέα εξαιρέσεων. Γιατί θεωρεί επίση η Επιτροπή ότι και οι τεχνικέ προδιαγραφέ έχουν να κάνουν με τον τομέα των TIC. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει δύο παράλληλα συστήματα και δύο ταχύτητε στο συστηματικοποίηση. Για τα κριτήρια του του 2 πρέπει να σκεφτούμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένα δεν τα λαμβάνει υπόψη ενώ άλλα τα προσθέτει. ποια είναι η αιτιολόγηση των επιλογών της αυτών. Επίσης για κάτι που θα πρέπει να είναι σαφές ε, γιατί δεν επιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση των ευρωπαϊκών βιντεογραφών στη διεθνή αγορά. Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον εκτό Ευρώπη θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο για τη χρήση και τη διάδοση των δικών μα προτύπων ε, στι διεθνεί αγορέ. Εξάλλου, η συνεργασία με τα τρίτα κράτη είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτόν τον λόγο οι διμερείς συζητήσεις που εξεγάγουμε με ξένα κράτη ελπίζουμε ότι θα αποφέρουν καρπούς, αλλά εδώ χρειάζεται εταιρική σχέση σαφώς με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε για διατλαντική συνεργασία και για την χρηματοδότηση των Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων που πηγαίνουν σε αναδυόμενες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες όπως έγινε πρόσφατα με την Κίνα. Επίσης ε, κάποια στιγμή ε, είχε ληφθεί απόφαση να, να αποσταλεί εμπειρογνώμονα στην Ινδία, αλλά κάποια στιγμή χάθηκε στο γραφειοκρατικό λαβύρινθο η ιδέα αυτή. Επίση και με τη Ρωσία θα έπρεπε να σκεφτούμε τι συνεργασία μπορεί να γίνει. Θα καλέσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θυμηθεί αυτό που προτείνει το 2010 κατά τι διαβουλεύσει μα. Δηλαδή την έναρξη ενό διαγωνισμού ε, που να συμπεριλαμβάνει συμμετέχοντα και εκτό Ευρώπη. Ε, με συμμετοχή Κίνα ή Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω χάρη. Και αυτό προκειμένου να ετοιμάσουμε πιο ολοκληρωμένα την ευρωπαϊκή διαδικασία. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Τροπή φαίνεται να εγκατέλειψε αυτή την ευρωπαικη διαδικασια βεβαια η ευρωπαικη επιτροπη φαινεται να εγκατελειψε αυτη την ιδεα και αυτό το αποδεικνύει η πρόταση κανονισμού. Μόνο οι ευρωπαϊκοί φορεί ε, τυποποίηση ε, θα πρέπει να έχουν ε, τη δυνατότητα να πιστοποιούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μόνο έτσι θα παραμένει συνεπέ το σύστημά μα και θα μπορούμε να σεβόμαστε πλήρω τι αρχέ του ΠΟΕ. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Uh, σα ευχαριστώ κύριε Προύστ για την ευρεία προοπτική που μας παρουσιάσατε με βάση τις ειδικές γνώσεις που έχετε και από την Επιτροπή σας και για κάποια ζητήματα που γίνατε επίσης σας ευχαριστώ ιδιαίτερα ιδίω το τι γίνεται με τις τεχνολογικές ε, προδιαγραφές και τους ειδικούς φορείς αυτά θα προκύψουν και στη συζήτηση αργότερα ελπίζω οπότε ίσως να λάβετε απαντήσεις στα ερωτήματά σας επειδή είμαστε στην αρχή της ακρόασης, ίσως να καλέσω τώρα την Επιτροπή να μας δώσει μια γενική εικόνα. Η κυρία Ρενάτα Βάισενχορν βρίσκεται επίσης εδώ που είναι υπεύθυνη για τις λεπτομέρειες της Επιτροπής μας με την κυρία Μπρίνκμαν. Αλλά κυρίω θα καλωσορίσω τον κύριο Καλέχα Κρέσπο, ο οποίο είναι αναπληρωτή διευθυντή τη ε, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανία. Θα έχετε και εσεί λοιπόν το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι. Είμαι ευγνώμων που το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ΙΝΚΟ διοργάνωσαν τη σημερινή συνεδρίαση, γιατί δίδεται ευκαιρία στους ενδιαφερομένους να έχουν λόγο σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Ο ρόλος της ε, ευρωπαϊκής ε, τυποποίησης ενισχύει την ανταγωνιστικότητα. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τον ε, εκ μέρους του Αντιπροέδρου Βαλιάνη γιατί ήθελε να είναι σήμερα εδώ. Δυστυχώς όμως τώρα λαμβάνει η χώρα η συνεδρία των Επιτρόπων της ε, Κομισιόν και έπρεπε να βρίσκεται εκεί γιατί και εκεί υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα τα οποία συζητώνται σήμερα. Θα ήθελα να αρχίσω ε, συμφωνώντας με τους προηγούμενους ομιλητές ότι η τυποποίηση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η συνεργασία ανάμεσα στη βιομηχανία, τους χρήστες, τις δημόσιες αρχές και τους οργανισμούς ευρωπαϊκής τυποποίησης έχει συνεισφέρει αποφασιστικά σε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρώπης, τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς 500 εκατομμυρίων ανθρώπων. Έχει παίξει ζωτικό ρόλο στην ε, τόνωση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη και έχει βοηθήσει τις ε, επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην ε, παγκόσμια αγορά και έχει διασφαλίσει την ε, διαλειτουργικότητα που προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Στην παρέμβασή μου θα αναφερθώ στον σημαντικό ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Όπως ξέρετε, μία από τις, είναι μία από τις αρμοδιότητές μου στην είναι λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις πολύ σημαντικέ διότι προσελκύουν καταναλωτές, μειώνουν κίνδυνο και αυξάνουν την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση που προκύπτει από την χρήση των ε, προτύπων στις αγορές. Και ακριβώς γι' αυτό είναι σημαντική η τυποποίηση. Και ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται να εξυγχρονίσουμε την τυποποίηση και να μπορούμε να εναρμονίσουμε το σύστημα με τις νέε προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και την σύγκληση των τεχνολογιών. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ε, εταίρων κλειδί και πρέπει να προσπαθούμε συχνά, ε, συνέχεια να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων. Στις αρχές Ιουνίου υιοθετήθηκε και από την Κομισιόν. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ορισμένα από τα στοιχεία κλειδιά. Καταρχάς την φιλοσοφία της τυποποίησης. Η φιλοσοφία λοιπόν πίσω από αυτό το πακέτο είναι ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία η ευρωπαϊκή τυποποίηση θα κληθεί να παίξει έναν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο διότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, στρατηγική Ευρώπη 2020 για προώθηση ολοκληρωμένης χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης. Στην βιομηχανική πολιτική, στην ε, ψηφιακή ατζέντα, στην, ε, στην καινοτομία, σε όλους αυτούς τους τομείς είναι, σημαντικό, ε, είναι ξεκάθαρο ότι η τυποποίηση θα παίξει σημαντικό ρόλο εάν θέλουμε να καταφέρουμε τους στόχους μας. Επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ενιαία αγορά. Γι' αυτό λοιπόν το πακέτο μας πρέπει να το βλέπουμε ως σύνολο. Έχουμε στρατηγική για την επικοινωνία και έχουμε μία πρόταση για ρύθμιση της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Έπειτα, το πακέτο θα αποτελεί μία εξέλιξη, όχι επανάσταση. Η τυποποίηση είναι ήδη επιτυχημένη, αλλά θέλουμε να, το, να την εξυγχρονίσουμε και να την βελτιώσουμε. Δεν θέλουμε όμως να αλλάξουμε αυτό που δουλεύει προς το παρόν. Δεν θέλουμε να το κάνουμε χειρότερο. Αν κάτι δεν είναι χαλασμένο, δεν χρειάζεται να το φτιάξουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να εξυγχρονίσουμε και να προσαρμόσουμε στα νέα στοιχεία την τυποποίηση. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης θα συνεχίσει να διαχειρίζεται από τρεις ε, ανεξάρτητους ε, ιδιωτικούς οργανισμούς και δεν θα αλλάξει τίποτα στην ε, εθνική στις εθνικές αντιπροσωπείες. Το υπάρχουν στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο ένας ε, κανονισμός θα συνδυάσει την απόφαση του 2006 για την χρηματοδότηση συν την οδηγία. Έτσι λοιπόν τρία διαφορετικά κείμενα θα ενωθούν σε έναν κανονισμό και θα απλοποιηθούν. Επίσης θα, θα αντιμετωπίσουμε ορισμένες ελλείψεις που έχει το παρόν σύστημα. Καταρχάς, η ταχύτητα. Και θα είμαι σύντομος γιατί ο πρόεδρος μου υποδεικνύει ότι πρέπει να κάνω πιο γρήγορα. Καταρχάς, πρέπει να μειώσουμε τον ε, μέσο όρο ανάπτυξης προτύπων. Μπορούμε να είμαστε καλύτεροι χωρίς να χάσουμε σε ποιότητα. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό για να είμαστε για να ακολουθούμε τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Οι οργανισμοί τυποποίηση θα ε, πρέπει να ε, αποδίδουν πιο γρήγορα, αλλά επίση χρειαζόμαστε και ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασία έτσι ώστε να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε τα κύρια σημεία με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Επίσης η χρηματοδότηση και η χρηματική υποστήριξη θα αποσκοπεί σε ε, τεχνολογική ανάπτυξη και βελτίωση των προτύπων χωρίς να, και το τονίζω αυτό, χωρίς να χαθεί η ποιότητα. Έπειτα, καινοτομία. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τη σχέση ανάμεσα στην τυποποίηση και την έρευνα και να δώσουμε επίσης και σημαντικό ρόλο στο, στην κοινή ομάδα έρευνας της Κομισιόν. Έπειτα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε, την προστασία του καταναλωτή, την ευελτίωση στην πρόσβαση, την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά τα ζητήματα απαιτούν αποδοτική και σωστή τυποποίηση και εδώ μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Επίσης, ολοκλήρωση, χωρίς αποκλεισμούς. Πρέπει να φροντίσουμε όλοι οι φορείς να, αντιπροσωπευ... Ε, να αντιπροσωπεύονται επαρκώς, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. ταυτόχρονα ε, θα ζητήσουμε από, τα, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ενδιαφερομένων και σε εθνικό επίπεδο. Έπειτα, ο τομέας των υπηρεσιών, η τυποποίηση και η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά των Υπηρεσιών. Η ευρωπαϊκή οικονομία ε, εξαρτάται όλο ένα και περισσότερο από τις υπηρεσίες και αυτό δεν ε, φαίνεται στην τυποποίηση. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τυποποίηση για να υποστηρίξουμε την ε, ενιαία αγορά των υπηρεσιών, όπως ακριβώς υποστηρίζουμε και την ενιαία αγορά στον τομέα των αγαθών. Έπειτα, η τυποποίηση των προτύπων ICT. Κάποιοι ομιλητές το ανέφεραν. Το ICT αφορά όλους μας, όμως πολλά από τα σημαντικά πρότυπα δεν, είναι, δεν ε, καταρτίζονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τυποποίησης. Οι προδιαγραφές πρέπει να εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές του ΠΟΕ και η Κομισιόν πρέπει να το φροντίσει αυτό. Είναι, είναι αυτό πολύ σημαντικό για, την ηλεκτρονική, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, μεταφορών και επίσης πρέπει να δημιουργηθούν πρότυπα και για τις δημόσιες προμήθειες. Επίσης, η Κομισιόν θα ζητήσει από τους CSO να ενισχύσουν τις, ε, τους δεσμούς τους με τα κονσόρτια. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άδεια που μου δώσετε να μιλήσω περισσότερο. Στην παγκόσμια αγορά. Η παγκόσμια αγορά είναι κάτι που δεν το έχουμε παραμελήσει και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Τα πρότυπα είναι κρίσιμη σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία επεκτείνουν το εμπόριο. Η Ευρώπη τα υποστηρίζει και πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τον ρόλο μας. Ωστόσο, το σύστημα ευρωπαϊκής τυποποίησης πρέπει να προωθηθεί και στον κόσμο. Και αυτό θα γίνει με περισσότερη και καλύτερη, καλύτερα συντονισμένη συνεργασία. Η Κομισιόν, και σας διαβεβαιώ γι' αυτό, υποστηρίζει τους ε, εμπειρογνώμονες τυποποίησης ε, στις διαφορές χώρες και επίσης θα διεξάγει στρατηγική σημασία συνομιλίες με τους, ε, με τους εταίρους μας. Την επόμενο μήνα θα έχουμε συζήτηση με τις Ηνωμένε Πολιτείε και, και συζήτηση με το ρυθμιστικό σώμα των τυποποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμω πρέπει να συνεχίσουμε και να επεκταθούμε και στην Ιαπωνία, στην Ινδία, την Κίνα και την Βραζιλία. Κλείνοντα λοιπόν, προσπάθησα σύντομα να υπογραμμίσω τα σημαντικά στοιχεία. Είναι φιλόδοξο το έργο που θέλουμε να κάνουμε, όμως δεν είναι μόνο η Κομισιόν που προτείνει κάτι. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στην διαδικασία τυποποίησης και αυτό που ζητούμε από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο των Υπουργών είναι να διεξάγουν εις βάθος συζητήσεις για το πακέτο αυτό και θα θέλαμε, εάν η διαδικασία συναπόφασης πάει προς την σωστή κατεύθυνση, να κάνουμε μεγάλη πρόοδο στην ε, επερχόμενη Δανική Προεδρία. Ευχαριστούμε την Πολωνική Προεδρία για την εξαιρετική δουλειά της και εάν είναι δυνατόν στις αρχές του 2013 θα θέλαμε να έχουμε μία επικαιροποιημένη διαδικασία τυποποίησης. Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για το έργο που έχουμε να κάνουμε. Θα, ακούσουμε, θα σας ακούσουμε με μεγάλη προσοχή και σας ευχαριστούμε τέλος για την, ε, για την υπομονή σας και σας ευχόμαστε μια παραγωγική ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ντάνιελ. Επειδή είπες ότι μόνο πέντε σημεία θα αναφέρεις, Ντάνιελ, πριν από στην αρχή της ομιλίας σου, είπα να σε ακούσουμε στο τέλος. Πάρα, πολύ καλό πλαίσιο είναι αυτό πάντως που δημιουργείται για το έργο μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάντως για την προσωπική σας προσήλωση και αυτή του Επιτρόπου Ταγιάννη επίσης. Όπως είπε ο Ντάνιελ λοιπόν, ο πρώτος στόχος του πακέτου είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας και χωρίς να θίξουμε την ποιότητα. Ερχόμαστε λοιπόν στην πρώτη παρέμβαση και χαίρομαι πολύ που μπορώ να δώσω το λόγο σε ένα άτομο που έχει παίξει ένα κομβικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και είναι τακτική επισκέπτη στην ε, Επιτροπή μας η Έλενα Σαντιάγο, η οποία είναι Γενική Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Τυποποίηση ΣΕΝ και της ε, Επιτροπής για Ηλεκτρομηχανική Τυποποίηση ΣΕΝΕΛΕΚ. Έξι λεπτά όπως όλοι οι άλλοι βέβαια. Έλενα και σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΙΜΚΟ για το γεγονό ότι δίνει στην, ε, στο σύστημα τυποποίηση τη Ευρώπη, την δυνατότητα να εξηγήσει το έργο μα, τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε και το ευχαριστώ που θέτεται σε υψηλό επίπεδο στην πολιτική ατζέντα το θέμα τη τυποποίηση. Τα πρότυπα βρίσκονται παντού, είτε τα βλέπουμε είτε όχι. Χωρί τα πρότυπα όμω, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τόσο ασφαλείς και τόσο αποτελεσματικοί όπως είμαστε σήμερα. Είναι σημαντικό λοιπόν να κρατήσω ένα σωστό ρυθμό αλλά να μην θίξω την ποιότητα της παρουσίασής μου. Το ίδιο πράγμα κάνουμε με τα προϊόντα και τα αγαθά και τα πρότυπα που τα διέπουν. Τα βασικά στοιχεία της παρουσίασής μου μπορούν να συνοψιστούν σε τέσσερα σημεία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι σημαντική η ταχύτητα στη διαδικασία τυποποίηση, πρέπει να ανταποκριθεί στι ανάγκε των τομέων, Κάθε τομέα έχει ειδικέ ανάγκες και πρέπει να είμαστε έτοιμοι επίσης να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία συνένεση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Η ταχύτητα από μόνη δεν μπορεί να είναι ο μόνος στόχος. Πρέπει να είμαστε έγκαιροι στην προσέγγισή μας και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκε τη αγορά. Και θέλω εδώ να τονίσω το δεύτερο σημείο. Δεν πρέπει να θυσιάσουμε την ποιότητα και τον διεθνή χαρακτήρα για να επιτύχουμε μονάχα την ταχύτητα. Χρειάζεται να είμαστε κοντά στην αγορά, να είμαστε σχετικοί με τις ανάγκες της αγοράς και θα πρέπει να υπάρξει ελκυστικότητα του τομέα τυποποίησης για την αγορά, γιατί πρέπει και αυτή να συμβάλλουν στο έργο μας. Πρέπει να κάνουμε και κάποιες προτάσεις για να εξασφαλίσουμε και την απλοποίηση και να μπορέσουμε να εμπλέξουμε όλους αυτούς που θέλουν στο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης, γιατί ξέρουμε ότι ορισμένε φορές μπορεί να είναι επαχθείς και πολύπλοκες οι διαδικασίες. Έχω δύο παραδείγματα για το, για το μέσο χρόνο που χρειάζεται για να επιτευχθούν τα πρότυπα σε διάφορους τομείς. Βλέπετε, ίσως δεν βλέπετε, ότι ορισμένοι τομείς πάνε γρήγορα γιατί χρειάζεται να περάσουν γρήγορα τα πρότυπα στην αγορά, άλλοι τομείς προτιμούν μεγαλύτερη σταθερότητα και μεγαλύτερη βεβαιότητα σε ό,τι αφορά την παραγωγή προτύπων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το χρόνο δημοσίευσης των προτύπων μέσα στην ευρωπαϊκή διαδικασία τυποποίηση τα τελευταία 5-6 χρόνια και αν λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες τυποποίηση μπορούμε να έχουμε κάποια πρότυπα τα οποία δεν θα φτάσουν ποτέ στο διεθνές επίπεδο γιατί δεν υπάρχει ανάγκη, αλλά έχουμε παράλληλα και διεθνή ευρωπαϊκά συγγνώμη, πρότυπα τα οποία προετοιμάζονται παράλληλα και μαζί με διεθνή πρότυπα. Αυτά απαιτούν λίγο περισσότερο χρόνο. Ο χρόνος λοιπόν προετοιμασίας για αυτά τα πρότυπα είναι κάπως πιο υψηλός. Αυτό εξαρτάται βέβαια από τον επιδιωκόμενο στόχο. Η σχέση ταχύτητος και ποιότητας. Και πάλι πρέπει να επανέλθω στην ε, αίτηση που διατύπωσε η Κομισιόν. Στι αιτήσει τη Κομισιόν, καλύτερα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι υποστηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή βιομηχανία σε διεθνέ επίπεδο. Ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στι παγκόσμιε αγορέ. Έχουμε μια άλλη αίτηση ότι τα ευρωπαϊκά στάνταρ θα πρέπει να εκπροσωπούν τα συμφέροντα όλων των κατηγοριών εμπλεκομένων. Και επίση, μέσα στη διαδικασία αυτή εξυγχρονισμού, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης των προτύπων. Πρέπει επίσης να το συνδυάσουμε αυτό με την ταχύτητα αλλά και την ποιότητα. Οι ΣΕΝ και οι ΣΕΝΕΛΕΚ λοιπόν έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στους παγκόσμιους φορείς τυποποίησης. Έχουμε εθνικές διαδικασίες διαβούλευσης Έχουμε την αρχή ότι πρέπει να συμμετέχουν εθνικές αντιπροσωπείες στη διαργασία μας. Γενικά λοιπόν προσπαθούμε να εμπλέξουμε όλους τους απαραίτητους εμπλεκομένους στη διαδικασία αυτή, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη δική τους θέληση και διαθεσιμότητα να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία για να επιτύχουν μια συνένεση. Φυσικά υποθενοείται ότι πρέπει να έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη και η διαδικασία έγκρισης των προτύπων γίνεται με γενική συμφωνία και συνένεση. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία να δούμε μέτρα εκπαίδευση για την υποποίηση. Ένα άλλο στοιχείο που μα απασχολεί είναι το να είμαστε εγγύ στην αγορά. Μα ενδιαφέρει πάρα πολύ τα πρότυπά μα να εκπροσωπούν το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογία το οποίο έχει επιτευχθεί. Πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή λοιπόν στι ανάγκε αυτών οι οποίοι βρίσκονται στο επίπεδο τη αγορά. Αν δεν το πράξουμε αυτό, αντί να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίηση, θα το αποδυναμώσουμε. Μας ενδιαφέρει τα πρότυπά μας να χρησιμοποιούνται από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί αυτοί θα είναι, ο ιδιωτικό τομέα είναι αυτοί οι οποίοι θα εφαρμόσουν αυτά τα πρότυπα. Ξέρουμε ότι 95% του κόστου του συστήματο το επομίζει το ιδιωτικό τομέα, αλλά συμβάλλει και κατά 99% <clears throat> σε σχέση με την εμπειρογνωμοσύνη για τι τεχνικέ και τεχνολογίε εχμής. Η ταχύτητα λοιπόν εξαρτάται από τη γνώση που έχουμε, από εμπορικά θέματα και από τι ανάγκε τη βιομηχανία. Η πρότασή μα είναι η εξή, να υπάρξει μια απλοποίηση των διαδικασιών και τη εκπαίδευση καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών και των διεθνών φορέων που συμμετέχουν στα θέματα αυτά, να αναπτύξουμε περισσότερο την ανάπτυξη και τι ηλεκτρονικέ πλατφόρμες για ταχύτερη ανάπτυξη εργαλείων πληροφορίας και επικοινωνίας, η Κομισιόν θα πρέπει να απλοποιήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο σύστημα τυποποίησης και επίσης πρέπει να εργαστούμε περισσότερο για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε την έρευνα στην ε, τυποποίηση και την καινοτομία, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν να προχωρήσουμε ταχύτερα τα συστήματά μας και πρέπει να έχουμε και μεγαλύτερη ορατότητα στα εθνικά προγράμματα Εκπαίδευση για να εκπαιδεύονται καλύτερα όλοι αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν στην υποποίηση. Μια κοινή προσπάθεια απλοποίηση θα βοηθήσει λοιπόν και την ταχύτητα ε, υιοθέτηση των προτύπων. Μου είπε ένα φίλο μου, πρέπει να δώσετε καλά παραδείγματα για αυτά που κάνετε. Να μερικά παραδείγματα λοιπόν καλών προτύπων. Έχουμε 20.000 τέτοια, αλλά σας δείχνω μόνο αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και για τις διαφάνειες. Πάντως ήταν πολύ καλή για μια από τις πρώτες παρουσιάσεις. Μας δώσατε νομίζω του σωστού προσανατολισμούς και ελπίζω ότι θα τους ακολουθήσουμε πιστά. Τώρα θα καλέσω τον κύριο Φάντερ Μπρακ, ο οποίος είναι μέλος της, της Philips και πρόεδρος του ομάδας εργασίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών. Έχετε 6 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις απόψεις της Business Europe σε αυτή την ακρόαση. Κάποια σημαντικέ Κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα. Η ευρωπαϊκή τυποποίηση πηγαίνει πολύ καλά. Καλωσορίζουμε λοιπόν τις βελτιώσεις χωρίς δραματικές ε, αλλαγές. Δεν το επιθυμούμε. Θα πρέπει να είναι εύστοχα και ποιοτικά τα πρότυπα που θα εγκριθούν. Έπειτα πρέπει να θέσουμε πρότυπα σε και ωφελεί βάση. Αυτό έχει εφαρμοστεί σήμερα και θέλουμε να συνεχιστεί και στο μέλλον. Έπειτα η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σε ισότιμη βάση είναι σημαντικό. Και αυτό ενδιαφέρει όλους τους ε, μετέχοντες στη διαδικασία. Έπειτα θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επαρκή ενημέρωση και οι ενώσεις ε, εκπαίδευση ή κατάρτισης έχουν, ε, μάλλον οι εμπορικέ οργανώσει έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτούνται αναλόγω. Επίση, θα πρέπει και για, τους δημόσιους, ε, για τις δημόσιες προμήθειες να υπάρχουν ε, σαφείς προδιαγραφές ICT. Αλλά για, τα πρότυπα εκτός των ICT δεν θα πρέπει να υπάρχει η ίδια διαδικασία. Ως τώρα η προσέγγιση μας είναι αρκετά ισορροπή, ιδίω με τι ε, αρχές που χρησιμοποιούνται για την πνευματική ιδιοκτησία. Έτσι τονώνεται η καινοτομία και οι προμηθευτέ, αλλά και οι χρήστε λοιπόν των προτύπων ωφελούνται από αυτή τη διαδικασία. Έπειτα θα πρέπει η νομοθεσία να στηρίζει την όλη διαδικασία και να μην αποτελέσει τροχοπέδι. Τα πρότυπα έχουν επιτρέψει την ε, καλή εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς. Πρώτον, επειδή δίνουν μεγάλες οικονομικές, καλά οικονομικά αποτελέσματα. Έπειτα, γιατί επιτρέπουν την καλή υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πολλές προτάσεις συνδέοντας με πολιτικούς στόχους την τυποποίηση. Όμως, το 70% των ευρωπαϊκών προτύπων έχουν ε, πολύ λίγο να κάνουν με τα δημόσια ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν τα πρότυπα να παραμένουν αυτό που είναι. Ιδιωτική σημαντικό και οικειοθελέ εργαλείο τη αγορά που να χρησιμοποιείται από τι επιχειρήσει σε βάση. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίζουν τι επιχειρήσει, αλλά να μην γίνουν πολιτικό εργαλείο τα πρότυπα. Διότι καθήκον των πολιτικών ε, είναι να ορίζουν τι πρέπει να γίνει και πώ να γίνει, όμω οι εμπειρογνώμονε θα πρέπει να δουν πώ ακριβώ θα πρέπει να εξελίσσονται τα πρότυπα. Νομίζουμε λοιπόν ότι οι πολιτικέ επιλογέ και στο μέλλον θα πρέπει να παραμείνουν στην πολιτική αρένα, ενώ οι επιλογέ για τα πρότυπα στου εμπειρογνώμονε των προδιαγραφών. Ας δούμε τώρα τα 12 αυτά κουτάκια, τα οποία όλα μαζί δημιουργούν αυτό το ενιαίο πακέτο. Σκεφτείτε πόση οικονομική αξία παρήγαγαν τα ε, πρότυπα μέσα στο πακέτο αυτό. Εδώ η λεγόμενη αποτελεσματική λογιστική οργάνωση ήταν μια ανάγκη της αγοράς που αφορούσε τους προμηθευτές, τους μεταφορείς, όλου του εμπλεκόμενου στη σχετική αγορά. Γιατί λοιπόν οι δημόσιε αρχέ να θέλουν να παρέμβουν σε μια τέτοια διαδικασία και να δημιουργήσουν σχετικά πρότυπα το 70% του συνόλου, όπω έλεγα. Τώρα, για να έχουμε καλά ε, πρότυπα που είναι αποτελεσματικά και δεν τα αγοράζουμε, ένα εύστοχο παράδειγμα. Όταν τα πρότυπα ε, δεν είναι αποτελεσματικά για τους χρήστες, μπορεί να γίνουν και επιζήμια. Πρώτα απ' όλα γιατί οι επενδύσει πάνε χαμένε για την αναπτύξη αυτών των προτύπων. Έπειτα γιατί τα πρότυπα αυτά μπορεί να γίνουν αναπόφευκτα για του οικονομικού φορεί και να αποστραγγίξουν την παραγωγικότητα ε, για τι ε, μεσαίου μεγέθου και μικρέ επιχειρήσει. Και εάν ε, ο σχεδιασμό του γίνει άνωθεν χωρί διαβουλεύσει με του ενδιαφερομένου, μπορεί να καταλήξουν να μην είναι έχρηστα. Έτσι λοιπόν και για την τεχνολογία και για τον τομέα εφαρμογής χρειάζεται ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Μια σημαντική επίσης διάσταση που να λάβουμε υπόψη είναι η διεθνή συνιστόσα. Πρέπει να έχουν χαμηλό κόστος τα πρότυπα και να υπάρχουν ισότιμοι όροι στην χρήση του ΣΕΝ και η ΣΕΝΕΛΕ και έχουν μια συμφωνία με την ΆΙΖΟ και την ΆΙΣΙ και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για την εξέλιξη τη ευρωπαϊκή τυποποίηση να συνεχίσει να, συνεχίσει να πηγαίνει στην διεθνή αυτή κατεύθυνση. Διότι για τους ενδιαφερομένους πρέπει να υπάρχουν διαβουλεύσεις προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι εξασφαλισμένο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει απαραίτητη πλατφόρμα για να γίνει αυτό. Συγκεκριμένα για την τυποποίηση των υπηρεσιών. Εδώ θα πρέπει να τεθούν στόχοι βάσει των αναγκών που υπάρχουν στην αγορά και όχι των πολιτικών φιλοδοξιών μας. Και ε, εξίσου σημαντικό, η συμμετοχή θα πρέπει να είναι από πραγματικού εμπειρογνώμονε που πραγματικά είναι αναφοσιωμένοι σε αυτό το θέμα. Ε, για την ε, συμμετοχή στον χώρο αυτό, λοιπόν, οι εμπειρογνώμονε θα πρέπει να ενημερώνονται και να λαμβάνουν μέρος στις αρμόδιους φορείς σε ισότιμους όρους όπως και τώρα. Θα πρέπει επίσης οι ενδιαφερόμενοι να οργανώνονται μεταξύ τους ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ακούγεται τη φωνή τους. Το γερμανικό μοντέλο μας δείχνει ότι αυτό μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καθοριστικό μήνυμα και για τις, αρχές των, τις εθνικές αρχές των κρατών μελών. Διότι αυτή τη στιγμή από την τυποποίηση έχουν άμεσα ε, ωφέλη. Όμως ε, είναι σημαντικό να υπάρξει συνεργασία για την εξέλιξη των προτύπων με ανάλογους κανόνες που να εκπροσωπούν τα δημόσια συμφέροντα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά σε αυτό τον τομέα. Πάντως υπάρχουν οργανώσεις επιχειρήσεων οι οποίες και πολύ καλά λειτουργούν και θα πρέπει να ακούγεται τη φωνή τους γενικότερα, όχι μόνο στο παράρτημα, στα θέματα του παράρτηματος 3. Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ γιατί ξεπέρασα ήδη το χρόνο μου. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την σαφέστατη παρουσίασή σας. Τα... Για όσους δεν τα παρακολούθησαν όλα οι διαφάνειες υπάρχουν στο φάκελο. Τώρα να καλωσορίσω και τον ε, γείτονά σα ε, που είναι ε, αναπληρωτή διευθυντή και θα τον ακούσουμε αργότερα. Και για μια συγκεκριμένη πτυχή των προτύπων που ήδη αναφέρθηκε για τον τομέα της, των τεχνολογιών επικοινωνίας. Εδώ θα ακούσουμε τον κύριο, τον πρόεδρο της ψηφιακής Ευρώπης. Έχετε το λόγο για έξι λεπτά. Mm. Τον κύριο Ζαν Λόρενς. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Εγώ εκπροσωπώ την Digital Europe, την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων ICT. Το νομοθετικό πακέτο που έχουμε μπροστά μας είναι αποτε... καρπός εξαιρετικού έργου που επιτέλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανιών τους ευχαριστούμε. Η Digital Europe ήταν μέρος της ε, διεθνή Επιτροπής που είχε αναλάβει το θέμα αυτό και έχει συμβάλει στο, στην όλη εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρώτο σημαντικό σχόλιο που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι ο προτινόμενος κανονισμός δεν έχει κανέναν αντίκτυπο για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Δηλαδή, η προσέγγιση θα συνεχιστεί στην ίδια κατεύθυνση και αυτό είναι σημαντικό για την ε, ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα κατάματα. Ο τομέας ICT, όπως τα ξέρετε, είναι ένας γοργά εξελισσόμενος τομέας. Με πολύ μεγάλη δόση καινοτομία και σημαντικό για τι διεθνεί ε, αγορέ. Χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή πλέον τα iPad, τα υφή ε, τηλέφωνα, τα smartphones παντού στην Ευρώπη και στον κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ειδικέ λεπτομέρειε για τα πρότυπα ICT και συγκεκριμένοι κανόνε. Ο νέο κανονισμό επιτρέπει την χρήση των υπερχόντων προτύπων και τη συμπλήρωσή του, προκειμένου να αναπτυχθούν νέα εφόσον χρειάζονται. Τα εργαλεία ICT και τα σχετικά προϊόντα είναι καθοριστική σημασία για όλου του τομεί. Παντού χρησιμοποιούνται συσκευέ ή έτσι είναι ένας καθοριστικός ε, συμμετέχων στον, στην όλη δικασία, υπάρχουν και άλλα φορά και κονσόρσια τα οποία παρέχουν πρότυπα για τον τομέα του διαδικτύου, τις εφαρμογές στο διαδίκτυο και αυτό που να το θυμόμαστε διαρκώς. Δεδομένης της σημασίας των προτύπων για τους δημόσιους διαγωνισμούς είναι Υπάρχουν και κυβερνήσει που έχουν αναπτύξει ειδικού κανόνε για την συμπερίληψη των προτύπων στου ε, διαγωνισμού. Θα πρέπει αυτό λοιπόν να το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να υπάρχει συνέπεια και συνοχή. Όχι μόνο για του δημόσιου διαγωνισμού αλλά και για την ευρωπαϊκή πολιτική και του σκοπού τη. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για την καινοτομία και προκειμένου να πετύχει αυτή στην Ευρώπη. Ένας πρωταρχικός στόχος μας για τον τομέα ICT είναι αυτό που ονομάζουμε διαλογικότητα. Τα προϊόντα βασίζονται στο hardware, αλλά υπάρχουν και πολλά διαφορετικά software λογισμικά, τα οποία θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο και από απόσταση, με τρόπο αποτελεσματικό. Ο κατάλληλος τρόπος είναι να χρησιμοποιούνται τέτοια πρότυπα κοινά που, για παράδειγμα, να λειτουργούν με όλα τα υπάρχοντα προϊόντα Δύο καθοριστικά άρθρα στο νέο κανονισμό είναι τα άρθρα 9 και 10 που αφορούν τον τομέα ICT. Όπως είπα είναι μεγάλη σημασία, ακριβώς γιατί το πρώτο άρθρο αφορά την συμπερίληψη των προτύπων στους δημόσιους διαγωνισμούς, αλλά πραγματικά θα το εκτιμούσαμε αν το Ευρωκοινοβούλιο βοηθούσε να γίνει ακόμη πιο ρητή η μνήμα των ευρωπαϊκών πολιτικών στα άρθρα αυτά. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για την κοινοτομία. Τα δύο αυτά άρθρα λοιπόν να παραμείνουν μεν στον κανονισμό, αλλά να ενισχυθούν. Να ενισχυθούν για την ε, κάλυψη και των ευρωπαϊκών πολιτικών. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια του παρατήματο 2, ευθυγραμμίζονται με τι αρχέ του ΠΟΕ, είναι ουσιαστικά και αυτά και στόχο εδώ ε, είναι να έχουμε απαριθμίσει τα πρότυπα που έχουν διαμορφωθεί με μια ανοιχτή διαδικασία, με διαφάνεια και με συνένεση. Μια σημαντική σύσταση εδώ είναι να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει ένας και μόνος τρόπος για να είμαστε διαφανείς, να οργανώνουμε τη συνένεση, να προκύπτει συμφωνία δηλαδή. Υπάρχουν διαφορετικά δημοκρατικά συστήματα με διαφορετικούς κανόνες, ποικίλουν, διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά είναι όλα δημοκρατικά. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη πλατφόρμα των ενδιαφερομένων ώστε να συζητούν μεταξύ τους και να βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει συμβατότητα με τα κριτήρια και ότι εντοπίζονται οι κατάλληλες ε, κινήσεις για τα πρότυπα. Οι ερευνητικές πλατφόρμες θα μπορούσαν να υποφελούνται και από την πείρα που έχει μέχρι τώρα αποκομίσει η Διεθνή επιτροπή, η Steering Committee. Η Digital Europe λοιπόν καλωσορίζει τον κανονισμό. Θεωρεί ότι είναι εξαιρετικό, άριστο το έργο που έχει επιτελεστεί και σε αυτή την αγορά με τόσο μεγάλη ανταγωνιστικότητα με ταχαίως αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα με τόσες ραγδαίες εξελίξεις θα πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση μας, να επικεντρωθούμε στη δημιουργία νέων προτύπων για νέες υπηρεσίες για καινοτόμους χώρους και όχι να κοιτάζουμε προς το παρελθόν. Το μέλλον θα πρέπει να αντικρίσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που στηρίζετε αυτή την πρωτοβουλία προς όφελος της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης και θα έλεγα και για την νεολαία στην Ευρώπη και για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λόρεντς. Δεν κρατήσατε τα τέσσερα λεπτά, νομίζω έξι μιλήσατε. Πάντως συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Νωρίτερα ακούσαμε για από την Business Europe για την σημασία της ευρωπαϊκής τυποποίηση. και γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πολύ να που καλωσορίζω έναν ε, από τους ηγητές του Ισπανικού Σύνδεσμου Τυποποίησης και Επιστοποίησης, τον κύριο τον συνάδελφο ο οποίος θα μας μιλήσει για το τι γίνεται στην Ισπανία κύριος Χαβιέ Γκαρσία Ντίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να κρατήσω το όριο των έξι λεπτών, όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοί μου. Καταρχάς, όμως, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Βερδέρα, που κανονικά θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ε, είναι άρρωστος και του εύχομαι καλή ανάρρωση. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας ενημερώσω στη θέση του και θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Σκεφτήκαμε μέσα στα έξι λεπτά να αναφέρουμε έξι σημαντικά μηνύματα για το γιατί η τυποποίηση των υπηρεσιών πρέπει να προωθείται έτσι όπως θέλουμε στον ε, παρόντα κανονισμό. Θα σα δώσουμε κάποιες ιδέες για τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα που η βιομηχανία των ε, υπηρεσιών βλέπει με την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Έπειτα, θα σας προσπαθήσουμε να σας πούμε πώς θα, η τυποποίηση θα προσπαθήσει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Έπειτα, πώς τα πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών συνεισφέρουν στην ποιότητα της ε, υπηρεσίας και την διαφάνεια ε, για τους χρήστες. Θα αναφερθούμε επίσης στο σύστημα SEN, που είναι κατά τη γνώμη μας η καλύτερη πλατφόρμα για τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις υπηρεσίες στην, ε, στον τομέα της εσωτερικής αγοράς. Έπειτα θα δούμε το πώς η ISO συμπληρώνει το σύστημα SEN στην βιομηχανία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και τέλος θα δούμε πώς τα ευρωπαϊκά πρότυπα μπορούν να συμπληρώσουν, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, το νομικό πλαίσιο με την εθελοντική επιχειρηματική δραστηριότητα. Όσον αφορά το πρώτο θέμα είναι η ανάγκη για ευρωπαϊκά πρότυπα στις υπηρεσίες. Τα κίνητρα για την ε, ανάπτυξη πρότυπων πρέπει να είναι θελοντικά και πρέπει να προέρχονται από τον τομέα της αγοράς και σε αυτό ε, είμαστε ε, δεσμευμένοι. Θέλουμε την συμμετοχή των πελατών στην αλυσίδα της επαροχής υπηρεσιών. Ε, ορισμένα από τα πλεονεκτήματα τα βλέπετε στην οθόνη. Θα σας αναφέρω αυτά που θεωρώ πιο σημαντικά φυσικά και το, το πρώτο. Οι απαιτήσει των ε, πελατών. Η καταπολέμηση του αθέμητου ανταγωνισμού και της ε, παροχής μη επαρκούς ποιότητας υπηρεσιών κτλ. Τώρα, δεύτερο σημείο, αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Εδώ αναφερόμαστε κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως ένα σημαντικό μέρος της ε, βιομηχανής παροχής υπηρεσιών στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις μικρές μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν και να διευκολύνουν την ε, αγορά. Η ανάπτυξη προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών συνεισφέρει στην δημιουργία και την διάχυση ε, προδιαγραφών στον τομέα των υπηρεσιών και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εμφάνισης ιδιωτικών προδιαγραφών από μεγάλους παίκτες, από μεγάλους φορείς οι οποίοι μπορούν να θέσουν περιορισμούς στην παροχή των υπηρεσιών. Όσον αφορά στους καταναλωτές, τους χρήστες, τους πελάτες, για αυτούς ποια είναι τα ωφέλη των ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών. Καταρχάς, τα πρότυπα διευκολύνουν τις υπεργολαβίες και διασφαλίζουν την ποιότητα όταν αναπτύσσονται στα πλαίσια των προδιαγραφών των ευρωπαϊκών αυτών προτύπων. Επίσης, τα πρότυπα είναι ανοιχτά σε οποιαδήποτε αξιολόγηση συμ... συμμόρφωσης από, το από, τους... από τους ε, πελάτες, τους τελικούς χρήστες, τους παραγωγούς έτσι όπως ε, άλλωστε αναφέρεται και στην ε, αντίστοιχη οδηγία στο άρθρο 26. Τέλος, τα πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών ενισχύουν την διασφάνεια και δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να συγκρίνουν διάφορες προσφορές από διάφορους παρόχους υπηρεσιών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του τομέα. Τέταρτο μήνυμα, γιατί το ΣΕΝ διότι το ΣΕΝ είναι ο πιο αξιόπιστος εταίρος στην ανάπτυξη προτύπων, πρώτον ε, επειδή έχει τεράστια εμπειρία. Η ανάπτυξη προτύπων δεν είναι αντίστοιχη του ειδικού βάρου στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά καλά παραδείγματα. Ε, η διαχείριση κτηρίων, για παράδειγμα, Και πρόσφατα, ε, όπως είδαμε, στον τομέα της αισθητικής, η τυποποίηση μας έχει δώσει θετικές εμπειρίες. Και έχει δημιουργηθεί ένα ε, έγγραφο το οποίο θέτει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα λειτουργούν τα πρότυπα στον τομέα των αυτών, στον τομέα αυτών έπειτα και τελειώνω παγκόσμια προοπτική πολλοί, πολλές ευρωπαϊκές SNB έχουν ηγετικό ρόλο στην ε, τυποποίηση, στο ίζο, στον τομέα του τουρισμού, στην ε, βιώσιμη διαχείριση Και βλέπουμε ότι ε, πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες και εταιρείε χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή πιστοποίηση για να εδραιωθούν στην παγκόσμια αγορά. Τελειώνω τώρα με την παρουσίασή μου. Πριν έκανα αναφορά στην εσωτερική αγορά και αυτό που θέλω να πω πάνω σε αυτό είναι ότι εμείς θέλουμε να πάρουμε αυτή την ευκαιρία και να ζητήσουμε από τους βουλευτές και από όλους τους ενδιαφερομένους να, ε, να δουν το προσχέδιο αυτό για την ευρωπαϊκή τυποποίηση και να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία αυτή για να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα ε, των παρόχων υπηρεσιών και να προστατεύσουν τους ε, καταναλωτές ε, έτσι της ευρωπαϊκής αγοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για τα έξι μηνύματά σας, παρότι δεν κρατήσατε το όριο του χρόνου. Τώρα προχωράμε και θα ακούσουμε τον κύριο Adrian Harris, είναι Γενικός Διευθυντής της Orgalim, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακών Βιομηχανιών. Και φυσικά αυτές οι βιομηχανίε είναι ένας ε, μεγάλος, ε, είναι χρήστη των προτύπων αυτών και οι βιομηχανίε αυτές είναι η πύλη προς την ε, ενιαία χώρα. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ Μάλκομ, ευχαριστώ και την Επιτροπή που μας καλέσατε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ, διότι για μα η τυποποίηση είναι, παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μα. Καταρχάς να σα δώσω μια συνολική εικόνα έχουμε 34 ε, συνδέσμους μέλη σε 22 χώρες της Ευρώπης. Έχουμε ένα πολύ ευρύ δίκτυο που λειτουργεί σε πολλά μέρη της Ευρώπης και αυτό βοηθά τις εταιρείες να μπορούν να συμμετέχουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στην διαδικασία τυποποίησης. Θα τονίσω ορισμένα επιμέρους σημεία διότι σε πολλά σημεία συμφωνούμε με αυτά που ανέφερε η Business Europe νωρίτερα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω κάποιες ιδιαιτερότητες ε, οι οποίες είναι σημαντικές για εμάς. Καταρχάς, η τυποποίηση είναι ένα εργαλείο για τις ε, επιχειρήσεις. Εάν χρησιμοποιούν την τυποποίηση οι οργανισμοί, οι οποίες καταρχάς είναι εθελοντικές, αν χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό το εργαλείο, θα βοηθήσουν τις αγορές, ιδιαίτερα τον τομέα των εξαγωγών. Ο τομέας των εξαγωγών είναι πολύ σημαντικός και αυτό κιόλας εξηγεί γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ε, επενδύσει πολύ για να διασφαλίσουν την ε, χρήση των προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα είμαι και ειλικρινής μαζί σας ανταγωνιστικά, χρειαζόμαστε να κάνουμε περισσότερα έτσι ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να είναι ανταγωνιστική στο, στην παγκόσμια αγορά. Και τα πρότυπα λοιπόν ελπίζουμε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εταιριών. Έπειτα, φυσικά, προσπαθούμε να διευκολύνουμε την συμμόρφωση με, τους, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όπως βλέπετε, έχουμε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ρυθμιστικό δίκτυο με πολλούς τομείς να αλληλοπικαλύπτονται και για μας η διαμόρφωση και η δημιουργία προτύπων λειτουργεί ως απλοποίηση της ε, νομοθεσίας ή των απαιτήσεων της νομοθεσίας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν η απλοποίηση και πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ε, πρέπει να συμμορφωθούμε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έπειτα ε, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι τα πρότυπα δεν είναι νομοθεσία. Για μας η τυποποίηση, όπως είπε και ο Πολ πριν, είναι κάτι τεχνικό, είναι τεχνική διεργασία και δεν εκτιμούμε καθόλου την προσπάθεια της ετυποποίησης να λειτουργήσει ως νομοθέτης. Αυτό την πολιτική την χαράζουν οι νομοθέτες, οι ρυθμιστές. Εμείς απλά έργο μας είναι να ερμηνεύουμε την νομοθεσία αυτή στα πρότυπα. Έπειτα δημόσιες ανάγκες ή ιδιωτικές ανάγκες. Η Business Europe πάλι μας έδωσε ένα καλό παράδειγμα το εμπόριο, όπως είδαμε, διευκολύνθηκε πάρα πολύ με την εισαγωγή του, ε, των εμπορευματικιβωτίων των 20 ποδών. Διευκόλυνε τις ε, μεταφορές και στον τομέα του ηλεκτρικού εξοπλισμού, για παράδειγμα, έχουμε και πάλι πρότυπα στις μπαταρίες. Και αυτά τα πρότυπα ε, δημιουργήθηκαν σε άλλα μέρη του κόσμου και υιοθετήθηκαν διεθνώς. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι το σύστημά μας είναι ήδη αρκετά ανοιχτό στην εισαγωγή προτύπων που δημιουργήθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου εάν αυτά τα χρειαζόμαστε και στην περίπτωση στην οποία τα χρειαζόμαστε. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, η Κομισιόν τόνισε το στοιχείο της ταχύτητας για να είμαι ειλικρινής, για μας η ταχύτητα δεν είναι αυτός σκοπός. Το πιο σημαντικό είναι η ποιότητα. Και η ποιότητα πρέπει να γίνει αποδεκτή από την αγορά. Θα ήταν παράξενο να... εάν πιστεύαμε ότι η βιομηχανία θα παράγει πρότυπα που δεν θα δεχτεί η αγορά. Δεν μπορούμε να παράγουμε λοιπόν πρότυπα που δεν θέλουν οι καταναλωτές. Δεν έχει νόημα να το κάνουμε αυτό διότι ε, εξαρτώμαστε από τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα αγοράσει τα προϊόντα μας. Και το στοιχείο της ταχύτητας διαφέρει από τομέα σε τομέα. Καταλαβαίνω ότι στον τομέα ICT οι εξελίξεις είναι ταχύτερες από ό,τι σε άλλους τομείς. Όπως για παράδειγμα στον τομέα των μηχανημάτων, όπου εκεί το... η ποιότητα είναι πολύ πιο σημαντική από την ταχύτητα. και ταχύτητα λοιπόν προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάστοτε τομέα. Τα πρότυπα Όσον αφορά τα πρότυπα ICT και τις ανάγκες για δημόσιες προμήθειες, βλέπουμε ότι τα πρότυπα αυτά είναι αναγκαία και θα θέλαμε να δούμε τα πρότυπα αυτά να εξαπλώνονται και σε άλλους τομείς. Όμως, όχι στα δημόσια κονσόρσια. Αυτό που θα θέλαμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε από, όλη αυτό, από αυτή τη συζήτηση είναι περισσότερη κατανόηση, περισσότερη, περισσότερη ευελιξία και όχι ευρωκρατικό έλεγχο. Δηλαδή, εάν θέλουμε να έχουμε μια πιο ανοιχτή πλατφόρμα εργασίας, πρέπει να, αυτή να είναι ανοιχτή σε όλους και για όλα τα πρότυπα και όχι μόνο τα πρότυπα ICT. Πιστεύω πως ακόμα χρειάζεται βελτίωση στην ε, συνένεση, στη δημιουργία συνένεσης και η διαδικασία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και διάφανη για όλους. Τέλος θα ήθελα να πω ότι οι ESO θα έπρεπε να λειτουργούν όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς καμία παρέμβαση από, δημόσια, από δημόσιους φορείς. Ευχαριστώ πολύ. Για τα τόσο σαφή αυτά παραδείγματα ήταν πολύ ενδιαφέρον το ότι και εσείς και ο συνάδελφος από την Business Europe επιλέξατε παρόμοια παραδείγματα. Εν τέλει σε αυτό το πάνελ θα ακούσουμε από ένα άλλο τομέα ο οποίος χρησιμοποιεί τα πρότυπα, πρόκειται για υγειακό εξοπλισμό. Ο Λουι Μελί, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του ΣΕΣΕΤ, θα μας παρουσιάσει τα προβλήματα αυτά. Έχετε έξι λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμβάλλω σε αυτή τη συζήτηση για ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Να σας πω ότι είναι η CCID. Εκπροσωπούμε 16 μέλη και 26 εθνικούς οργανισμούς. Έχουμε μια σχεδόν πανευρωπαϊκή κάλυψη. Ναι, λειτουργεί, λειτουργεί το μαραθέτη αυτό. Ευχαριστώ. Για μας η τυποποίηση υπήρξε πάντα ένα κομβικό στοιχείο από την αρχή της λειτουργίας μας και παρά το γεγονός ότι είμαστε ένας σχετικά μικρός τομέας, πιστεύω ότι η τυποποίηση έχει, σημάνει, έχει παίξει σημαντικό ρόλο μέσα στην λειτουργία του φορέα μας. Η παρουσία των οικιακών συσκευών σε όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά λοιπόν έχει ευνοηθεί ιδιαίτερα από την τυποποίηση θα ακολουθήσω μια κάπως διαφορετική προσέγγιση χωρίς να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου από την Digital Europe για τα προβλήματα της ταχύτητας. Είναι σημαντικό όταν μιλάμε για την ταχύτητα να έχουμε μια πλήρη προσέγγιση τυποποίησης στο μυαλό μας. Δηλαδή από μια αρχική σύλληψη ιδεών μέχρι την εφαρμογή. Υπάρχουν τρία στοιχεία. Υπάρχει η προετοιμασία, η τυποποίηση αυτή καθεαυτή <clears throat> και η συντήρηση των προϊόντων. Πιστεύω ότι η ταχύτητα εφαρμογής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σύνολη διαδικασία. Γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε σωστά την ταχύτητα αυτής της εφαρμογής των προτύπων. οι προηγούμενοι ομιλητές έχουν παρουσιάσει ήδη μερικές βασικές αρχές και μερικά ισχυρά σημεία. Να εστιάσω περισσότερο στις αδυναμίες. Υπάρχει πράγματι ένας μακρός χρονικός ορίζοντας από την αρχική ε, προετοιμασία μέχρι την εφαρμογή ενός προτύπου. Όταν εμπλέκεται λοιπόν η Κομισιόν στην εκπόνηση ενός προτύπου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και ο χρόνος προετοιμασίας ο οποίος καταδαπανείται έτσι. Δεν μπορούμε εμείς να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο από το τμήμα αυτό της διαδικασίας. Είναι απαραίτητο οι εμπλεκόμενοι να έχουν και κάποια συμβολή στη διαδικασία αυτή. Γιατί όσο μεγαλύτερη συνένεση υπάρχει στην αρχική αυτή φάση, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει υπό μορφή προτύπου. Ένα δεύτερο βασικό στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Σύρο είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία. Το γεγονός ότι οι δημόσιες αρχές εποπτείας μειώνουν την συμμετοχή τους, αυτό υποσκάπτει και την ταχύτητα αλλά και την των προτύπων. Μειώνει την εγκυρότητα των προτύπων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Όταν τα πρότυπα τα οποία απαιτούν μια σημαντική επένδυση από εμά είναι υποδιαφυσβήτηση στη συνέχεια. <clears throat> Ποιοι είναι οι κίνδυνοι τους οποίους πρέπει να αποφύγουμε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι η απόκληση μεταξύ των ευρωπαϊκών και των διεθνών προτύπων είναι όσο το δυνατόν μικρότερη γιατί αλλιώς καταλήγουμε σε μια επικάλυψη προσπαθειών και οδηγεί και σε έλλειψη ταχύτητος και έγκαιρου χαρακτήρα των προτύπων. Αν χρειάζεται λοιπόν να επανέλθουμε στα πρότυπα αυτά, διότι δεν λάβαμε υπόψη τη διεθνή εξέλιξη των προτύπων, αυτό ουσιαστικά αυξάνει την προσπάθεια και τους πόρους που πρέπει να αφιερωθούν σε αυτή τη διαδικασία και φυσικά υπονομεύει και την εγκυρότητα ενός προτύπου για τη δημόσια αγορά. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και μια ισότητα συνδικών ανταγωνισμού. Το ανέφερε και οι προηγούμενοι ομιλητές. Εάν έχουν τη δυνατότητα να ε, συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε για τα πρότυπα, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο ισότητος για όλους τους συμμετέχοντες. Επίσης, εφόσον υπάρχει δυνατότητα να διαμφισβητηθεί ένα πρότυπο, θα πρέπει να γίνεται αυτό με έναν τρόπο ο οποίος προϋποθέτει την προηγούμενη συμμετοχή. Δεν μπορεί κανείς να απόσχει από τη διαδικασία συνένεσης και μετά εκ των υστέρων να διαμφισβητεί ένα πρότυπο. Επομένως η συμμετοχή και η διαφάνεια είναι τα κέρια στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν να εξασφαλίσουν ότι έχουμε την κατάλληλη ταχύτητα εφαρμογή χωρίς να θέσουμε να αμφιβόλο την ποιότητα. Επομένως έχω αυτούς τους τέσσερι πυλώνες που είναι η ταχύτητα, η ποιότητα, η βεβαιότητα και η διεθνής ε, διάσταση των προτύπων. Σας είπα ότι η ποιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά η ποιότητα υπερέχει. Δεν μπορούμε να θίξουμε την ποιότητα λόγω ταχύτητας γιατί αυτό μειώνει την εγκυρότητα των προτύπων. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια βεβαιότητα σε σχέση με τα πρότυπα γιατί αυτό εξασφαλίζει και τη μακροβιότητα των προτύπων και τέλος όπως είπα προηγουμένως η διεθνή διάστασή τους για να είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σαφήνειά σας. Και για την ταχύτητα που επιδείξατε. Τώρα το συζητούσα εδώ με την εισηγητριά μας και μου προτείνει, επειδή υπάρχει κάποια χρονική πίεση, να περάσουμε απευθεία στο δεύτερο πάνελ για την ευρύτερη τη συμμετοχή. Και μετά να έχουμε ρωταπαντήσει από του συναδέλφου. Ελπίζω οι, οι συναδέλφοι να μπορούν να το δεχτούν αυτό, γιατί αλλιώ δεν θα προλάβουμε. Κρατήστε λοιπόν τι ερωτήσει σα. Ο κατάλογο των αγορτών είναι ακόμη ανοιχτό γιατί νομίζω ότι όλοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε για την ευρεία συμμετοχή. Και μετά, ούτω ή άλλω, η διεθνή διάσταση θα είναι ένα ξεχωριστό τμήμα. Εάν λοιπόν ο κύριο Στίβεν Ράσελ είναι έτοιμο, να προχωρήσουμε. Και εκείνο είναι γνωστό πρόσωπο ως, ε, στις συναντήσεις μας, ως Γενικός Γραμματέας της ΑΝΕΚ, που ξέρετε ότι ασχολείται με τα θέματα καταναλωτών στην τυποποίηση και ακριβώ θα εκφράσει την Ευρωπαϊκή, την φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών, ο κύριο Ράσελ, στη σημερινή παρουσίαση. Έχετε το λόγο για 6 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι, η ΑΝΕΚ δημοσίευσε τη θέση τη για το σχέδιο κανονισμού τυποποίηση ε, αρκετά έγκαιρα πιστεύω. Νομίζω την ίδια μέρα με τα γενέθλια τη κυρίας Σαντιάγκο, στις 14 Οκτωβρίου 2011. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το ίντερνετ ε, μέσω του link που θα δείτε στην οθόνη. Εδώ επιβεβαιώνουμε τη στήριξή μας ε, για την ε, ευρωπαϊκή διαδικασία τυποποίησης, αν και κάποιες φορές δεν αγγίζουμε τα υψηλότατα επίπεδα που θα θέλαμε ασφάλειας για τους καταναλωτές. Πραγματικά υπάρχουν στιγμές όπου η κανονισμοί και οι κανόνες θα έπρεπε να προτιμώνται. Αλλά αυτό το προτιμούν συνήθω οι πολιτικοί φορείς και όχι οι υπεύθυνοι τη τυποποίηση. Από τον πρώτερο βίο μου, όταν οι διάφοροι ρυθμιστέ έδιναν τις κοιτάλεις τους ε, υπεύθυνο τη τυποποίηση, αυτό ήταν σαφέ. Τώρα για το σχέδιο κανονισμού, προφανώ καλωσορίζουμε την πρόταση που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα φορέα που να εκπροσωπεί του καταναλωτέ, ο λεγόμενο φορέα του παρατήματο 3. Ξέρουμε ότι εδώ θα επικεντρωθεί ο φορέα αυτό στη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα και νομίζω ω καταναλωτέ όλοι θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε σε αυτόν τον νέο κανονισμό που θα προσφέρει ευρύτερη προστασία και ευημερία των καταναλωτών ανά την Ευρώπη. Πρόσεξα, όταν μιλήσαμε για το μέλλον της ευρωπαϊκής Τυποποίηση, ότι αναφέρθηκαν πολλές μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι οι ειδικέ γνώσεις των καταναλωτών για την ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι ε, ελλειπείς ή απουσιάζει τελείως σε κάποιε χώρε. Η απουσιαζει τελειω σε βεβαίω είναι βεβαιω ειναι όπως και κάποιες άλλες χώρε, αλλά μόνο αυτέ. Ακριβώς για αυτό το λόγο η διεθνής προσέγγιση, εάν και αναγκαία, δεν επαρκεί. Δεν αρκεί να εκπροσωπούνται όλα τα, για να όλα τα συμφέροντα στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Ο φορέας του παρατήματος 3 συμπληρώνει τις εθνικές αντιπροσωπείες εν Σένελεκ και διασφαλίζει το ότι οι εθνικές πλατφόρμες θα καθορίζουν το κατά πόσο εύστοχα θα είναι τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Από την προηγούμενη ακρόαση έγινε μια μελέτη για τα θέματα των καταναλωτών που επιβεβαιώνει την ανάγκη να εκπροσωπούνται τα συμφέροντα των καταναλωτών των περισσότερων κατών μελών στη διαδικασία διαμόρφωση των προτύπων. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γνωρίσουμε την έτσι, αλλά κάποιε φορέ πρότυπα όπω αυτά για τα GSM κάνουν τη ζωή των καταναλωτών πιο εύκολη. Οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώ θα προστατεύεται καλύτερη ασφάλεια και ευημερία των καταναλωτών. Βεβαίω υπάρχουν προτάσεις για συμμετοχή, συμμετοχή στο σύστημα των ε, προτύπων, αλλά σε οικειοθελή βάση. Οι αποφάσεις των ενδιαφερομένων γίνεται βάσει των προτεραιοτήτων και των αναγκών των ε, ιδίων. Εάν λοιπόν ε, οι δημόσιοι φορείς μπορούν να διασφαλίσουν τα πρότυπα, και τη χρηματοδότησή του, τότε θα πρέπει να βρουν και μια εναλλακτική γραμμή παραγωγής, όπως αναφέρει η ΣΕΝ, ΣΕΝΕΛΕ και η ΕΤΣΙ. Δεν συμφωνούμε λοιπόν εδώ με το σχέδιο πρόταση κανονισμού να να αξιολογούνται μάλλον οι φορεί εκπροσώπηση των καταναλωτών ανάλογα με το έργο του. Η εκπροσώπηση χωρί την ε, δυνατότητα επιρροή δεν έχει κανένα νόημα. Οι φορεί του παρατήματο 3, όπω προτείνονται, είναι μόνο παρατηρητέ ε, στα τεχνικά σώματα τη ΕΝ και τη ΕΝΕΛΕΚ. Παρά το ρόλο του στη συμπλήρωση των εθνικών αντιπροσωπιών, όπω του προτείνει ο κανονισμό, δεν μιλά καθόλου για την πραγματική ε, την ουσιαστική συμμετοχή, όπως ε, πρότεινε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, την πρότασή του του Οκτωβρίου του 2010. Εδώ λοιπόν αυτό που θεωρούμε ότι είναι καλύτερο για τους ευρωπαϊκούς φορείς είναι να αξιολογούνται βάσει της πραγματική συμμετοχή. Όμω, γιατί χρειάζεται αυτή η πραγματική συμμετοχή. Α σκεφτούμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του ε, προτύπου για τα το μοτοποδήλατα. Αυτά τα οχήματα μπορεί να είναι επικίνδυνα, ε, να σκοτώσουν και πολλές φορές έχουν προκαλέσει απώλειες. Δεν είναι παιχνίδια. Δεν μπορώ να σας δώσω, μάλλον θα μπορούσα να σας δώσω συγκεκριμένα αριθμούς από τη στατιστική βάση για τα ατυχήματα όπω και η κυρία Σαλντεμόζα, αλλά 7 θανάσιμα ατυχήματα τουλάχιστον ε, σημειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 2004 και 2006. Και πρόσφατα αυξήθηκαν τα σχετικά ατυχήματα ανά τον κόσμο. Τα περισσότερα μάλιστα αφορούσαν παιδιά. Επειδή λοιπόν τα μοτοποδήλατα ακριβώ ε, είναι ευρέω διαδεδομένα και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα, πρόσφατα δημιουργήθηκε σχετικό πρότυπο. Δεν υπάρχουν όμως όρια για αυτά τα μήνυμο τοποδήλατα που να αφορούν την ηλικία και την ταχύτητα πέραν του βασικού προτύπου της ΑΝΕΤ. Ε, Έτσι λοιπόν, εάν υπήρχε εδώ κάποια αντίρρηση, κάποια διαφωνία από, μια εθνική, από έναν εθνικό φορέα εκπροσώπησης των προτύπων, τότε μπορεί να μην είχε ψηφιστεί το πρότυπο αυτό. Το μόνο που έχει ψηφιστεί ω κανόνα είναι ότι θα πρέπει τα αυτά μοτοποδήλατα να μην χρησιμοποιούνται από παιδιά κάτω των 6 ετών. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους φορείς του παρατήματος 3 αλλά όχι να ενισχυθεί ο κεντρικό χαρακτήρα όπω προτείνεται από το παράρτημα αυτό και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο με την ψήφο του να μην ενισχύσει αυτήν την τάση, αλλά να παραμένουν και τα εθνικά κράτη στο ρόλο του. Έτσι κι αλλιώ το δικαίωμα ψήφου θέλουμε να παραμείνουμε, χωρί να έχει κανεί βέβαια το δικαίωμα έρνηση κυρία, αλλά τουλάχιστον η αρχή τη διαφωνία να μπορεί να γίνει σεβαστή, όπω έγινε στην περίπτωση των μήνυμα των ποδηλάτων. Και για να κλείσω, πιστεύουμε ότι η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να αφορά το δυνατόν περισσότερου συνομιλητέ, να είναι ανοιχτή στου ευρωπαϊκού φορεί ανά το ευρύτερο οικονομικό φάσμα τη ευρωπαϊκή αγορά και να εκπροσωπεί το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίηση, ώστε τα ζητήματα τυποποίηση να συζητούνται στο κατάλληλο πλαίσιο με, τις ανάλογες, με του ανάλογου ρυθμιστικού στόχου. Θα παραμένω σε αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ήταν ε, πολύ ε, εύστοχη η παρουσίασή σα και πολύ σαφή η θέση σα. Ευχαριστούμε λοιπόν για όλα αυτά. Τώρα θα προσκαλέσω τον Ραλφ Λότε, Γενικό Γραμματέα Τη Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Οργάνωση για του πολίτε και την Τυποποίηση και ο οποίο είναι ενεργότατο μέλο στην όλη διαδικασία τη τυποποίηση να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο για έξι λεπτά. Ε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Κόμη για την πρόσκληση στην σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ τα μέλη του Κοινοβουλίου. Αγαπητά μέλη, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σα ε, πω την γνώμη του ΙΚΟΣ που αντιπροσωπεύει τα, τους περιβαλλοντικούς ε, Έχουμε 25 οργανισμούς μέλη σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρυθήκαμε το 2001 για να αντιπροσωπεύσουμε τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ στην τυποποίηση. Έχουμε εμπειρογνώμονες και προσπαθούμε λοιπόν να επιτύχουμε συνένεση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να πάτε στην ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες. Στην σελίδα της Ίνκο θα βρείτε επίσης και το πλήρες έγγραφο που αναλύει τις θέσεις μας. Λοιπόν, η ΕΚΟΣ υποστηρίζει έντονα την πρόταση της Κομισιόν και για μας το κύριο άρθρο είναι το άρθρο 5, διότι ενσωματώνει την κατάλληλη αντιπροσώπηση στην διαδικασία τυποποίησης μπορούμε να συζητήσουμε αν θα πούμε κατάλληλο, ισορροπημένο ή κάτι άλλο, όμως πιστεύουμε πως ε, όπως και να έχει είναι θεμελιώδης ε, η συμμετοχή στην τυποποίηση. Επίσης να ορίσουμε τι είναι κατάλληλο, τι είναι ισορροπημένο, τι χρειάζεται. Να δούμε ότι χρειάζεται η εφαρμογή της αρχής αυτής και επίσης ότι δεν είναι και εύκολο. Γιατί χρειάζεται αυτοί οι οργανισμοί να αντιπροσωπεύονται κατάλληλα. Για μα ένα σημείο είναι η αρχή τη εθνική αντιπροσωπευση. Είναι μια βασική αρχή του οργανισμού μα, όμω δεν λειτουργεί για αυτή την ομάδα ενδιαφερομένων. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Οι περιβαλλοντικέ ΜΚΟ συστηματικά αντιπροσωπεύονται σε μόνο ένα κράτο μέλο τα τελευταία 15 χρόνια, στη Γερμανία. Μόνο εκεί αντιπροσωπεύονται. Από τότε και χάρη σε ένα επιτυχημένο project ε, συμμετέχει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και γιατί υπάρχει αυτή η απουσία. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Πιστεύουμε ότι δύο από τις 31 χώρες μέλη του ΣΕΝ και του ΣΕΝΕΛΕΚ δεν πιστεύουν ότι είναι κατάλληλη αντιπροσώπευση ή ισορροπημένη αντιπροσώπευση. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι χρειάζεται μία ε, διόρθωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να συμμετέχουν και αυτοί οι ενδιαφερόμενοι θα ήθελα να σα εξηγήσω τι σημαίνει η αρχή τη εθνική αντιπροσώπευση. Σημαίνει ότι σε εθνικό επίπεδο για ένα συγκεκριμένο θέμα όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχή, να συζητήσουν, να ακουστούν και οι εθνικέ αυτέ επιτροπέ ε, φέρνουν στην ΣΕΝ και τη ΣΕΝΕΛΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι εθνικέ θέσει στι οποίε ε, συμμετείχαν και οι εθνικοί φορεί και ενδιαφερόμενοι. Όπω είπαμε, μόνο σε μία και τώρα σε δύο χώρε αντιπροσωπεύονται επαρκώς οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Ε, πρόεδρος, μπορείτε να συνεχίσετε με, τα, με τις διαφάνειες. Ναι. Τι σημαίνει για μας επαρκής αντιπροσώπευση. Καταρχάς η απώλεια εμποδίων. Υπάρχουν δυστυχώς ε, κάποια εμπόδια σε ορισμένα τυπο, σώματα τυποποίησης Επίσης, η ιδιότητα του μέλους, όπως είπε και ο συνάδελφος Ράσελ, είναι ιδιαίτερα σημαντική και φυσικά είναι σημαντικό να πάμε από την αντιπροσώπευση στην πραγματική άσκηση επιρροής. Έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των περιβαλλοντικών ΜΚΟ συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα για τα περιβαλλοντικά συμφέροντα υπάρχουν αρκετά εργαλεία έτσι ώστε να ε, ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές ε, ΜΚΟ στην ε, διαδικασία τυποποίησης. Δυστυχώς το περιβάλλον ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί ολοκληρωτικά σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν ορισμένα εργαλεία που έχει δημιουργήσει η ΣΕΝ και πιστεύουμε ότι θα δώσουν παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών και θα πρέπει να εφαρμοστούν και από άλλα σώματα. Τέλος, τα στάδια της αντιπροσώπευσης. Πιστεύουμε ότι το άρθρο 5 υπογραμμίζει την ε, ανάπτυξη των σταδίων πάρα πολύ καλά και πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτά. Ωστόσο υπάρχει ένα που λείπει και είναι πολύ σημαντικό, το στάδιο της ψηφοφορίας. Δηλαδή, το πέρασμα μιας ε, διαδικασίας ενός προτύπου από το ένα στάδιο στο άλλο με οριστική ε, και τελική ψηφοφορία πριν τη δημοσίευση. Επίσης, η εκτίμηση δικτύπου της ΕΣΥ, της Επιτροπής, δεν ε, βλέπει κάποιες, ε, κάποια ε, δύσκολα σημεία, απλά διερωτάται για το πόσο εφικτή είναι η εφαρμογή. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι πραγματικά θα έπρεπε να υπάρχουν όρια για τους δικαιούχους των δικαιωμάτων ψηφοφορίας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο οργανώσεις ενδιαφερομένων οι οποίες έχουν συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία δημιουργίας των προτύπων και επίσης ε, όσον αφορά τον χρόνο, εάν ένας, ε, ένας οργανισμός δεν έχει, δεν, δεν έχει ασχοληθεί συστηματικά με την διαδικασία τυποποίησης, δεν θα έπρεπε να έχει δικαίωμα ψηφοφορίας. Θα έπρεπε να το έχει μόνο εάν ασχολείται συστηματικά και σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, όσον αφορά το άρθρο 12, η χρηματική υποστήριξη όπως ήδη έχει αναφερθεί, υπάρχει ανάγκη για ταχύτητα για να γίνει αυτό γρήγορα και τέλος πιστεύω ότι θα έπρεπε να ε, δούμε τις ε, εσωτερικές διαδικασίες των ε, ευρωπαϊκών οργάνων για να δούμε πώς θα επιταχυνθεί η διαδικασία. Και όσον αφορά την επέκταση της τυποποίησης σε άλλους τομείς πολιτικής, για παράδειγμα την αποδοτικότητα των πόρων και την κλιματική αλλαγή, Πιστεύουμε ότι η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην άσκηση πολιτικής είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε, έχουμε ανάγκη την υποστήριξη του JRC στην διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Οι συστάσεις ήταν ξεκάθαρες και να έχουν άμεση, άμεση σχέση με το ΑΝΕΚ. Τώρα, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνδικάτων έχουμε τον Στέφανο Μπόι που θα μας μιλήσει και θα μας μιλήσει για τις απόψεις ε, του Ινστιτούτου Συνδικάτων. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια Κόμη για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαίρουμε καταρχάς την Επιτροπή για την εξαιρετική πρόταση η οποία έχει, βρίσκεται ενώπιον σας μετά από πολλή δουλειά πολλών εμπειρογνωμόνων και όλα αυτά τα έγγραφα που έχετε αναφέρουν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση στην ε, δημιουργία των προτύπων. Θα ήθελα να προτείνω να προχωρήσουμε σε, από κάτι ανοιχτό σε κάτι κλειστό έτσι ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη σύνδεση των παραγωγών και των χρηστών των προτύπων. Αυτό που εμείς πιστεύουμε και οι θέσεις μας βασίζονται σε 15 χρόνια δουλειάς. Τα συνδικάτα άρχισαν να εργάζονται στον τομέα της τυποποίησης με δύο στόχους. Καταρχάς την ανάλυση του αντικτύπου των προτύπων στους εργάτες και έπειτα προσπαθώντας να συνεισφέρουν στην δημιουργία λύσεων για τα προβλήματά τους. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τις εμπειρίες μας πάνω και τις ε, αντιρρήσεις. Η εμπειρία μας δεν διαφέρει από εκείνη της, ε, δημόσιας, της αρχής ε, δημόσιας επιτήρησης. Η δημιουργία προτύπων δεν μπορεί προς το παρόν να θεωρηθεί επαρκής μηχανισμός για να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις. Η διαδικασία θα δείτε ότι είναι πολύ περίπλοκη. Στο θα δείτε ότι για να φτάσει κάτι από το πρόβλημα ως την επίλυση με τη διαδικασία προσήπων χρειάζονται τρία χρόνια. Πολύ καιρός. Το κύριο ζήτημα και η κύρια ανησυχία μας είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο δίκτυο ασφαλείας για, για τον μεγάλο αριθμό προτύπων που παράγονται εκτός αυτής της προσέγγισης. Και αν δείτε το σχέδιο δράσης της Κομισιόν, θα δείτε ότι υπάρχουν ελάχιστες, ε, ε, ελάχιστοι τομεί πολιτικής που υποστηρίζονται από την ε, οδηγία της προσέγγισης. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η τυποποίηση έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά και στους πολίτες, στους καταναλωτές και στο περιβάλλον. Επομένως, ε, στους τομείς όπου δεν υπάρχουν επίσημες ε, αντίρρησεις χρειάζεται να σχεδιαστεί ένας μηχανισμός έτσι ώστε να δοθεί στις ε, δημόσιες αρχές και σε όλους τους ενδιαφερομένους η δυνατότητα να αμφισβητήσουν αυτά τα υπάρχοντα πρότυπα. Και εδώ, με, εδώ θα συνδεθώ με την έκθεση IMCO. Εάν διαβάσετε την έκθεση πάνω από μία φορά, θα δείτε ότι εύκολα συνειδητοποιούμε ότι ότι εάν εφαρμοστεί, εφαρμοστούν οι συστάσεις της ΙΝΚΟ στο υπάρχον σύστημα θα πάμε από αυτό το σύστημα σε αυτό που βλέπετε τώρα στη διαφάνεια. Είναι μια σχηματική επικόνηση ορισμένων συστάσεων της ΙΝΚΟ και θα δείτε πόσο κεντρικός είναι ο ρόλος μιας πλατφόρμας πολλών ενδιαφερομένων όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Πρόεδρε, θα ήθελα να, να τονίσω ότι αυτό που βλέπετε προκύπτει άμεσα από την σύσταση της ΣΥΜΚΟ και δεν έχουμε πειράξει τίποτα. Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα, η ουσία όμως είναι η ίδια. Και αφού είναι ακόμα απεικόνηση, θα ήθελα να καλέσω τους ενδιαφερόμενους και την εισηγήτρια να το λάβουν ως σημείο εκκίνησης. Αυτό ο κατάλογος είναι μόνο ενδεικτικός των ε, συστάσεων των συνδικάτων. Αλλά, κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σε μια εποχή που κάνουμε περικοπές στον προπολογισμό σε όλη την Ευρώπη και οι επιπτώσει είναι ότι οι αρχές δεν δύναται να συμμετέχουν σε, στους, ε, σε, στους τομείς της προτυπωποίησης. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα χρηματοδότησης. Όμως πρέπει να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε τους ε, μικρότερους ενδιαφερομένους. Θα σας δώσουμε όμως λεπτομερώς τις δικές μας προτάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για τις συστάσεις σας λοιπόν. Θα τα λάβουμε υπόψη μας ιδιαιτέρως. Όλα αυτά δείχνουν τη σημασία της προπαρασκευαστικής εργασίας που πρέπει να προηγηθεί της ε, πολύπλοκης νομοθετικής διαδικασίας. Ένας άλλος φορέας ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο έργο μας τα τελευταία χρόνια είναι η Norm Arme, APME, που γνωρίζετε πολλοί από εσά, η οποία έχει συμβάλει ιδιαίτερα από την ε, οπτική γωνία της, ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κύριος Τίλμαν είναι, το, είναι ο Γενικός Γραμματέας της και τον καλό να λάβει το λόγο για 6 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ακόμη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Όπως ξέρετε, ο φορέας μας είναι γνωστός και στις Βρυξέλλες και στην Ευρώπη. Θα ήθελα στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα να σας εξηγήσω για τον οργανισμό μας. Δημιουργηθήκαμε το 1946 και η Κομισιόν και οι άλλοι φορείς οι οποίοι ίδρυσαν αυτόν τον οργανισμό τόνισαν τη σημασία, είχαν τονιστό τη σημασία τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τυποποίηση. Small is beautiful είναι το γνωστό σύνθημα, κάτι που είναι μικρό και όμορφο. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα μικρό όμω, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω σε αυτό το σύνθημα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτουν 98% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Μαζί με τους οργανισμούς που θεσπίζουν πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις Βρυξέλλες, αλλά και με τους φορείς που βρίσκονται στην Σοφία Αντίπολη στη Γαλλία, είναι πολύ σημαντικό ότι μπορέσαμε να συνεργαστούμε με φορείς βιομηχανικούς σε όλη την Ευρώπη και μπορούμε να ασχοληθούμε με την εντατική προώθηση των θεμάτων αυτών και την παρότρινση της όλο και μεγαλύτερης συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο γίγνεσθε το ευρωπαϊκό για τη δημιουργία τυποποίηση. Είμαστε μια οικογένεια, νιώθουμε σαν οικογένεια και γι' αυτό εμείς έχουμε χαιρετήσει το πακέτο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για την τυποποίηση, την ανακοίνωσή της και το σχέδιο οδηγίας που έχουν πρόσφατα δημοσιευτεί. Είμαστε μια πολυπληθής οικογένεια και είναι πολύ δύσκολο σε μια τέτοια οικογένεια να έχει κανείς μια εύκολη διαδικασία σφυριλάτησης κοινών θέσεων. Μόνο στα τέλη Οκτωβρίου μπορέσαμε να ε, οριστικοποιήσουμε τη διαδικασία για την λήψη αποφάσεων και έχουμε στείλει όλα αυτά τα στοιχεία στα μέλη μας. Αν θέλετε μπορούμε να σας δώσουμε και σε εσά περαιτέρω στοιχεία για αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πακέτο αυτό τυποποίηση. Το πακέτο αυτό τη Κομισιόν εξάλλου αναγνωρίζει εκπεφρασμένα την ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο, να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή ω τμήματα τη ευρωπαϊκή οικονομία στι διαδικασίε αυτέ τυποποίηση. Θα ήθελα τώρα να σα δείξω πού βρισκόμαστε. Δεν λειτουργούμε σε εθνικό επίπεδο, λειτουργούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι και ο Ρομπ Στίλ εδώ, γιατί θέλω να τονίσω ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε πάντα εστραμμένοι προς το μέλλον. Αυτό κύριε Πρόεδρε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δούμε το μέλλον γιατί βλέπουμε ότι τα διεθνή πρότυπα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία και ακόμα περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αρχή της εθνικής αντιπροσωπείας, μια αρχή που αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές, αποτελεί βέβαια πυλώνα του συνολικού συστήματο. Είτε το θεωρεί κανείς κανεί στοιχείο. Λειτουργεί αυτή η αρχή. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει όταν συμμετέχουν εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω, κύριε Πρόεδρε, είμαι Γερμανός βέβαια, αλλά θέλω να αναφέρω και το παράδειγμα της Ολλανδίας, το παράδειγμα της ΝΕΜ και θεωρώ ότι τα παραδείγματα αυτά είναι πολύ καλά και πρότυπα τα οποία θέλουν και άλλοι να μιμηθούν μέσα στην ευρωπαϊκή διαδικασία τυποποίηση. λειτουργία λοιπόν και η, η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόσο σε εθνικό ευρωπαϊκό όσο και διεθνέ επίπεδο είναι κάτι το οποίο εμεί το υποστηρίζουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική συμμετοχή χωρί τη δυνατότητα ψηφοφορία χωρί τη συμμετοχή στη λήψη απόφαση. Το να έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει το δικαίωμα να ψηφίζουν και να λαμβάνουν μέρο στι αποφάσεις θα εξάρει και την ε, σημασία της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό διεκδικούμε και δικαιώματα ψήφου στη λήψη απόφαση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές της αγοράς. Δεν μας εντυπωσιάζει λοιπόν μονάχα η ταχύτητα, η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Θα πρέπει να γνωρίζετε, να έχετε επίγνωση του γεγονότος ότι τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει τη σημασία, σημασία την ποιότητα. Είναι σημαντική η ταχύτητα, το δεχόμαστε και οι οργανώσεις μας συμμερίζονται αυτή την άποψη, αποτελεί ένα τμήμα από την αντιμετώπιση μας. Οι φόρεις μας λοιπόν στην Norm APME πάντα συμμετέχουν στην ε, διαδικασία αυτή. Έχουμε πάρα πολλές συζητήσεις στα κράτη-μέλη μας. Θέλουμε σε κάθε τομέα υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών να υπάρχουν πρότυπα. Αυτή είναι μια ανοιχτή ακόμα συζήτηση, δεν έχει επιληθεί. Μπορείτε να δείτε όμως τη θέση μας στο διαδίκτυο και θα κατανοήσετε ότι υπάρχει μια ευρεία συζήτηση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το θέμα αυτό. Όταν μιλάμε τώρα για εθνικούς φορείς. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε πάντα σε επαφή με αυτούς τους φορείς. Δεν είμαστε πάντα επιτυχείς για τα θέματα αυτά. Το 2010 και το 2011 δεν υπήρξε πάντα η απαραίτητη συμμετοχή. Ένα άλλο στοιχείο όμως το οποίο είναι σημαντικό, όπως είπαμε το να είναι κανείς κοντά στην αγορά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα νέα προϊόντα, για τις νέες υπηρεσίες είναι απαραίτητο το να έχουμε <clears throat> προσαρμογή στα πρότυπα για να είναι επιτυχής η δραστηριότητα μια επιχείρηση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσει θέλουν να επιτύχουν την επιτυχία στον τομέα αυτό και βοηθήστε παρακαλώ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να είναι πιο ανταγωνιστικές. Για να κλείσουμε τώρα την, ε, το πάνελ αυτό, έχουμε πάλι δύο μιλητέ που εστιάζουν σε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Ζαν Μάρκ Λεπάρκο από τη γαλλική κυβέρνηση που θέλει να μας παρουσιάσει το έργο της Γαλλίας για να εμπλέξουν περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διαδικασία τυποποίησης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία σας και την εμπειρία που θα μας μεταφέρετε και σας δίνω για έξι ολόκληρα λεπτά το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω συλλογικά έχουμε ευθύνη εναντί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αντιγευτολή με τους μεγάλους ομίλους οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν ειδικέ υπηρεσίες που να ασχολούνται με τα πρότυπα, ούτε καν ε, υπάλληλο για το θέμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να του εξηγούμε ότι η τυποποίηση είναι κάτι το σημαντικό και να έχουν και πραγματική συμμετοχή στην όλη προσπάθεια. Να σα πω τι έχουμε κάνει στη Γαλλία ω τώρα για να παροτρύνουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία τη τυποποίηση και μετά να διεξάγουμε κάποια συμπεράσματα και κάποιε συστάσει ίσω για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρία μέτρα λάβαμε βασικά στη Γαλλία. Το πρώτο ήταν πριν από δύο χρόνια όταν αναθεωρήσαμε το σύστημά μας, την νομοθεσία μας για την τυποποίηση, κάτι που συμβαίνει τώρα και στην Ευρώπη. Καταργήσαμε τα τέλη εισόδου για τις επιχειρήσεις στην όλη διαδικασία, στο όλο σύστημα τυποποίησης. Διότι κάποια στιγμή πρέπει να πληρώνουν οι μικρόμεσες επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν στον καθορισμό των προτύπων. Δεν ήταν πολύ αυξημένα τα τέλη βέβαια, κάποια στιγμή όμως τα καταργήσαμε πλήρως. Αυτό είχε ψυχολογικό αντίκτυπο. Όταν σαν να λέμε στις επιχειρήσεις καλο... είστε καλοδεχούμενοι στην όλη προσπάθεια. Ελάτε. Και έτσι αυξήθηκε κατά 25% η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις εργασίες τυποποίησης. Δεύτερο μέτρο εργαστήκαμε επί του κόστους, του βασικού κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή ο χρόνος επένδυσης που απαιτείται στις εργασίες τυποποίησης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή και διεθνές υπάρχουν και τα έξοδα της μετακίνησης, αλλά και ο άνθρωπος που λόγω των εργασιών της τυποποίησης χάνει από το χρόνο εργασίας του την ίδια την επιχείρηση επειδή βρίσκεται στο πόστο του. Το 5% λοιπόν του κόστους αυτό αποφασίσαμε να το καλύπτουμε τον, τα έξοδα μετακίνησης και το χρόνο εργασίας των ανθρώπων που ασχολούνται με την τυποποίηση. Προβλέψαμε λοιπόν κάτι τέτοιο με την, ε, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά με μια μεγάλη διαφορά ότι ομαδοποιούνται οι μικρομεσαίε για να ε, λάβουν αυτέ τι επιστροφέ. Δεν μπορούμε κι εμεί να διασπείρουμε όλη την προσπάθεια. Φροντίσαμε να γίνονται όλοι ένα σύνολο. Δεν μπορεί όλοι να πηγαίνουν να ασχολούνται ξεχωριστά με την τυποποίηση του ε, παροτρύναμε να οργανωθούν σε μια ένωση ανα πολλές μικρομεσαίες. Έτσι μπόρεσαν να υποφεληθούν από το δικό μας σύστημα βοήθειας, βέβαια με μια σχετική απογοήτευση, γιατί όταν δεν ήταν αρκετοί τους λέγαμε βρείτε μας κι άλλους και ξαναελάτε. Τελικά ήρθαν σε εμά και από την πείρα που έχουμε αποκομίσει από την παροχή αυτής της βοήθειας είναι ότι τελικά μας ευχαριστούν. Μας λένε ευτυχώ που συγκεντρωθήκαμε πολλές μικρομεσαίες μαζί για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να βρούμε κοινέ θέσεις και προφανώς η, η, η, η Ένωση μάλλον κάνει τη δύναμη, ισχύει τη ενώση. Πραγματικά οι επαγγελματικέ λοιπόν ενώσει έχουν ένα ρόλο εδώ να διαδραματίσουν στην συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά το σημαντικότερο είναι να εμπλακούν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Όχι να γίνουν ε, κατεχώρηση και να ληφθούν κατεχώρηση αποφάσει για αυτού. Ε, να είναι άμεση η συμμετοχή του στην ε, πρόοδο των εργασιών. Αυτό ήταν το δεύτερο μέτρο μα. Και το τρίτο ήταν στα πλαίσια του, εθνούς, του εθνικού μας φορέα τυποποίησης, της ΑΦΝΟΡ, να προβλέψουμε ειδική επιτροπή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες. Αυτή η επιτροπή τα πηγαίνει πολύ καλά, διότι παρακολουθεί το σύνολο των προδιαγραφών και προτύπων που ετοιμάζονται, προτείνονται ή μελετώνται και εντοπίζει αυτέ που ιδιαιτέρω μπορεί να ενδιαφέρουν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Τι ειδοποιεί λοιπόν, του λέει προσοχή. Εδώ μπορεί να υπάρχει ένα θέμα που σα αφορά άμεσα. Είναι ένα έργο διαλογή αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τι μικρομεσαίε. Δεν μπορούν οι μικρομεσαίε καθημερινά να παρακολουθούν την εξέλιξη των προτύπων, άρα αυτό είναι πολύ εύστοχο. Ε, Τα αποτελέσματα τώρα τι συμπεράσματα μπορούμε να διεξαγάγουμε για το ευρωπαϊκό επίπεδο και τι μα ενδιαφέρει από όλα αυτά τα παραδείγματα. Το πρώτον, πρέπει να συνεχίσουμε να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να θεσπίζουν μηχανισμού που να ενθαρρύνουν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στη συμμετοχή. Αυτό το Ευρωκοινοβούλιο το έχει κάνει επανειλημμένω με τι διάφορε ε, με τα διάφορα ψηφίσματα που έχει εγκρίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να κάνει κάτι ανάλογο και στις επιτροπές μας έχουμε πολύ συχνά συμμετοχή από άλλα εθνικά κοινοβούλια που μας λένε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο, να βοηθήσουμε κάτι ανάλογο στα υπόλοιπα κάτι μέλη. Μα και εμείς αυτό θέλουμε. Είναι σημαντική η διάδοση αυτών των ιδεών ακριβώς για όσους δεν κάνουν ακόμη τίποτα. Και είναι σημαντικό να δώσουμε το ρόλο στο άλλα κράτη-μέλη και να τους πούμε τι κάνετε για το θέμα αυτό, ώστε να τους παροτρύνουμε. Δεύτερο σημείο, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μπορέσει, να προβλέψει ένα κόστο ε, κάλυψη το κόστου για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάτι έστω ω μια μικρή επιστροφή, κάτι σαν αυτό που γίνεται στη Γαλλία. Να υπάρχει μια συγχρηματοδότηση δηλαδή από τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν ώστε να μπορεί ε, να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει να έχουν ένα συμπλήρωμα για τη συμμετοχή του στην όλη προσπάθεια. Αυτό θα μπορούσε να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και κάτι ακόμη σημαντικότερο, να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίες να εντοπίζουν τα θέματα που του αφορούν άμεσα. Εδώ νομίζω και εσεί, συνάδελφοι, έχετε έναν ρόλο πολύ σημαντικό να διδραματίσετε. Πολύ καλά ε, ε ειδοποιείτε τι μικρομεσαίε για αυτά που του αφορούν. Όμως θα πρέπει μετά να παροτρύνονται και από το εθνικό επίπεδο οι μικρόμεσες επιχειρήσεις και όχι μόνο να απευθύνονται χάρη σε εσά τα εθνικά κοινοβούλια για να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι όμως λύση το δικαίωμα ψήφου, φοβάμαι. Φοβάμαι ότι αυτό τελικά μπορεί να πάρει κάθε ευθύνη από τις μικρόμεσες επιχειρήσεις, γιατί καταλήγουμε να λένε ίσως στο μέλλον ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με τι ομάδε εργασία, δεν χρειάζεται να συμμετάσχουμε, θα υπάρξει ψήφο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι λοιπόν το αντίστροφο ακριβώ από αυτό που θέλουμε. Εμεί τι θέλουμε, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να πηγαίνουν στι ομάδε, να συμμετέχουν, να παρακολουθούν αυτά που συμβαίνουν. Δεν θέλουμε στη θέση του να λαμβάνονται αποφάσει, να γίνονται οι διαδικασίε, να τι ειδοποιούμε, αλλά να μην συμμετέχουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα και προ το δικό σα το φορέα και προ όλου του άλλου οργανισμού. Πρώτη ειδοποίηση, πρώτο μήνυμα ειδοποίηση ναι, αλλά μετά ισχυροποίηση των ίδιων. Διότι αν είμαστε 25 κράτη-μέλη και α, ε, συμμετέχουν στην ομάδα μικρομεσαίε επιχειρήσει από 25 κράτη-μέλη που έχουν τι ίδιε θέσει σε εθνικό επίπεδο, καταλαβαίνετε πόσο ωφέλιμο θα είναι αυτό για τι ίδιε τι μικρομεσαίε. Σταματώ εδώ. Αυτά ήθελα να πω λίγο πολύ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη μα για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι έτσι μόνο θα καλλιεργήσουμε πραγματικά την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως μας δώσατε μια εισφάθος θέση για την εμπειρία σας στις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το να μοιράζετε κάποιους στις πρακτικές το θεωρούμε πάρα πολύ καλό. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που τώρα θα σας ε, παρουσιάσω την τελευταία παρουσίαση είναι από μια μικρή και μαχαία επιχείρηση που είναι άμεσα αναμεμειγμένη σε αυτό. Ο κύριος Φρανκ Τόρστεν, Γενικός Διευθυντής της Κοροκόρτ, θα σας ενημερώσει για τα SpaceNet. Ίσως λοιπόν κύριε Τόρστεν θα μπορούσατε να συμπληρώσετε την παρουσίαση του προηγούμενου συνομιλητή και ε, να μας δώσετε τις εμπειρίες σας για την διαδικασία τυποποίησης. Χαίρομαι πολύ που σήμερα έχω τη δυνατότητα να σας μιλήσω εκ μέρους της Κοροκόρτ, να σας μιλήσω για την τυποποίηση. Θα σας μιλήσω λίγο για την εταιρεία μας. Είμαστε βασισμένοι στο Βερολίνο και στην Τσεχία έχουμε 46 υπαλλήλους και ο κύκλος εργασιών μας είναι 10,5 εκατομμύρια. Φτιάχνουμε εξοπλισμό παιδικό, για παιδικές χαρές Ίσως έχετε δει, αν έχετε παιδιά ή εγγόνια, τα σχοινιά που παίζουν στις παιδικές χαρές. Η τυποποίηση για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα ε, το πρότυπο EN 1176 για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς. Υπάρχει το πρότυπο αυτό από το 1998 και μας έχει δώσει πολλές δυνατότητες και έχει κάνει την ε, εργασία μας πιο εύκολη όσον αφορά την κατασκευή των εξοπλισμών. Καταμερίζουμε τις ε, εργασίες μας στην Κοροκόρντ. Τώρα, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ε, και συμφωνώ μαζί του, εάν μια επιχείρηση συμμετέχει στη διαδικασία τυποποίηση, πρέπει να έχει κάποιο όφελος ε, από αυτό, διαφορετικά δεν έχει νόημα. Δυστυχώ, οι περισσότεροι δεν δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία τυποποίηση. Οι δημοκρατικές διαδικασίες δεν είναι τόσο διάφανες. Οι διαδικασίες αυτές συνήθως γίνονται από τις ανώτερες ε, διοικητικές θέσεις και σε εθνικό επίπεδο Σε εθνικό επίπεδο οι συνεδριάσεις για, τις, ε, για την ε, τυποποίηση λαμβάνουν χώρα μόνο κατά τη διάρκεια μίας ημέρας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως κρατούν περισσότερο. Όσον αφορά το κόστος, το κόστος ε, στην εθνικό επίπεδο, για μας για παράδειγμα, ανέρχεται σε 5.000 ευρώ το χρόνο για τα διάφορα έξοδα μετακίνησης. Όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα έξοδα μετακίνησης είναι πολύ ψηλότερα, 4 ή 5 φορές περισσότερα. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πιστεύω ότι είναι λογικό να συμμετέχουν στη διαδικασία τυποποίησης. Καταρχάς θα παρέχουν τις δικές τους εμπειρίες και θα παρέχουν επίσης χρήσιμες πληροφορίες ε, σχετικά με το ποιες αλλαγέ πρέπει να γίνουν. Να παρέχουν επίσης την ε, εμπειρία τους από την, επαφή, την άμεση επαφή με τους καταναλωτές. Όπως και για εμάς και στη δική μας περίπτωση. Επίσης, έχουν επιρροή στην δημιουργία των προτύπων και δεν κάθονται απλά ως ε, παρατηρητές. Κάτι που ίσως δεν είναι γνωστό είναι το στρατηγικό στοιχείο της διαδικασίας προτυποποίησης. Το κόστος για την αλλαγή των προτύπων σε κάποιο προϊόν μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλό και ίσως δεν, είναι, ε, δεν έχει πλεονεκτήματα και δεν έχει όφελος για κάποια εταιρεία όταν το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Πολλές φορές ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Επίσης υπάρχει πάντα ο κίνδυνος εάν δεν συμμετέχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη διαδικασία ε, ε, τυποποίησης ε, να αποσυρθούν προϊόντα τους από την αγορά. και έτσι να παρεμποδίζεται η καινοτομία. Τελειώνοντας, η παρουσία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να ε, ενδυναμωθεί πάνω απ' όλα σε εθνικό επίπεδο, εκεί όπου δεν υπάρχουν προβλήματα, γλωσσικά κιόλας αν θέλετε που δεν χρειάζεται για παράδειγμα μετάφραση, διερμηνία όπως εδώ. Το κόστος είναι πολύ ε, λιγότερο από ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο. Όσον τώρα, όταν πάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειάζονται αυτές οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρηματική υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχει ένας αντιπρόσωπος αυτών των επιχειρήσεων και επίσης να είναι αντικειμενικός αυτός ο εκπρόσωπος και να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα όλων και όχι μόνο κάποιων. Επίσης πρέπει να φροντίσουμε για το κόστος. Το κόστος να είναι εφικτό έτσι ώστε οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να μην αποκλείονται από τη διαδικασία τυποποίησης. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μας παρουσιάσατε και την πρακτική σας πείρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σήμερα γιατί βλέπουμε ότι η τυποποίηση μπορεί να είναι και ένα θέμα χρόνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την ε, συνεισφορά σας. Νομίζω και εσείς και ο κ. Λεπάρκο συμφωνείτε πάρα πολύ για την ε, συμμετοχή των εθνικών φορέων. Έχουμε λοιπόν τώρα περίπου μισή ώρα για να ακούσουμε ερωτήσεις από τα μέλη και απαντήσεις ε, ελπίζουμε από τους εμπειρογνώμονες. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει ο καθένας να λάβει άμεση απάντηση στην συγκεκριμένη του ερώτηση, αλλά αν μπορούσε ο καθένας την ερώτηση του να αναφέρει σε ποιον απευθύνεται θα ήταν το καλύτερο. Τώρα να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γκρόβιτσμαν, μετά η κυρία Γκέπχαρντ, η κυρία Ρούιλε, η κυρία Σαλτεμόζο, ο κύριο Σβάμπ, όλοι φαίνεται να θέλουν το λόγο και κυρία Κόμη, φαντάζομαι, ως εισηγήτρια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Εάν μπορείτε να είστε σύντομοι συνάδελφοι, πιο εύκολα θα απαντηθούν. Thank you, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ομιλητές για τις εξαίρετες παρουσιάσεις τους. Έχοντας ακούσει αυτά που είπαν, που είπανε και, έχω, και έχοντας δει και την πρόταση της Κομισιόν και τι τροπολογίες της ΕΝ και της ΕΝΕΛΕΚ, εγώ βλέπω να υπάρχουν αντιμαχόμενες προσεγγίσεις μεταξύ του Συμβουλίου και των φορέων τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. τυποποίηση στην Ευρώπη θα πρέπει να έχει διάφανο, συνεκτικό χαρακτήρα και φυσικά απαιτεί μια συνένεση μεταξύ των κυριωτέρων εμπλεκομένων, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, των κοινωνικών ομάδων, ιδίω των πιο ασθενών ομάδων, των οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος κτλ. Ζητούμε να υπάρξει από την Κομισιόν πλήρη συνεργασία με του φορεί τυποποίηση και με του άλλου κύριου εμπλεκομένου για να μπορέσουν να παροτρύνουν μια διαδικασία τυποποίηση στην Ευρώπη που θα είναι σωστά συντονισμένη και διαρθρωμένη για να μπορέσει να βοηθήσει τον Ευρωπαίο πολίτη σε μια ανταγωνιστική Ευρώπη. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να αντανακλάται και στο κείμενο του προτινόμενου κανονισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα που ακριβώ ήταν το ερώτημά σα. Ο κύριο Κρόιτσμαν ακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ. Έχω να ρωτήσω κάτι όσον αφορά τον χρόνο της αλλαγής των ε, προτύπων. Δεν πρέπει να είναι πολύ λίγος αυτός ο χρόνος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κόστος ε, που αυτό θα έχει για τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Από την άλλη, οι τεχνικές ε, η τεχνική πρόοδος και οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας καθιστούν σημαντική την ανάπτυξη των προτύπων και εάν μια αλλαγή στα πρότυπα έχει πλεονεκτήματα, τότε φυσικά είναι λογικό να το επιταχύνουμε. Καταλαβαίνω βέβαια και το, αυτό, και το, τις επιπτώσεις που έχει αυτό στο κόστος για τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Και φυσικά είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Ο χρόνος για τις αλλαγές στα πρότυπα. Schneller Μάλιστα. Καταρχάς, ευχαριστώ όλους. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σε ένα σημείο θα εστιάσω. Μιλάμε για ταχύτητα. Και βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε η ΣΕΣΕΚ, γιατί και από τη δική μου εμπειρία είναι, εξαρτά, εξαρτώνται όλα από τις εντολές της ε, Κομισιόν από το, γενικότερα από το τι θα κάνει η Κομισιόν. Όσον, ε, για παράδειγμα, η οδηγία για τα παιχνίδια. Από την οδηγία αυτή ε, γνωρίζω ότι η Κομισιόν χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να δώσει αυτή την εντολή. Και φυσικά δεν έχει κανένα νόημα όταν εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ασκούμε κριτική και λέμε ότι τα πρότυπα ε, αναπτύσσονται πολύ αργά όταν η Κομισιόν θέλει τέσσερα χρόνια για να φτάσει από το σημείο Α στο σημείο Β επιπλέον. Φυσικά ακούγεται ωραίο ε, το ότι σε εθνικό επίπεδο όλοι πρέπει να εμπλέκονται. Πρέπει όμως να έχουμε και να λαμβάνουμε τις πληροφορίες για την συμμετοχή ε, στο εθνικό επίπεδο των ενδιαφερομένων. Από την άλλη άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτά που είπε ο αντιπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης. Και βλέπω και θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ασχοληθεί ώστε η ανάμειξη σε εθνικό επίπεδο να γίνει πολύ ε, μεγαλύτερη. Κυρίως από τους ε, ενδιαφερομένους και πιστεύω πως ε, πρέπει να ε, φροντίσουμε το σχέδιο που θα συντάξουμε να ε, αναφέρεται και να απευθύνεται στους ενδιαφερομένους. σε ευχαριστώ πολύ. Θα το σημειώσουμε. Επόμενος, κυρία Κέπχαρτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι φανερό ότι η οι Γερμανοί ευρωβουλευτέ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά, αλλά φυσικά το θέμα τη τυποποίηση για τα τροφιμικά προϊόντα έχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στο Γάλλο εκπρόσωπο τυποποίηση. Μου φάνηκε πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία είπε μέχρι, μέχρι να φτάσει όμως στο τέλος της ε, παρουσίασής του. Αναφέρε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τις ε, ε, επιχειρήσεις να συμμετέχουν και να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις. Αυτό μου φαίνεται κάπως παράξενο. Εγώ νομίζω ότι ίσως δεν υπάρχει αρκετή υπευθυνοποίηση των επιχειρήσεων. Θα ήθελα να μου επαναλάβει αυτή την ε, επιχειρηματολογία που παρουσίασε γιατί μου φάνηκε κάπως παράξενη. Θα ήθελα όμως να θέσω το εξή ερώτημα, ένα διαφορετικό ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο με απασχολεί εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα. Όταν μιλάμε για τυποποίηση για τα τροφιμικά προϊόντα, μιλάμε πάρα πολύ για τα προϊόντα τα ίδια και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Αναφέρθηκε το θέμα των ε, βακτηρίων, των άλλων προβλημάτων που μπορούν να είναι παρόντα και αυτό σίγουρα η τυποποίηση στον τομέα αυτό βοηθάει τι επιχειρήσει, βοηθάει τον καταναλωτή, οδηγεί σε εξοικονόμηση κόστου και για τον καταναλωτή και επομένω έχει μεγάλη σημασία και προφανώ επέχει και ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά συζητάτε όλο και περισσότερο το θέμα της παροχής υπηρεσιών. Και υπήρξαν οι προτάσεις ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία τυποποίησης και για την παροχή υπηρεσιών. Εδώ έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε κανείς να τυποποιήσει την παροχή υπηρεσιών, γιατί η παροχή υπηρεσιών είναι προς την κατεύθυνση των ανθρώπων, των καταναλωτών και αυτοί οι οποίοι ζητούν την παροχή υπηρεσιών έχουν εξατομικευμένες ανάγκες. Πώς θα μπορέσει λοιπόν να τυποποιηθεί η παροχή υπηρεσιών. Θα ήθελα να θέσω λοιπόν το ερώτημα αυτό. Αυτοί που είναι οι υπέρμαχοι της τυποποίησης για τις υπηρεσίες, πώς θα μπορέσουν να με πείσουν ότι είναι απαραίτητη τυποποίηση, γιατί ακόμα κρατάω μια ιδιαίτερη σκεπτικιστική στάση απέναντι στην τυποποίηση των υπηρεσιών. Δεν καταλαβαίνω ποιο νόημα θα είχε. Ωραία. Ο κύριος Γκαρσία Ντίας θα επανέλθει στα έξι σημεία του για τα θέματα. Η κυρία Σάλντε Μόζε έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκομένους για τις πολύ καλές τους παρουσιάσεις σήμερα. Ίσως θα ήθελα να θέσω τρία ερωτήματα, θα είμαι σύντομη όμως. Μιλάμε καταρχήν για το θέμα της ταχύτητας στη διαδικασία τυποποίησης. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ανάγκη να επιταχύνουμε τις διεργασίες αυτές. Μήπως όμως αυτά εξαρτώνται από το είδος των προτύπων για τα οποία αναφερόμαστε. Αυτό το πρώτο μου ερώτημα. Όταν μιλάμε για τεχνολογίε πληροφορία και επικοινωνία, καταλαβαίνω θα πρέπει να επιταχύνουμε στο βαθμό του δυνατού την τυποποίηση. Για τα κατασκευαστικά υλικά όμω ίσω χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την τυποποίηση. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξή. Θα ήθελα να ακούσω και σχόλια των άλλων ομιλητών για αυτά που είπε ο Στεφαν Μπόι για την τροποποίηση του παρατήματος 3 να περιλάβει έτσι και τους εργαζομένους και τις αρχές εποπτείας των αγορών. Μου φαίνεται εμένα ότι είναι μια καλή ιδέα, θα ήθελα να ξέρω όμως την άψη των άλλων εμπλεκομένων. Και τρίτον, θα ήθελα να θίξω το εξής ερώτημα του εκπροσώπου της ΑΝΕΚ για τα δικαιώματα ψηφοφορίας των εμπλεκομένων από την κοινωνία των πολιτών, των διαφόρων φορέων, καταναλωτών, ενώσεων κτλ. Θα ήθελα και εδώ να ακούσω την άποψη των υπολείπων για τη δυνατότητα αυτή να έχουν δικαιώματα ψήφου. Ο κύριος Σουάμπ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρουσε τις παρουσιάσεις των ομιλητών. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές και την εισηγητριά μας για τη διοργάνωση αυτή. Ελέγχθηκαν πάρα πολλά ήδη και γι' αυτό θα είμαι σύντομος. Όλοι νομίζω ότι συμφωνούμε ότι μέχρι στιγμής η διαδικασία τυποποίηση βασίστηκε πάρα πολύ στην εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων και δεν υπάρχει νομοθετική, ναι, νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κατά την άποψή μου θα έπρεπε να την καλύψει. Φυσικά είναι διαφορετική η μορφή της τυποποίησης από τη μορφή της νομοθεσίας. Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα της νομοθεσίας με την τυποποίηση γιατί υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις στα θέματα αυτά. Θα ήθελα εδώ να θέσω το ερώτημα μήπως θα πρέπει να υπάρχουν και πολύ περισσότεροι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία γιατί έχουν ενδιαφέρον και ευθύνη. Σε ορισμένου τομεί όπω η τηλεφωνία, παραδείγματο χάρη, χρειάστηκε να ασκηθεί πίεση στη βιομηχανία για να προβούν σε σε τυποποίηση. Σε άλλες περιπτώσει όμω υπάρχει κίνδυνο να είναι υπερβολικά ευρεία η συμμετοχή των ενδιαφερομένων και όπως είπε και η κυρία Γκέπχαρτ και εγώ έχω κάποιες, ε, κάποιες αμφιβολίες για το αν είναι δυνατόν να υπάρχει πλήρης τυποποίηση των υπηρεσιών διότι αναφέρονται σε εξατομικευμένους καταναλωτές. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένε υπηρεσίες οι οποίες θα ήταν χρήσιμο να έχουν μια τυποποίηση. Επίσης αναφέρατε ότι η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό είναι πραγματικά το πιο σημαντικό, γιατί αυτοί είναι, αυτοί, αυτές είναι επιχειρήσεις που είναι πιο κοντά στον εργαζόμενο και στον καταναλωτή και γι' αυτό είναι απαραίτητη και νευραλική η ταχύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εσείς τονίσατε ότι είναι πιο σημαντικό όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμμετέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν θέσω το ερώτημα αυτό το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια να μειώνεται αισθητά η συμμετοχή τους στις διαδικασίες αυτές. Έχουμε κάποιους εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα απαντήσουν για τα θέματα των ε, ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τέλος η συγγητριά μας. Εγώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ε, παρουσίαση του, Ιταλ, του Γάλλου Υπουργού, διότι κατά κάποιο τρόπο βλέπω να κινείται αντίθετα στο ρεύμα των θέσεων των υπολείπων. Και εγώ θα ήθελα να αναφέρω μερικές από τις δικές μου σκέψεις. Και εγώ έρχομαι από την Ιταλία, όπου είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει μια έλλειψη σύνδεση μεταξύ του εθνικού επίπεδου και του ευρωπαϊκού επίπεδου. Αλλά ακόμα και μέσα σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει απόλυτη ενότητα μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και στη Γαλλία είναι πολύ διαφορετικές οι μικρομεσαίες μεταξύ τους. Πώς συνεργάστηκαν όμως τελικώς, ε, πώς εσείς βελτιστοποιήσατε την εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οργανώθηκαν σε επιτροπές, σε κονσόρσια ή σε άτυπες ανεξάρτητες ομάδες. Και οι ομάδες αυτές εφόσον ήταν ε, σαν ε, κονσόρσια συγκεντρώθηκαν ανατομέα ή ανα επιχειρησιακό κλάδο. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα χρόνου ούτως ή άλλως και Εάν έπρεπε να εφαρμόσουμε κάτι ανάλογο στην Ιταλία, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήδη με το βάτσερ τη κοινοτομία για να διοργανωθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, έχουμε πολύ ε, μικρή ανταπόκριση ακόμη. Μπράβο λοιπόν στου Γάλλου ε, για τη δωρεάν διαδικασία που προέβλεψαν. Πρόεδρο, πολλέ ερωτήσει. Να ξεκινήσουμε αντίστροφα. Νομίζω η κυρία Σαντιάγκο πρώτη θα έπρεπε να λάβει το λόγο για το θέμα της ταχύτητας και τη όλης διαδικασίες ε, θα πρέπει τρεις πρώτοι ομιλητές μας να παρέμβουν. Ο κύριος Γκαρσία Ντίας για το θέμα των υπηρεσιών, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο κύριος Λεπάρκο και ο κύριος Τόστεν και ο κύριος Στούρμαν. Νομίζω και για την πρόταση του κύριου Μπόη τέθηκε ένα ερώτημα. που φαντάζομαι ότι και η κυρία Σαντιάκο και οι υπόλοιποι μπορεί να θέλουν να σχολιάσουν. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Εάν υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να συμβάλλουν, παρακαλώ. Ο κύριος Εάν μπορείτε σε ένα λεπτό καθένας, θα ήταν τέλεια. Θα σας βάλουμε και χρονόμετρο, για να μην χάσετε το μέτρημα. Κυρία Σαντιάγκο, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα να απαντήσω στο θέμα της διατήρησης των ευρωπαϊκών ε, προτύπων. Όντως, η διαδικασία υπάρχει κανένα πενταετία, αναθεωρούμε τα πρότυπά μα. Υπάρχει τεχνική επιτροπή που αποφασίζει αν πρέπει να αναθεωρηθεί ένα πρότυπο ή όχι. Για να βοηθήσουμε λοιπόν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να γνωρίζουν τι ακριβώ συμβαίνει, το σημαντικότερο είναι να τι εμπλέξουμε στην όλη διαδικασία σχεδιασμού των προτύπων και στι εθνικέ τεχνικέ επιτροπέ. Πραγματικά υπάρχει απόφαση πρωτού αναθεωρηθεί ένα πρότυπο ή όχι. Επίση, για το θέμα τη ταχύτητα την ερώτηση τη κυρία Ρούλε. Κάποιες φορές χρειάζεται πολύς χρόνο για να προετοιμαστεί μια εντολή. Υπάρχουν ανάλογε προτάσει για, ε, για πλατφόρμε πλατφόρμες και ΣΕΝΙΣ ΣΕΝΕΛΕΚ έχουν ε, ταχθεί υπέρ μια τέτοια πλατφόρμα όπου να συμμετέχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Αυτό είναι το καλύτερο για να γνωρίζει κανεί τι συμβαίνει με το διά, διάβλο ε, προώθηση των σχεδίων ε, για, τον, για τα πρότυπα και να υπάρχει πλήρη ενημέρωση. Τώρα, η διαδικασία του ευρωπαϊκού Πεπέδου είναι ότι καλύπτουμε όσο περισσότερε ανάγκε. Και όσο περισσότερο πληθυσμό καλύπτει κάποιο, τόσο περισσότερη ε, βαρύτητα έχει η ψήφο ε, ανάλογα με την εκπροσώπηση στην Επιτροπή των Προτύπων. Εάν δώσουμε δίκαιο ένα χώρο, ασχέτω του πληθυσμού, θα αλλάζει αυτό ανάλογα με του τομεί τι ακριβώ προτείνεται. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε πραγματικά ε, βαρύτητα στην όλη διαδικασία και να βαραίνει η άποψή μα. Κάτι που δεν ανέφερε ίσω στην ε, παρουσίασή μου αρκετά ήταν η κατάρτιση. Κατάρτιση και ξανά κατάρτιση και άλλη κατάρτιση. Αυτό είναι ότι σημαντικότερο και από την άποψη της συντήρησης, της ε, ενημέρωσης, της ε, συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να γνωρίζει κανείς ποια είναι τα ωφέλη του συστήματος και για τις επιχειρησιακές επενδύσεις, για να συμμετάσχουν δηλαδή οι επιχειρήσεις στη δικασία των προτύπων. Τώρα, οι εμπορικέ οργανώσει έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν και για την ευρωπαϊκή την εθνική διαδικασία δημιουργία των προτύπων, κυρία Κόμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Κόμπερκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ταχύτητα. Οι νέε τεχνολογίε έρχονται και παρέρχονται, βεβαίω. Τα ωφέλη των νέων τεχνολογιών και η ταχεία εισαγωγή προτύπων θα πρέπει να εξισορροπεί την το μειονέκτημα του κατά πόσο γρήγορα αποσύρονται και τα απομεινάρια του παρελθόντος. Ε, κυρία Σαλντεμόζε, λοιπόν, αυτό όντω πρέπει να οργανωθεί ένα τομέα. Τώρα για την εκπροσώπηση, γιατί έγιναν κάποιε παρατηρήσει σχετικά. Ποια είναι η κατάλληλη εκπροσώπηση. Αυτό εξαρτάται και από τα συγκεκριμένα αγορά κάθε φορά και από το για ποιο πρότυπο μιλάμε. Οι ενδιαφερόμενοι από αυτό καθορίζονται. Επίσης, οι επίσημοι κανόνε εκπροσώπηση δεν θα καλύψουν τι ανάγκε τη πραγματικότητα. Αυτό που πραγματικά ε, έχει σημασία είναι να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, δηλαδή συμμετοχή. Και θα επαναλάβω κάτι που είπε ο κύριο Σφαμπ. Πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο χρήσιμο είναι να προσκαλούνται όλοι γύρω από ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, όπου δεν υπάρχει πραγματικά η δυνατότητα, η εντολή για να εκπροσωπήσουν κάποιους. Πρέπει αυτή η κατάσταση λοιπόν να ληφθεί υπόψη. Έπειτα, για το κατά πόσον κάποια δικαιώματα των φορέων του παρατήματος 3 πρέπει να διευρυνθούν ή κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι φορείς στο παρατήμα 3. Ναι, το σημερινό σύστημα πιστεύουμε πρέπει να παραμείνει ως έχει όχι να μην βαρύνει περισσότερο με δικαιώματα ψήφου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα για τι υπηρεσίε. Είπαμε ότι πρέπει οι στόχοι μα να καθοριστούν βάσει των αναγκών τη αγορά. Συμφωνώ λοιπόν απολύτω με μια καθοριστική παρατήρηση που έγινε γι' αυτό. Και πρέπει να πω πρώτα να σκεφτόμαστε εάν λειτουργήσε για τα προϊόντα η ενιαία αγορά και αν μπορούμε να την ε, μεταφέρουμε αυτούσια την ίδια ιδέα και στις υπηρεσίες. Δεν θα λειτουργήσει απαραίτητα έτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα σημαντικό σημείο για τα πρότυπα είναι ότι στόχος μας εδώ δεν είναι να περιορίσουμε την ανταγωνιστικότητα, είναι να την τονώσουμε. Θέλουμε νέα προϊόντα να φτάσουν στην αγορά και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Άρα αυτή τη θεμελιώδη ιδέα πρέπει να την έχουμε κατά νου όταν μιλάμε για πρότυπα. Δεύτερο σημείο. Πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ του ρυθμιστικού πλαισίου και της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των ρυθμίσεων με κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες που αναφέρθηκαν την EMC, εδώ μιλάμε για πρότυπα που έχουν σχέση με την μέτρηση. Πρέπει να γίνονται απαραίτητε μετρήσει για να βεβαιώνεται κανεί ότι ένα προϊόν βρίσκεται εντό των κριτηρίων που ορίζει ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Για να δούμε αν ένα προϊόν είναι ασφαλέ για του χρήστε, για να μην ε, δημιουργήσει οκλήσει για του υπόλοιπου καταναλωτέ. Αυτά δημιουργούνται αργά και με τρόπο ομαλό από ένα χρονικό σημείο σε ένα άλλο. Κάποια στοιχεία ενίοτε αλλάζουν, αλλά δεν είναι ταχύε εξελίξει. Είναι σταθερά περίπου αυτά τα κριτήρια. Στον τομέα όμω τη ανταγωνιστικότητα έχουμε ραγδαίε εξελίξει. Και εδώ πρέπει βεβαίω να διατηρήσουμε το ρυθμό. Πρέπει οι εξελίξει να λαμβάνονται υπόψη και τα πρότυπα που σχεδιάζονται να επιτρέπουν στου χρήστε και του καταναλωτέ να τα χρησιμοποιούν. Ένα Παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, λόγου χάρη. Έχουμε τα smartphones πλέον, τα οποία είναι πολύ πιο περίπλοκα, έχουν πολλές ε, λειτουργίες από ότι τα αρχικά κινητά τηλέφωνα, τα λεγόμενα GSM. Όμως και αυτά λειτουργούν μια χαρά ακόμη. Κάποιοι τα χρησιμοποιούν κιόλα. Σημαντική λοιπόν ε, διαφορά στην εξέλιξη του σχετικού προτύπου θα είναι η διαλογικότητα στον τομέα των ICT, όπου καλύπτουμε και επηρεάζουμε κάθε τομέα δραστηριότητα, οποιονδήποτε και να σκεφτούμε, όλοι οι υπόλοιποι στηρίζονται σε αυτόν. Εδώ πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε συνεπεί. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία μεταξύ όλων των τομέων μεταξύ του. Άρα, στο πλαίσιο αυτό και όταν σχεδιάζουμε νέα πρότυπα ή αναθεωρούμε κάποιο υπάρχον, πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει συμβατότητα με την προηγούμενη εκδοχή. Παρακαλώ, δεν έχουμε τόσο χρόνο. Συντομεύστε αν μπορείτε. Δύο προτάσεις. Πρώτον, θα πρέπει οι διάφορε οργανώσει, και τα διάφορα πρότυπά του να λαμβάνουν υπόψη τι προδιαγραφέ των κονσόρσια και επίση πολύ γρήγορα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αν επιτρέπετε, στην ψηφιακή, την Digital Europe μάλλον. Έχουμε ε, κατασκευαστές ε, τηλεπικοινωνιών, ε, ICT, ηλεκτρικών συσκευών και ούτω καθεξής. Όμως, ως πλήρη μέλη, συμμετέχουν και ενώσεις εθνικών μηχάνων ICT. Αυτό έχει αποδώσει πολύ καλά αποτελέσματα ως τώρα. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις μεγάλες εταιρείες και να τις βάλουμε σε αντίπαλα στρατόπεδα. Θα πρέπει όλοι να συνεργάζονται να συμπλέουν και να υπάρχει και ε, στήριξη του ενός προς τον άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Γκαρσία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, για την τυποποίηση στις υπηρεσίες. Πολύ εύστοχο το ερώτημα. Διότι το έχουν θέσει οι ίδιοι οι βιομηχανικοί κλάδοι όταν ανακύπτει το ερώτημα αυτό. Όπως το προανέφερα στην παρουσίαση. Πρέπει να υπάρχει συμβατότητα και με την ποιότητα των υπηρεσιών και με τον θεμητό ανταγωνισμό και το καθεξή. Θα επικεντρωθώ λοιπόν στο εξή, το πώ γίνονται όλα αυτά μετά από όλη αυτή τη συζήτηση. Πώ να τυποποιηθεί κάτι που τόσο πολύ επικεντρώνεται, η αξία του μάλλον επικεντρώνεται στο πώ το βλέπει ο πελάτη. Δηλαδή πώ κάνει την διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων προμηθευτών είναι σαφές εδώ. Το καταλαβαίνουμε και η πείρα μας ε, από κάποιες από τις περιπτώσεις που είχα αναφέρει μας έχει οδηγήσει στο εξής. Επικεντρωνόμαστε στον κύκλο ζωής μιας υπηρεσίας. Επικεντρωνόμαστε σε οριζόντια θέματα, όπως η ικανοποίηση των πελατών, ε, η τιμή, οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται. Αυτό κάποιες φορές αφορά διατομεακά ζητήματα, όπως ο σχεδιασμός της υπηρεσίας, το μάρκετινγκ της υπηρεσίας, οι ε, αποκρίσεις των ε, πελατών στην περίπτωση των υπηρεσιών μετάφρασης λόγω χάρη, όπως είχα αναφέρει και νωρίτερα. Πρέπει να υπάρξει μια αρχική μετάφραση από έναν επαγγελματία, μετά διόρθωση από κάποιον άλλον επιμέλεια δηλαδή. Μετά πρέπει να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση προηγουμένω, κάποια συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα. Όλα αυτά αφορούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Έτσι καλύπτουμε τι υπηρεσίε με ένα πρότυπο. Τώρα, ένα άλλο παράδειγμα, το facility management. Τι θα τυποποιήσουμε εδώ. Το συμβασιακό περιεχόμενο ενδεχόμενο μεταξύ του παρέχοντο στην υπηρεσία και του πελάτου. Τώρα, ο ορισμό των υπηρεσιών που παρέχονται αυτομάτω. Δεν υπάρχει κοινή συνεννόηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τι υπηρεσίε. Δεν εννοούμε όλοι τα ίδια πράγματα από τη μια χώρα στην άλλη. Άρα προσπαθούμε να έχουμε ένα βασικό έγγραφο στον φορέα μα για να μπορέσουν και οι προμηθευτέ και οι καταναλωτέ να καταλάβουν πώ μπορεί να ωφεληθούν από τη δημιουργία προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτό που σε κάθε περίπτωση επιζητούμε με το έγγραφο αυτό και με το σχέδιο του κανονισμού είναι ότι θα μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον τομέα των υπηρεσιών για το δυναμικό που παρουσιάζει η δυνατότητα των προτύπων να ενισχυθεί ανταγωνιστικότητα και να βασιστούμε σε επιτυχημένα παραδείγματα. Ευχαριστούμε κύριε Χάρης.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 θα σχολιάσω αυτά που υπόθηκαν, αλλά δεν θέλω να επαναλάβω τα λόγια μου. Δύο πολύ γρήγορα σχόλια. Ναι, οι αλλαγέ στα πρότυπα καθορίζονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά τώρα ολόνα και περισσότερες αλλαγέ ε, που επηρεάζουν τις μισέ εταιρείε προκύπτουν από την ομοθεσία. Αρκετές εταιρείε έχουν παραπονεθεί σε εμά λέγοντα ότι η μισή του δουλειά είναι να εφαρμόζουν τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από την νομοθεσία. Έπειτα, τα πρότυπα των υπηρεσιών. Εξαρτάται από τον τομέα. Ορισμένοι τομείς χρησιμοποιούν υπηρεσίες επιπροσθέτως και ορισμένες αυξάνονται και εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα. Για εμάς αυτό που είναι σημαντικό είναι τα πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών να είναι χρήσιμα και δεν υπάρχει γι' αυτό δικαιολογία για να εισάγονται, εισάγονται καινούργια και πιο περίπλοκα πρότυπα. Θα ήθελα να σχολιάσω και να πω δύο λόγια τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις πριν προχωρήσω. Κύριε Λεπάρκο, εσείς είχατε κάποια σχόλια, Κύριε Στόρστεν επίσης. Κύριος Λεπάρκο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρωτού απαντήσω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να απαντήσω στην κυρία Ρούλα, Ρούλε μάλλον που μου έθεσε το θέμα των άλλων συμμετεχόντων πλέον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Προφανώ δεν μίλησα για το θέμα αυτό, γιατί μου ζητήσαν να μιλήσω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει μόναχα σε αυτή τη συνεδρίαση. Αλλά όλο αυτό ο μηχανισμό που ανέφερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει υπάρχει και για του καταναλωτέ, για τα συνδικάτα, για του εκπροσώπου των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Δηλαδή ότι είναι δωρεάν η συμμετοχή του, ότι υπάρχει μια υποστήριξη σε αυτού και υπάρχει και μια συμβουλευτική επιτροπή που του περιλαμβάνει. Όπω είπα εγώ στην αρχή, περιλαμβάνω όλε αυτέ τι ομάδε οι οποίε θα πρέπει να έχουν την ίδια δυνατότητα συμμετοχή και θα πρέπει να έχουμε την ίδια δυνατότητα παρότρινση όλων αυτών των φορέων από τη δική μα πλευρά. Για τα consortium τώρα που αναφέρθηκε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμεί δεν ενθαρρύνουμε τη δημιουργία τέτοιων consortium. Ζητούμε να ομαδοποιηθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αλλά για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε διαδικασίε που ήδη υφίστανται. Θέλουμε να αποφύγουμε παράλληλες διαδικασίες τυποποίησης. Θέλουμε όλες οι μικρομεσαίες να συμμετέχουν στις υπάρχουσες διαδικασίες που νομίζουμε ότι σέβονται πλήρως το γενικό συμφέρον. Αυτό μας ενδιαφέρει με τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ευρωπαϊκού χαρακτήρα τυποποίησης να, να σέβονται και να προωθούν το, το κοινό συμφέρον. Και αυτή την οδό ακολουθούμε. Και για να απαντήσω στα άλλα ερωτήματα για τα δικαιώματα ψήφου δεν είπα ότι είμαι κατά του δικαιώματο ψήφου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αντίθετο, θέλω να μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει εκεί που μπορούν να ψηφίζουν, δηλαδή στι εθνικέ ομάδε τυποποίηση, όπου γίνεται ουσιαστικά μια, ένα συγκερασμό των θέσεων για να υπάρξει μια γενική θέση. Αυτό το οποίο είναι διαφορετικό είναι το να έχουν δικαίωμα ψήφου σε παράλληλες ομάδε, παράλληλα με του σχηματισμού που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να έρθει κάποιο να δώσει την άποψή του. Φυσικά θα εκπροσωπήσει μια θέση, αλλά πώς ξέρουμε ότι με την ψηφοφορία του σε εθνικό επίπεδο θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει όλε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που δουλεύουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το επιτύχει κανεί. Χρειάζεται να γίνουν προσπάθειε. Εγώ υποστηρίζω αυτού που κάνουν την προσπάθεια αυτή, αλλά είναι ένα εγχείρημα πραγματικά μεγάλη δυσκολία. Θα πρέπει να ξαναφτιάξουμε από την αρχή συστήματα όπως αυτά που είχαμε στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. Γι' αυτό εγώ προτιμώ να δώσουμε τη δυνατότητα σε εθνικό επίπεδο να συμμετέχουν και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενσωματώνονται στο γενικό πλαίσιο και όχι να δημιουργηθούν παράλληλες δομές για το ψηφοφορία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εγώ θα ήθελα. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω στις ερωτήσεις της κυρίας Γκέμπχαρτ και του κυρίου Σφάμπ. Πώς να αναμίξουμε τους ενδιαφερόμενους, τους επλεκόμενους στην διαδικασία τυποποίησης. Συμφωνώ πως η απάντηση είναι απλή και μία απάντηση θα μπορούσε να είναι να κάνουμε τα πρότυπα ελκυστικά, να τα κάνουμε σεξι, έτσι ώστε όλοι να θέλουν να αναμειχθούν, γιατί ξέρουμε όλοι ότι όταν, αν φτιάξεις τα πρότυπα, φτιάχνεις και την αγορά σου. Έπειτα, πληροφορία και εκπαίδευση. Κατανοώ ότι σε όλα τα κράτη-μέλη ότι δεν έχουμε σε όλα τα κράτη-μέλη την κατάλληλη εκπαίδευση. Για παράδειγμα, οι μηχανικοί ε, δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση στον τομέα της, ε, της ετυποποίησης. Μέρος της δουλειάς μας είναι να το φροντίσουμε αυτό και να το κάνουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Επιπλέον, ε, θα σας δείξω αυτήν την εικόνα. Αυτή η εικόνα που έγινε ίσως από τον Κυριακόμη, από τον Πρόεδρο, μας δείχνει πώς λειτουργεί η τυποποίηση. Τι είναι η τυποποίηση και επίσης μας δείχνει πώς λειτουργούν ε, οι υπηρεσίες. Και θα ήθελα να σας ε, επιστήσω την προσοχή στην μικρή εικόνα ε, στα αριστερά, στους κομωτές. Στο παράδειγμα αυτό, αν δείτε αυτό το παράδειγμα, θα, αναρωτη... θα αναρωτηθείτε πραγματικά χρειαζόμαστε όντως τα πρότυπα στις υπηρεσίες. Ε, νομίζω πως αυτή η εικόνα προήλθε από την έκθεση της Enelex και, μας, ε, και η Σάνελεξ μας έδωσε άδεια να τη χρησιμοποιήσουμε. Μας τελειώνει ο χρόνος. Θέλει, ήθελε κάποιος άλλος να σχολιάσει. Ο κύριος Τόρστεν μας έδειξε ήδη πώς να κάνουμε τα πρότυπα σεξι και ας το κρατήσουμε αυτό για τη σημερινή μέρα. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσω στο τελευταίο μέρος της ε, συνεδρίασής μας. Έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Ρόμπερτ Στήλ ανάμεσά μας Γενικό Γραμματέα του ΆΙΖΟ. Έχουμε, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Είμαστε ευγνώμονες να σας ακούσουμε. Επίσης την κυρία Έιμι Μαράσκο, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμερικανικού Ινστιτούτου Εθνικών Προτύπων και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ την εβδομάδα των ευχαριστειών που για σας είναι εθνική γιορτή. Δυστυχώ όμω εμεί έπρεπε να οργανώσουμε την ε, συνεδρίαση τώρα, αλλιώ θα έπρεπε να περιμένουμε μετά τα Χριστούγεννα. Τέλο, ε, χαίρομαι που καλωσορίζω τον κύριο Φεν Τσουνκουάν από την ε, Κινέζικη Αντιπροσωπεία και τον David Τόσετ ο οποίος είναι πρόεδρος της Σένελεκ και τον κύριο Βάιλερ, πρόεδρο της ΕΤΣΙ και μόλις τώρα κατέφθασε ο κύριος Βίλκινσον από την JRC. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς καθυστέρηση ας προχωρήσουμε και αν έχουμε χρόνο ίσως καταφέρουμε να απαντήσουμε και σε μερικές ερωτήσεις. Τώρα όμως κύριε Στυλ έχετε το λόγο για 10 λεπτά μάξιμου. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Εκτιμώ την ευκαιρία που μου δώσατε για να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Ο τίτλος της ε, παρουσίασής μου είναι «Η τυποποίηση στο, παγκόσμιο περιβάλλον και τα στοιχεία που έχουμε». Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην ε, διαδικασία τυποποίησης, αν και οι προηγούμενοι ομιλητές ε, μίλησαν αρκετά, την αρχή της εθνικής αντιπροσώπευσης, επίσης θα ήθελα να τονίσω, και επίσης ένα γενικό, μια γενική συζήτηση για το τι δουλεύει καλά. Και θα ήθελα να πω ότι η Ευρώπη σε αυτό το τομέα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Εμείς δημιουργούμε πρότυπα και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της αγοράς και γι' αυτό χρειαζόμαστε βιώσιμα μοντέλα για να το καταφέρουμε. Τα μέλη της ISO είναι 163 ανά τον κόσμο Λειτουργούμε με την αρχή της ε, μίας ψήφου για κάθε χώρα και φυσικά η Ευρώπη έχει, δεν έχει μία ψήφο, έχει μία ψήφο για κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε πάνω από 200 τεχνικές επιτροπές και αν προσθέσετε και τις υποεπιτροπές έχουμε περίπου 3.300 τεχνικές ομάδες. Και σήμερα έχουμε περίπου 11 συνεδριάσεις σε όλο τον κόσμο. Κάτι που όλα τα μέλη της ISO και η ίδια η ISO είναι αναμεμειγμένα είναι το εξής. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσφατα δημοσίευσε μία έκθεση σχετικά με την συνένεση για τα πρότυπα ISO και για, για τις κατασκευές για την ε, ανάμειξη των ενδιαφερομένων στα νέα έργα, για την εθνική συμμετοχή, για την ανάπτυξη πρότυπων ISO, για την ανάπτυξη και οργάνωση επιτροπών, οι οποίες θα παρακολουθούν την διαδικασία ανάπτυξης και τέλος των εθνικών επιτροπών. Πιστεύω πως αυτά τα έγγραφα είναι ξεκάθαρα και ελπίζω να τα να δοθούν στην διάθεση του Κοινοβουλίου. All Μάλιστα. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε ενεργά αναμειγμένοι με δύο ομάδες που αναφέρθηκαν στο σχέδιο του κανονισμού, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Και οι δύο αυτές ομάδες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις εθνικές ε, αντιπροσωπείες των Επιτροπών και κάνουν καλή δουλειά. Είναι αποδοτικές. Πιστεύω πως πρέπει να ενισχύσουμε την, ε, τη συμμετοχή αυτή σε τοπικό επίπεδο. Επίσης η ΕΝΕΚ έχει συνδέσμους με αρκετές από τις επιτροπές ΆΙΖΟ. Συμμετέχει σε πολλές επιτροπές και υποεπιτροπές, για παράδειγμα για τον τουρισμό και τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Και σε περιβαλλοντική διαχείριση και οικονομική διαχείριση. Επίσης, έχουμε την ομάδα πολιτικής καταναλωτών που ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα των, των καταναλωτών. Η αντιμετώπιση της ΆΙΖΟ στις ε, παγκόσμιες αλλαγές είναι εξή. Όταν μιλάμε για πρότυπα, δεν μιλάμε μόνο για οικονομικά πρότυπα και βιομηχανικά και μηχανικά πρότυπα, αν και αυτά συμπεριλαμβάνονται. Μιλάμε όμω επίση και για βιωσιμότητα, για το περιβάλλον και για την κοινωνία. Θα δείτε πως έχουμε ένα ευρύ φάσμα νέων προτύπων, τα οποία δημιουργήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια και αυτό είναι μια ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να αναφέρω κάτι που υπόθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου περιγράφηκαν τα, οι έξι σημαντικότεροι ε, κίνδυνοι, η κλιματική αλλαγή, η, οικονομική, παγκόσμια διακυβέρνηση και η αποτυχία της. Κάποιες από αυτές ήταν, ήταν τεχνικές και οικονομικές, όμως όλες αφορούσαν τους ε, καταναλωτές και τις ομάδες ενδιαφερομένων και όλοι αυτοί εξαρτώνται και έχουν άμεση σχέση με τα πρότυπα. Σίγουρα κοιτάζοντας αυτή την ομάδα, ο ορισμός, η δυνατότητα να υπάρχει ένας διεθνής ορισμός είναι πολύ σημαντικό για την τυποποίηση. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη για τις ε, επερχόμενες αλλαγές, εμπιστοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο, εμπιστοσύνη σε εμπορικούς εταίρους, εδώ στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Κάτι που αναφέρθηκε πριν σε ερώτηση ήταν η αξία των προτύπων και η σχέση τους με αυτούς που πραγματικά συμμετέχουν στην ε, διαδικασία δημιουργίας τους και σε αυτούς που δεν συμμετέχουν. Μου φαίνεται πως εδώ έχουμε δύο, δύο επίπεδα. Τα μέλη της ΆΙΖΟ ε, και των άλλων οργανισμών τυποποίησης έχουν εργαστεί ήδη αρκετά και πιστεύω ότι υπάρχει, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αυτά που βλέπετε στον ε, πίνακα προέρχονται τρία από αυτά που βλέπετε στο πίνακα προέρχονται από τον ευρωπαϊκό χώρο. Σε επιχειρησιακό επίπεδο τώρα πιστεύω πως πρέπει να δείξουμε στις επιχειρήσεις και στις μεγάλες και στις μικρές τι ανάγκες υπάρχουν. Σίγουρα ένα από τα σημεία που πιστεύω πως πρέπει να τονιστούν είναι το τέταρτο στη διαφάνεια η μη συμμετοχή στη διαδικασία τυποποίησης δίνει προβάδισμα στον ανταγωνιστή. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν δεν σας ενδιαφέρει, μην πείτε στον κοπέ. Αν σας ενδιαφέρει όμως, ασχοληθείτε. Αν δεν σας ενδιαφέρει να παίξετε με τους κανόνες, τότε σας παρακαλώ να μην συμμετέχετε, με άλλα λόγια. Τώρα η αξία των προτύπων είναι πολύ σημαντική. Η Άιζο μόλις δημοσίευσε αυτό το έγγραφο που υπάρχουν 11 μελέτες που έγιναν από επιχειρήσεις ε, ανά τον κόσμο, δείχνουν αύξηση στις, προ... στις πωλήσει, βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά, καλύτερη σχέση με τους ε, καταναλωτές, ικανοποίηση των καταναλωτών και αυτό, όλα αυτά ως ε, αποτέλεσμα έχουν αύξηση των κερδών για τις μικρές επιχειρήσεις. Τώρα, η ανάμειξη της Ευρώπης με την ISO, 17% ε, των μελών της ΆΙΖΟ βρίσκονται στην Ευρώπη. Έχετε πολλές τεχνικές επιτροπές και συμβάλλονται σημαντικά στην διακυβέρνηση. Η ανάμειξή σας στην ΆΙΖΟ και η ενασχόλησή σας είναι τεράστια. Ένας τομέας είναι η Συμφωνία της Βιέννης, που τώρα μόλις έκλεισε τα 20 χρόνια. Και τα πλεονεκτήματα τα βλέπετε στην οθόνη σα τη συμφωνία σας αυτής. Και σίγουρα από την ε, προοπτική της ISO ε, είναι πολύ σημαντικό τα πρότυπα της ISO ε, να, υιοθε... να υιοθετούνται από την Ευρώπη και να λειτουργούν ως ευρωπαϊκά πρότυπα. Τέλος, σε αυτή τη διαφάνεια μπορείτε να δείτε ότι η Ευρώπη μέσω της ε, Συμφωνίας της Βιέννης έχει πολύ σημαντική ε, θέση στην διαδικασία δημιουργίας προτύπων στην Άιζο. Έπειτα όσον αφορά την αρχή της εθνικής αντιπροσώπευσης, τους ε, κανόνες για την ψηφοφορία στην Άιζο. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για την Άιζο. Τα μέλη μας τα μέλη μας και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως σας είπα, λειτουργούν με την αρχή της μίας χώρας σε μία ψήφος. Το επιχειρηματικό μοντέλο της ISO έχει ως εξής. Λειτουργούμε με βάση την αντικειμενικότητα, την διαφάνεια και την ανοιχτή πρόσβαση σε όλους. Πρέπει να βρισκόμαστε και να έχουμε παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο Χρειάζεται να είμαστε απλοί και να είμαστε γρήγοροι και σε αυτό θα επανέλθω. Και τέλος χρειάζεται να έχουμε σεβασμό στους ε, πόρους που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία δημιουργίας προτύπων. Αρκετοί από τους συνομιλητές μου έκαναν λόγο για, για πιο γρήγορη διαδικασία, για πιο απλή και για καλύτερη. Και συμφωνώ, πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι. Πρέπει να είμαστε πιο απλοί. Δεν πρέπει να χαλάμε τον χρόνο των άλλων. Χρειάζεται επίσης να μιλήσουμε και για τις συνθήκες, για παράδειγμα τα οικοδομικά υλικά. Σε περίπτωση ενός ε, μεγάλου σεισμού, τα οικοδομικά υλικά πρέπει να αλλάξουν και να, να αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα. Τα εργαλεία επικοινωνίας μας. Χρησιμοποιούμε για παράδειγμα το WebEx. Επίσης χρησιμοποιούμε τα ε, social media. Και το διαδίκτυο, πάρα πολύ το διαδίκτυο. Θα ήθελα να καλέσω τα μέλη μας, εάν έχετε υπνίες, να ρίξετε μια ματιά στο, στην, στον ιστότοπο της ΆΙΖΟ. Εκεί θα βρείτε πάρα πολλά, θα διαβάσετε πάρα πολύ για αυτό που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, είναι μεγάλη χαρά να είσαστε εδώ. Ξέρετε ότι έχουμε επισκεφθεί στο παρελθόν δύο φορές τον Άιζο και παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Η κυρία Μαράσκο τώρα από το Άνση έχει το λόγο για έξι λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Άννη Μαράσκο και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμερικανικού Ινστιτούτου Προτύπων, ANSI. Μιλάω εξ ονόματος της ANSI σήμερα και θέλω να σας ε, τονίσω ότι ο πρόεδρος μας χαίρεται πάρα πολύ για αυτή την ε, πρόσκληση για να δώσει την κατάθεσή του σε αυτή την ακρόαση και τον εκπροσώπω εγώ φυσικά. Για αυτούς από εσάς που δεν γνωρίζουν τι είμαστε, το ANSI είναι ένας ιδιωτικό μη κερδοσκοπικός φορέας ο οποίος διαχειρίζεται και συντονίζει τα εθελοντικά πρότυπα στι Ηνωμένες Είμαστε το εκπρόσωπο της Αμερικής, τη Ηνωμένων Πολιτείων στον Άιζο και μέσω της Εθνική μας επιτροπής το IEC. Εκπροσωπούμε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περιφερειακά φόρα. Σήμερα θέλω να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση της αμερικανικής προσέγγισης στη τυποποίηση. Το σύστημα μας θεωρείται ότι είναι ένα σύστημα εκ των κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πρότυπα είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν τη διαδικασία τυποποίησης. Εμείς βασιζόμαστε στη συμμετοχή και στη συνεργασία πολλών εμπλοκομένων, διαφόρων εμπλοκομένων από τον επιχειρηματικό τομέα, από, την κυβε... τις κυβερνήσεις, από τους καταναλωτές που έχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις. Πιστεύουμε ότι αυτή η πολυμορφία είναι αυτή που δίνει μεγαλύτερη ευρωστία στο σύστημά μας. Ένα ισχυρό και εύρωστο σύστημα προτύπων είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό για την επιτυχία σε παγκόσμια οικονομία. Πάνω από 100.000 πρότυπα έχουν αναπτυχθεί στην, στην Αμερικανική ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες από ενώσεις, επιτροπέ και κονσόρτσια. Πάνω από 10.000 από αυτά τα πρότυπα έχουν υποβληθεί στο Άνσι και έχουν εγκριθεί ως αμερικανικά εθνικά πρότυπα. Αυτό καταδεικνύει ότι τα έγγραφα αυτά ακολουθούν τις βασικές προαπαιτήσεις μας και έχουν αναπτυχθεί με μια ανοιχτή, ε, ισορροπημένη και βασιζόμενη σε συνένεση διαδικασία. Ποιοι συμμετέχουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία, στην εθελοντική αυτή διαμόρφωση των προτύπων. Είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε ο οποίο έχει υλικό συμφέρον σε αυτή τη διαδικασία. Περιλαμβάνει αυτό κυβερνητικού φορεί, επιχειρήσει, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταναλωτές, ε, εμπορικά επιμελητήρια και οργανώσεις. Όλοι που θέλουν μπορούν να είναι με αυτές τις διαδικασίες. Όλοι αυτοί οι οποίοι αναπτύσσουν πρότυπα θέλουν να εξασφαλίσουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες της δημιουργίας προτύπων. Πολλές φορές έχουμε Εκατοντάδε ατόμων τα οποία συμμετέχουν σε τεχνικέ επιτροπέ, προετοιμασία. πρότυπων. Αυτό εξασφαλίζει ότι αυτά τα πρότυπα ενσωματώνουν τι πιο καινοτόμε προσεγγίσει την τελευταία ε, ε, ε στιγμή τεχνολογία και την τεχνολογία χμής. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται και η δυνατότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να συμμετέχουν μέσα από το διαδίκτυο και έτσι δεν έχουν άχθος διοικητικό ή έξοδα ταξιδίου. Με την λειτουργία αυτή μέσω από το διαδίκτυο υπάρχουν μεγαλύτερε δυνατότητε για να μπορούν να συμμετέχουν και οι καταναλωτέ στη διεργασία αυτή. Το σύστημα προτύπων των Ηνωμένων Πολιτειών βασίζεται και καθοδηγείται από τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει όμως να τονίσω ότι και η Αμερικανική κυβέρνηση είναι ένας σημαντικός χρήστης προτύπων και συμμετέχει απόλυτα ενεργά στην διαμόρφωση των προτύπων αυτών. Η Άνση πάντα θέλει να έχει μια σχηρή εταιρική σχέση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτής της εταιρικής σχέσης είναι η νομοθεσία για την τεχνολογία για τη μεταλαμβάνευση τεχνολογίας και την πρόοδο, το NTTAA. Ο στόχο είναι να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για πρόθεση τεχνολογικών καινοτομιών. Μετά από την έγκριση αυτή τη νομοθεσία στην δεκαετία του 1990 έχει υπάρξει με τη συμμετοχή τη κυβέρνηση μεγαλύτερη λειτουργική ικανότητα και έχουν μειωθεί σημαντικά το κόστο των δημοσίων προμηθειών. Πάνω από χίλια τέτοια πρότυπα έχουν ενσωματωθεί με τον τρόπο αυτό σε εθνικού κανονισμού, Σύμφωνα με τον νόμο αυτό και το Α91, το, την εγκύκλιο που συνοδεύει αυτό τον νόμο, για να χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν πρέπει να αναφέρεται στο έγγραφο αυτό περί προτύπων. Η Υποεπιτροπή των Εθνικών Προτύπων για τα θέματα αυτά δημοσίευσε μια έκθεση που αφορά τις ε, εθνικές προδιαγραφές και τις ε, εθνικές δεσμεύσεις για τα θέματα αυτά και αυτό το έγγραφο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο ίντερνετ. Αυτό το έγγραφο δείχνει ποιο είναι το πλαίσιο, το πολιτικό και το νομικό για την συμμετοχή της κυβέρνησης σε ιδιωτική διαδικασία τυποποίησης και καταδεικνύει ποιε είναι οι κύριε κατευθύνσει πολιτική από το Λευκό Οίκο προ την κατεύθυνση τη συμπλήρωση των κατευθυντήριων γραμμών προ του εθνικού φορεί. Ανοιχτό χαρακτήρα, ισορροπία, ισορροπία συνένεση, ισοδίκαια συμμετοχή, όλα αυτά βοηθούν να υπάρχει ένα πλαίσιο χωρίς διακρίσεις για να υπάρξει και προστασία των πνευματικών ε, δικαιωμάτων. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αμερικανικής διαδικασίας που είναι πάρα πολύ σημαντικά όταν μια εθνική δημόσια αρχή πρέπει να αναφερθεί σε πρότυπα μέσα στους κανονιστικούς, μέσα στους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις της. Όλες αυτές οι αρχές λοιπόν που αναφέρθηκα εκμετα... Ε, τη χάνουν εκμετάλλευσης με στο πλαίσιο αυτό. Έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση και ένα ενιαίο πλαίσιο που αντανακλάται σε αυτό το έγγραφο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους εμπλεκομένους σε επίπεδο ΗΠΑ για να επιτύχουμε τους κατάλληλους στόχους τεκμηρίωσης και τυποποίηση. Οποιοδήποτε τομέα τη βιομηχανία μπορεί να αποφασίσει τι αποτελεί επιτυχή τυποποίηση σε σχέση με τους δικούς του εμπλεκομένου το ANSI είναι πλήρως προσιλωμένο σε ένα σύστημα στο οποίο οι ανάγκες της κοινωνίας καθορίζουν την χρονική αλληλουχία και το περιεχόμενο της τυποποίησης και βασίζεται στην επίτευξη συνένεσης για αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουμε ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την, ε, τις απαιτήσει ελέγχου ε, συμμόρφωση με τα πρότυπα και έχουμε και ένα έγγραφο το οποίο εξηγεί τη διαδικασία που ακολουθούμε για τον έλεγχο τη συμβατότητα και τη συμμόρφωση. Όταν μιλάμε επίση και για την παγκόσμια τυποποίηση δεν αναφερόμαστε μονάχα στο ISO και στην IEC. Πρόκειται για πρότυπα τα οποία συμμορφώνται με τι βασικέ αρχέ του ΠΟΕ σε σχέση με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο έχουν μεγάλη σημασία για μας και εμείς υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα τις αρχές αυτές που αναφέρονται εδώ. Εν τέλει, η αρχή μας είναι ότι υπάρχουν πολλαπλοί δρόμοι για να υπάρξουν παγκόσμια πρότυπα, είτε αυτά που αναπτύσσονται με το μοντέλο της εθνικής εκπροσώψης, με το μοντέλο της άμεσης εκπροσώψης ή με την ανάπτυξη από κονσάρτσια. Όλα αυτά θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς και δεν θα πρέπει ποτέ να αποτελούν φραγμού στο εμπόριο. Το σύστημα προτύπων των ΗΠΑ είναι ανοιχτό και προσβάσιμο και έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σαν υπόδειγμα. Το... Οι Ηνωμένε θέλουν να, να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα όχι μόνο των Αμερικανών, αλλά να υποστηρίξουν ένα παγκόσμιο σύστημα εμπορίου που είναι ισορροπημένο και χωρί φραγμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή. Χαίρομαι που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να λάβω το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την διεξοδικότατη παρουσίαση και πραγματικά στα 8 λεπτά που σας δώσαμε ήσασταν ιδιαίτερα εύστοχοι. Προφανώ, πολλοί από εμά θα προσπαθήσουν σήμερα να βρουν τα έγγραφα που αναφέρατε στο διαδίκτυο. Πάντω, η δεσμευσή σα για τι αρχέ του ΠΟΕ είναι κάτι που νομίζω ότι θα το εκτιμήσουν όλοι εδώ. Και θα το ακούσετε μετά και στον χρόνο των ερωταπαντήσεων. Τώρα, ο κύριο Φeng Τσουν Κουάν, συγγνώμη για την προφορά μου στα κινέζικα, σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και με τα χαρά σα δίνω το λόγο για 6 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το όνομά μου είναι Και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας σήμερα και έχω αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την τυποποίηση στην Κίνα. Εκ μέρους του κυρίου Τσέινγκ που είναι υπεύθυνος και το όνομά του βλέπετε στην οθόνη, θα ήθελα στην παρουσίασή μου να επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα το τι γίνεται με τη διαδικασία προτύπων στην Κίνα και έπειτα η ευθυγράμμιση, η συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα. Σε πρώτη φάση λοιπόν, τι γίνεται με την κινέζικη τυποποίηση. Τρία στοιχεία, βασικά στοιχεία. Πρώτον, το εθνικός φορέας προτύπων, εθνικός φορέας τυποποίησης στην Κίνα. Υπάρχουν δύο επίπεδα εδώ. Το εθνικό όπου με την έγκριση του, της κυβέρνησης ο φορέας τυποποίησης της Κίνας ασκεί την διαχείριση της διαδικασίας τυποποίησης σε εθνικό επίπεδο και εκπροσωπεί την Κίνα σε δραστηριότητες της ΆΙΖΟ, της IC και άλλους διεθνείς και περιφερειακούς φορείς τυποποίησης. Τώρα, το επίπεδο των περιφερειών, των επαρχιών, οι τοπικές κυβερνήσεις αναλαμβάνουν, μάλλον οι υπηρεσίες ποιότητας και τεχνικής ε, παρακολούθησης, αναλαμβάνουν την τυποποίηση εντός της κάθε ξεχωριστής επαρχίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της έγκρισης, της απαρίθμησης, της ε, καταχώρησης δηλαδή, της διάδοσης και της καταγραφής των προτύπων. Να επικεντρωθώ τώρα στο εθνικό επίπεδο. Οι βασικές ευθύνες του Εθνικού Φορέα Τυποποίησης ε, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νομοθεσίας για την τυποποίηση, την θέσπιση στατηγικών στόχων για την τυποποίηση στην Κίνα, μαζί με τον συντονισμό και την ανάπτυξη, καθώς και την αναθεώρηση των εθνικών μας προτύπων. Τρίτον, η έγκριση των εθνικών προδιαγραφών. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την ε, στενή συνεργασία με τις ε, επιτροπές τεχνικού, ε, με τις τεχνικές επιτροπές που παρακολουθούν την επιστημονική πρόοδο επίσης τον συντονισμό της καταγραφής ανατομεία ε, και σε τοπικό επίπεδο, την επίβλεψη της υλοποίησης των εθνικών προτύπων, τη διαχείριση των εθνικών πληροφοριών για την τυποποίηση. Επιπλέον υπάρχει εκπροσώπηση της Κίνας ώστε να συμμετέχει ο φορέας αυτός, τον ΆΙΖΟ, την ΟΕΣΥ και άλλους ε, διεθνείς και περιφερειακούς φορείς τυποποίησης Μπορεί έτσι να υπογράφει ο φορέα και να υλοποιεί διεθνή συμφωνίε συνεργασία που την τυποποίηση. Η δεύτερη πτυχή που θα ήθελα να αναπτύξω είναι η διαχείριση της τυποποίησης στην ε, Κίνα. Βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα πώς έχει το σύστημα τυποποίησης στο κάτω μέρος του διαγράμματος υπάρχει η Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την δημιουργία προτύπων. Είτε με ίδια πρωτοβουλία, είτε μετά από αίτηση των ε, ενδιαφερόμενων φορέων. Επαρχιών, λόγου ή περιφερειών ή υπουργείων δηλαδή κυβερνητικών υπουργείων ή κατόπιν αιτήματο του Εθνικού Φορέα Τυποποίησης. Εάν τώρα η πρόταση υιοθετηθεί από μια επαρχία ή αυτό θα είναι ένα πρότυπο που θεωρηθεί τοπικό ε, στην Κίνα, εάν εγκριθεί από τον Εθνικό Φορέα, θα θεωρηθεί τομεακό. Μάλλον ε, θα θεωρηθεί εθνικό σε αυτή την περίπτωση, ενώ από το συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο θα θεωρηθεί τομεακό πρότυπο. Να εξηγήσω ότι ως τώρα υπάρχουν συνολικά 497 τεχνικές επιτροπές στην Κίνα πραγματικά θα ήθελα πολύ να μα παρουσιάσετε όλε τι διαφάνειε μία-μία, αλλά μήπω να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα, να δούμε τη διεθνή διάσταση, γιατί αυτό μα ενδιαφέρει περισσότερο. Καλά. από την ε, ίδρυση του Εθνικού φορέα το 2001, η τυποποίηση στην Κίνα έχει πάει πολύ καλά. Οι σχετικέ εργασίε στηρίζονται από την κυβέρνηση, καθορίζονται από τι ανάγκες της αγορά, συντονίζονται από τους βιομηχανικού κλάδους, τα ε, ιδρύματα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ε, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια και βεβαίως υπάρχει συμμετοχή της αγοράς και όλων των ενδιαφερομένων. Τα εθνικά μας πρότυπα σχεδιάζονται και πολλά από τα πρότυπα στον τομέα της ε, διατροφικής ασφάλειας, της προστασίας των καταναλωτών, της τεχνικής και τεχνολογικής προσαρμογής και ανανέωσης των ε, τεχνολογιών εχμής, των πόρων και της ενεργειακής ε, αποτελεσματικότητας. Όλα αυτά αναπτύσσονται γοργά. Το δεύτερο λοιπόν θέμα που ήθελα να σα παρουσιάσω σήμερα ήταν η ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα. Η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην έγκριση των διεθνών προτύπων. Αυτό εφόσον έχουν αποδειχθεί χρήσιμα. Όταν λοιπόν προτάσει υποβάλλονται από τα, για μάλλον τα εθνικά πρότυπα υποβάλλονται στον εθνικό μα φορέα τυποποίηση, Στόχος είναι να υπάρξει ευθυγράμμιση και συντονισμός με τα διεθνή πρότυπα. Έπειτα η ενημέρωση των εθνικών φορείων, των εθνικών προτύπων και των, ε, ανάλογα με τα διεθνή είναι διαδικασίες συνήθως ταχείες. 80% των ε, τομέων του χάλιβα και του ατσαλιού, των ε, ηλεκτρικών συσκευών, ε, των ναυπηγικών, των εργαλείων και των μετρητών. Επίσης 98,5% εκπροσωπεί άλλους 12 τομείς που έχουν όλα ήδη μελετηθεί και εγκριθεί πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η έγκριση διεθνών προτύπων έχει βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων, έχει ενισχύσει την ε, παραγωγικότητα, την ε, προστασία και την ασφάλεια. Η προστασία λοιπόν της ανθρώπινης και της ζωικής ευζοίας είναι σημαντικά στοιχεία γιατί θέλουμε να αρθούν οι τεχνικοί φραγμοί για ε, το διεθνές εμπόριο. Θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε. Ήδη έχετε ξεπεράσει τα 8 λεπτά και πρέπει να κάποια στιγμή να κλείσουμε. Τις έχουμε τις διαφάνειές σα, αν θα τις διαβάσουμε αν είναι. Έχω μόνο τέσσερις ακόμα. Να σταματήσω. Ναι. Πρέπει να σας ευχαριστήσω. Σίγουρα θα έχετε ερωτήσει μετά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλιά σα. Αλλά δεν θα είναι δίκαιο για του υπόλοιπου ομιλητέ. Σα ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερω. Uh, uh, και τώρα ο κύριος Ντόσετ από την Σένελεκ, γνωστός σε όλους μας. Για έξι λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την συγκεκριά για την πρόσκλησή της. Απλώς να πω λίγα λόγια για τις ε, διεθνείς διασυνδέσεις της ΕΝΣΕΝΕΛΕΚ, κυρίως με την ΆΙΖΟ και την ΆΙΣΗ. Αυτοί είναι οι οργανισμοί που υπάρχουν σε εθνικό και διεθνέ επίπεδο ουσιαστικά και βλέπετε ότι υπάρχει συμφωνία της Βιέννης μεταξύ ΑΙΖΟ και ΣΕΝ ενώ της Δρέσδης μεταξύ των άλλων δύο φορέων. Οι αρχές των συμφωνίων αυτών ε, αναφέρονται στην οθόνη είναι ουσιαστικά να μην υπάρξει επεκάλυψη των εργασιών στα δύο επίπεδα, να υπάρχουν πάνω πανομοιότυπα πρότυπα και στην Ευρώπη και παγκοσμίω, εφόσον αυτό είναι δυνατό, να ε, θεσπίζονται συμφωνίες βάσει των πρωτοκόλων μα για την κατανομή των εργασιών, στην Ευρώπη και το διεθνέ επίπεδο ένα από τα δύο μάλλον και όχι και στα δύο ταυτόχρονα και βεβαίως να υπάρχει ταυτόχρονη διαδικασία έγκρισης με συγκεκριμένες προτάσεις για τα πρότυπα. Τα αποτελέσματα των συμφωνιών τώρα. Για την ε, Συμφωνία της Βιέννης αναφέρονται ήδη εδώ. Βλέπουμε ότι 30% του χαρτοφυλακίου τη ΕΝ είναι πανομοιότυπο με τα πρότυπα τη ΆΙΖΟ. Ενώ αν δούμε τη συμφωνία τη Δρέσδης με τη ΣΕΝΕΛΕΚ, περισσότερο από 20 χρόνια από την Βιέννη έχουμε φτάσει το 75 περίπου τη 100 πανομοιότυπων ή πολύ συγκλινόντων προτύπων μεταξύ ΣΕΝΕΛΕΚ και ΆΙΖΟ. Τώρα, εάν δούμε τα εναρμονισμένα πρότυπα, δηλαδή πρότυπα που παράγονται ανάλογα με τι απαιτήσει τη νομοθεσία, Το 20% των εναρμονισμένων προτύπων είναι πανομοιότυπα με την ISO, ενώ αν δούμε τι γίνεται με την IEC, είναι περίπου το 75% των προτύπων που έχουν πια γίνει πανομοιότυπα ή προσωμιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα, τα πλεονεκτήματα των ε, συμφωνιών αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι καθορίζουν ποια είναι τα πρότυπα που χρειάζονται σε διεθνέ και ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα η διαδικασία ορίζεται βάσει των αναγκών και των προτεραιοτήτων των ε, ενδιαφερομένων. Έπειτα η εναρμόνιση των χαρτοφυλακίων των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων επιτρέπει την εξαγωγή προτύπων προς άλλες περιοχές και επίσης διασφαλίζουν τα προϊόντα που έρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά βρίσκονται στην, ε, ε, κοντά στην πραγματικότητα και στην επικαιρότητα και υποθέτουμε ακριβώς λόγω της σύγκλησης των προτύπων ότι είναι συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανόνες. Πιστεύουμε ότι οι συμφωνίες αυτές και η επιτυχής υλοποίησή τους σημαίνουν ότι η ΣΕΝ και η ΣΕΝΕΛΕΚ είναι οι πλέον επιτυχημένοι περιφερειακοί συνεργάτες για την ΆΙΖΟ και την ΆΙΣΥ. Επίσης, πέραν των επίσημων συμφωνιών μας καθορίζουμε σχέσεις συνεργασίας και για την ε, διεθνή εναρμόνιση προκειμένου να ανοίξει η ευρωπαϊκή αγορά για διεθνείς ε, κατασκευαστές, να αρθούν οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο, να μην υπάρχουν ε, τελωνιακά θέματα μεταξύ των χωρών των περιοχών, να υπάρξουν διεθνείς πλατφόρμες συνεργασίας και να βελτιωθεί η υποδομή ποιότητας. Αυτό σημαίνει συμμετοχή, συνεργασίες και μνημόνια συνεννόησης, ε, συνεργασία μεταξύ των ε, περιφερειακών τομέων, ε, των ρυθμιστικών και τεχνική υποστήριξη προς άλλες περιοχές του κόσμου. Ως αποτέλεσμα του συνολικού μας προγράμματος, το βλέπετε και στο διαφάνεια, έχουμε 19 μέλη πλέον από τις ε, χώρες τη Ευρωπαϊκή Γειτονία όπως ονομάζονται, ε, τα σχέσεις ε, συνεργασίας με την Αυστραλία νομίζω, προγράμματα προβολής όπως λέγονται, μαζί με συνεργάτες από με τους συναδέλφους μου από την έτσι, στην Κίνα λόγω χάρη και σύντομα θα δημιουργηθεί ένα και στην Ινδία. Το ανέφερε και κάποιος βουλευτής νωρίτερα Εδώ λοιπόν οι προτάσει τη Επιτροπή σχετικά μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερω. Υπάρχουν, υπάρχουν τακτικέ ανταλλαγέ με την Άνση. Συναντηθήκαμε μόλι πριν από ένα δεκαπενθήμερο και υπάρχουν μνημόνια κατανόηση και συμφωνίε συνεργασία με πολλέ περιοχέ του κόσμου. Την ε, Ήπειρο τη Αμερική, την Αφρικανική, τη Ρωσία και τον φορέα τυποποίησή τη, με τα κράτη του κόλπου με την SAC στην Κίνα, την Κορέα, τον Καναδά, την Ιαπωνία. Με όλου αυτού του διεθνεί εταίρου έχουμε διμερεί διευθετήσει τη συμφωνίε. Και απλώ για να δείτε την επίδραση των ευρωπαϊκών προτύπων παγκοσμίω, αυτή η εικόνα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δείχνει ότι για του ανελκυστήρε ε, τα ευρωπαϊκά πρότυπα χρησιμοποιούνται σχεδόν παντού στον υπόλοιπο κόσμο. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και τον χρόνο σα, Πρόεδρο. Αρχίσατε, αρχίσαμε νωρίς, οπότε είστε εντό χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσίασή σας. Και είδαμε επίσης ότι ε, η δουλειά σας συνεργάζεται ε, και με το Μιστίν Κίνα. Τώρα θα ακούσουμε την παρουσίαση του κυρίου Βάιλερ από την ΕΤΣΙ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που δώσατε σε μένα και στην ΕΤΣΙ για να συμπληρώσουμε τις ε, απόψεις των άλλων οργανισμών τυποποίησης με τις δικές μας. Ε, οφείλω να πω πως ε, χαίρομαι πάρα πολύ ότι ο Μάλκομ έχει την ίδια γραβάτα με εμένα, η οποία είναι γραβάτα της έτσι. Βασικά θέλω να αναφερθώ σε τρία σημεία. Η έτσι καλωσορίζει τη μεταρρύθμιση του συστήματος ευρωπαϊκής τυποποίησης και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κομισιόν που μας παρήχε αυτό το σχέδιο και το όλο πακέτο. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις της Επιτροπής και για τις δημόσιες προμήθειες και για την ε, ρύθμιση υπό ορισμένες συνθήκες όπως η ε, διαφάνεια, η προσβασιμότητα διότι εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την ε, παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρατήσει την βιομηχανία ανταγωνιστική ε, όσον αφορά την ε, τυποποίηση. Έτσι λοιπόν θα δοθεί η δυνατότητα στα πρότυπα να γίνουν ευρέως δεκτά, ανεξάρτητα από το πού προέρχονται, είτε από κονσόρτια είτε από αλλού και ταυτόχρονα μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τις ε, περιφερειακές απαιτήσεις που υπάρχουν. Έπειτα, ε, θα ήθελα να πω ότι αναμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τα δικά της ε, σώματα για να διαδώσουν τις ανάγκες της τυποποίησης και αυτές οι ανάγκες είναι διαφορετικές ανατομέα. Εδώ η βιομηχανία ICT διαφέρει από τους άλλους τομείς έχει ε, έχει πολύ μεγάλες ε, διαφορές και αν θυμάστε ίσως έτσι δημιουργήθηκε το 1988 κατόπιν συνένεση της ε, Κομισιόν των Κρατών Μελών και της, των αντιπροσώπων των... της βιομηχανίας έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σώμα στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την δημιουργία κοινών προτύπων. Και αυτό έχει φέρει την Ευρώπη σε ηγετικό ρόλο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καταρχάς δημιουργώντας πρότυπα υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη και μετά καθιστώντας τα παγκόσμια και συνεργαζόμαστε με άλλους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίηση, για παράδειγμα την CCSA στην Κίνα. Ήταν ένας οργανισμός πιστοποιημένος από την Άντζη επίσης με την Ιαπωνία και την Κορέα. Τώρα έχουμε 5,3 δισεκατομμύρια χρήστες ε, κινητής τηλεφωνίας, συστήματα GSM και LTA. Και έχουμε πάνω από 90 συμφωνίες με διά, συνεργασίες με διάφορους οργανισμούς. Επίσης χρησιμοποιούμε ε, την διεθνή συνεργασία, τις διεθνείς σχέσεις με τους άλλους οργανισμούς για την επίτευξη των στόχων μας. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, βλέπουμε την σημασία της, ε, του ορισμού του πώς τα πρότυπα αυτά θα γίνονται δεκτά σε ευρωπαϊκά πλαίσια για τις δημόσιες προμήθειες. Υπάρχει η πλατφόρμα διαβούλευσης με, το, ε, με τους ενδιαφερόμενους, υπάρχει η διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και επίσης είναι σημαντικό να, καθορίσουμε, να, να διασφαλίσουμε ότι θα, η διαδικασία θα είναι διαφανής. Και ελπίζουμε αυτή η πλατφόρμα Ελπίζουμε να ανακοινώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου ότι η πλατφόρμα αυτή θα αρχίσει να λειτουργεί από τις αρχές του επόμενου και το αργότερο όταν ο κανονισμός θα υιοθετηθεί το 2013. Θα ήθελα τώρα να κάνω ένα άλλο σχόλιο σχετικά με την συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αντίθετα με αυτά που ακούσαμε πριν, στην ΕΤΣΙ και στο project ε, συνεργασίας τρίτης γενιάς ανάπτυξης ε, προτύπων κινητής τηλεφωνίας, η συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί παρά μειωθεί. Α, θα ήθελα λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι βλέπουμε τα πρότυπα και τις ε, προδιαγραφές να αναπτύσσονται πολλές φορές ε, θελοντικά από τη βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο για την παγκόσμια αγορά. Ο στόχος του, ε, αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου θα είναι να επηρεάζεται η αγορά όπου αυτό χρειάζεται για να διασφαλίζεται η υγιής ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ε, για, το πώς η, ε, για το πώς η έτσι κάνει σωστά τη δουλειά της λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Εν τέλει ο David Wilkinson από το KKR, από το Κοινό Συμβούλιο ε, Ερευνών. Βλέπω ότι έχεις πολλέ πολλές αλλά ίσως πρέπει να συντομεύσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που εμπλέκεται και το Κοινό Κέντρο Ερευνών σήμερα εδώ στην σημερινή ακρόαση. Όπως ξέρετε, είμαστε το, αν θέλετε, το εντό των τυχών κέντρο ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνουμε την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στην ε, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων πολιτικών. Γιατί τώρα εμπλεκόμαστε στη διαδικασία τυποποίησης. Το κλειδί αυτής της διαδικασίας είναι το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν πολλές διαδικασίες τυποποίησης, πολλές, ε, πολλά πρότυπα που απαιτούν το να εξασφαλίσουμε και μία εξισορρόπηση της αποτελεσματικότητας, της ανταγωνιστικότητας της ε, βιομηχανίας από την μια πλευρά, αλλά από την άλλη μεριά την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία και μια αλληλεπίδραση μεταξύ της διαδικασίας της ρύθμισης και των αναγκών της βιομηχανίας. Εδώ το κομβικό θέμα είναι ότι πολλέ φορέ η επιστημονική γνώση μπορεί να μα δώσει τα κέρια στοιχεία για να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η συνολική ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί. επομένω το Κοινό Κέντρο Ερευνών κάνει διαδικασίες προτυποποίησης, προσπαθεί να εξασφαλίσει την εναρμόνιση των μεθοδολογιών, δίνει άμεση τεχνική και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη που χρησιμοποιούν οι φορείς τυποποίησης. <clears throat> Πολλές φορές προχωρούμε και σε δράσεις πιστοποίησης. Το άλλο το οποίο σημαντικό είναι ότι μπορούμε να επαναλάβουμε και να επιβεβαιώσουμε διαδικασίες αναφοράς μέτρησης ε, που είναι χρήσιμε στα πρότυπα. Για να σα αναφέρω τους τομεί που εργαζόμαστε. Ενέργεια και μεταφορές είναι στην κορυφή τη ατζέντα, ψηφιακή ατζέντα, ασφάλεια και προστασία από κινδύνους εν γέννη. Πολύ σημαντικό είναι η προστασία των καταναλωτών, όπου έχουμε παραγάγει σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν για τον ορισμό των υλικών. Ένα παράδειγμα μονάχα. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών εδώ και πολλά χρόνια έχει το εργαστήριο δοκιμασίας στην Ίσπρα που αντιμετωπίζει τη μεθοδολογία της ε, καταμέτρησης των εκπομπών ρήπων από αυτοκίνητα οχήματα. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διαδικασία τυποποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε ήδη στο πακέτο της Κομισιόν ότι υπάρχει μια να υπάρχει ένα σαφή ρόλο για το κοινό κέντρο ερευνών. Λέει ότι το κοινό κέντρο ερευνών θα δώσει επιστημονικά στοιχεία και την εμπειρογνωμοσύνη του για να εξασφαλίσει ότι τα πρότυπα λαμβάνουν υπόψη και την οικονομική παραγωγικότητα αλλά και τι κοινωνικέ ανάγκε όπω είναι η βιωσιμότητα του περιβάλλοντο, η ασφάλεια των πολιτών κτλ. Υποστηρίζουμε ιδιαίτερα επίση μία διαδικασία προ, αντιμετώπισης των νέων προτύπων τα οποία θα χρειαστεί να εφαρμοστούν στο μέλλον από την Κομισιόν. Όλο και περισσότερο το θέμα αυτό παίρνει ένα πιο παγκόσμιο χαρακτήρα, Επομένω και η προσέγγιση μα πρέπει να γίνει πιο παγκόσμια. Η βιομηχανία και η μεταποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται πιο παγκόσμια και αν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορέ, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη ισορροπία, θα πρέπει να έχουμε τη σωστή επιστημονική βάση αλλά και σε πιο παγκόσμιο επίπεδο για να υποστηρίξουμε αυτά τα πρότυπα. Ένα τμήμα της αποστολής μας λοιπόν είναι ακριβώς να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτήν την σωστή ισορροπία, ιδίως σε μια στιγμή που συνεργαζόμαστε με συναδέλφους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και ένα μνημόνιο προθέσεων την επόμενη εβδομάδα που θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο και θα μπορέσουμε να έχουμε τα θεμέλια επί των οποίων θα μπορέσουν να εδράζονται τα ε, πρότυπα για την ηλεκτρονική κινητικότητα και τα εφή e δίκτυα πληροφορίας. Βλέπετε ότι έχουμε πολλούς φορείς οι οποίοι εμπλέκονται και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού. Είναι σαφώς ότι αυτό είναι ένα κομβικό θέμα για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης των οικονομιών μας. Και είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε τα σωστά τεχνικά πρότυπα γιατί η βιομηχανία μπορεί να κάνει σωστές επενδύσεις όταν ξέρει ποια θα είναι η μορφή και η διαμόρφωση των προτύπων στο μέλλον και πώς θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη ισορροπία. Λοιπόν, το μήνυμα που μας δίνουν οι βιομηχανίες, οι, βιομηχανοί και από τις δύο πλευρές και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού είναι πράγματι να υπάρξει και μία συμμετοχή των δημοσίων αρχών για τον καθορισμό των προτύπων. Αυτό το οποίο θα δημιουργηθεί είναι θα έχουμε δύο κέντρα διαλειτουργικότητας ένα στην Ίσπρα στην Ιταλία κοντά στο Βαρέζε και το άλλο στο Εθνικό Εργαστήριο Argon κοντά στο Σικάγο, το οποίο το διαχειρίζεται το Εθνικό ε, η Εθνική Υπηρεσία Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να έχουμε την ε, βασική επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη που πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να βοηθήσει τις βιομηχανικές το βιομηχανικό, τους βιομηχανικούς φορέας, φορείς για να έχουμε τα κατάλληλα πρότυπα. Θέλουμε να καταλήξουμε σε παγκόσμια πρότυπα. Έχουμε ξεκινήσει βέβαια με μια εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά τώρα εργαζόμαστε και πιο πολύ με τους εταίρους μας στις ΗΠΑ. Θα θέλαμε όμως να διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία και στη συνέχεια για να συμμετάσχουν και άλλα μέρη του κόσμου. Δεν θα μπω τώρα στα τεχνικά διαγράμματα, γιατί αλλιώς θα θέλουμε τουλάχιστον μισή ώρα παραπάνω. Θα τα καταπιώ λοιπόν και θα φτάσω στο συμπέρασμα. Το συμπέρασμα μου είναι ότι τα πρότυπα είναι κομβικά για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, ανταγωνιστικότητας και για την παγκόσμια παραγωγικότητα. Η επιστήμη είναι απαραίτητη βάση για τα καλά πρότυπα. Πρέπει να προχωρήσουμε τρίτον σε ένα πιο παγκόσμιο τρόπο προσέγγισης και τέταρτον το κοινό είναι τμήμα του, της δομής της Κομισιόν γιατί δίνει τις κέρυες επιστημονικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τη δημιουργία των προτύπων και τη διεθνοποίηση της διαδικασίας διαμόρφωσης προτύπων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους, λέει ο Μαρκόμ Χάρμπορ. Συγγνώμη που μείναμε από χρόνο, στο τέλος. Ούτε ερωτήσεις, ούτε απαντήσεις θα μπορέσουμε να έχουμε. Φαντάζομαι ότι κάποιοι συνάδελφοι θα έρθουν να σας μιλήσουν αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τονίσαμε και την παγκόσμια διάσταση στη συνεδρία σήμερα το πρωί. Υπήρξε ίσω ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, αλλά όλα αυτά είναι μια πολύ καλή βάση για τους συναδέλφους μου και είναι πολύ θετικό ότι φέραμε το Κοινό Κέντρο Ερευνών για πρώτη φορά σε αυτό το πλαίσιο και επίσης χαιρόμαστε για τις διατλαντικές συμφωνίες οι οποίες θα υπογραφούν την επόμενη εβδομάδα. Αυτό το οποίο προτείνω λοιπόν είναι να προτείνω στην συγγήτριά μας την κυρία Λάρα κόμη να κάνει απλώς μερικές καταληκτικές παρατήρησεις και μετά θα σας δώσουμε το χρονοδιάγραμμα για το επόμενο στάδιο των δραστηριοτήτων μας και θα προσκαλέσω όλους τους καλεσμένους μας και όσους άλλους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν να εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Λάρα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξανά θέλω να ευχαριστήσω όσους συνεισέφεραν οι παρουσιάσει του ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε και αναγκαίε και για μένα και για τους σκιώδη εισηγητές, διότι από αύριο, δηλαδή από σήμερα το απόγευμα, θα αρχίσουμε να συμπληρώνουμε το σχέδιο της πρότασης. Όλοι μαζί, ώστε να είναι όσο το δυνατόν η θέση μας πιο συμπαγής και πιο συνενετική. Σας ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερος. Στο πρώτο τμήμα της ε, ακρόασης εκτιμήσαμε την ανάγκη για ταχύτητα που δεν πρέπει όμως να ζημιώσει την ποιότητα. Άρα, ε, πολλές φορές ε, πρέπει να διευκρινίζουμε ότι το γοργόν και χάρη να έχει και το εύστοχο για ορισμένους τομείς πρέπει να είναι και ταχύ. Επίσης, επικεντρωθήκαμε στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις μα απασχόλησε αν μπορούν να εκπροσωπηθούν καλύτερα με δικαίωμα ψήφου και πώ σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον μπορούν να ε, ομαδοποιηθούν, να συγκεντρωθούν καλύτερα και να συντονιστούν μεταξύ του. Αυτό ευθύ εξ αρχή το είχαμε συμμεριστεί ότι θα πρέπει να ξεκινούμε από το εθνικό επίπεδο για να καταλήγουμε στο ευρωπαϊκό. Με μια δομή την οποία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεχτεί με την ε, έκθεση πρωτοβουλία που έχουμε ετοιμάσει για αυτό το θέμα. Διατηρώντα βεβαίω και την ιδιωτική τη διάσταση και την εθελοντική. Να διευκρινίσω εδώ ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στι διαφορετικέ διαδικασίε μεταξύ τη εκπροσώπηση διαφορετικών κατηγοριών. Κάποιε φορέ επικεντρωνόμαστε στι μικρέ αντιδιαστολή με τι μεγάλε επιχειρήσει, αλλά μάλλον πρέπει να διακρίνουμε καλύτερα τομεί. Από αυτό εξαρτώνται τα πρότυπα και η ποικιλία, καθώ και η χρόνη ταχύτατα τώρα. Το πρόβλημα της εκπροσώπησης όπως θα εξελιχθεί και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ δεν ε, έχω αντίρρηση ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του GRC, όπως ε, έχει αναφερθεί και σε άλλες ευκαιρίες με το 8ο πρόγραμμα πλαίσια για την έρευνα για καινοτομία. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι και ούτε εγώ μπορώ να το αρνηθώ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να μην δοθεί μεγαλύτερη εξουσία σε αυτές τις επιτροπές από ότι τον ιδιωτικό τομέα της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Είδαμε άλλωστε ότι άλλοι πολλές φορές που αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες ε, ήρθαν κάποιες φορές οι ΗΠΑ, όπως βλέπουμε τώρα τις ΗΠΑ, να μας την πάνε την πόρτα για να μας δώσουν ιδέες, αλλά εμείς θα πρέπει επίσης να είμαστε πηγή έμπνευσης για τους υπόλοιπους. Βεβαίω χρειάζεται και απλούστευση του συστήματο των προτύπων και η τόνωση τη ανταγωνιστικότητα με τη δημιουργία μια πλατφόρμα ώστε να υπάρχει ομοιογένεια για όλου του και ισότιμη όρη για όλου του ε, ενδιαφερόμενους με εκπροσώπηση των πάντων, έπειτα συντονισμός μεταξύ διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων. Το τελευταίο τμήμα της ακρόασης νομίζω ήταν από τα πλέον σημαντικά, διότι μας ενδιαφέρει ακριβώς η παγκόσμια διάσταση, εμένα και τους υπόλοιπους και Μιλάμε εδώ για ευρωπαϊκά πρότυπα υψηλότατης ποιότητας μεν, καλό αυτό, αλλά θέλουμε να τα συμμερίζεται και ο υπόλοιπος κόσμος. Θέλουμε να επικεντρωθούμε στη διεθνή διάσταση. Αυτή ήταν, αυτό το κενό είχαμε. Αυτό μα έλειπε ω στοιχείο. Ήταν πολύ ευχάριστο λοιπόν σήμερα να ακούσουμε με τι προθυμία μα παρουσιάσατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία στο τελευταίο αποφασιστικό τμήμα τη ακρόαση. Είμαι στη διάθεση όλων για όσου θέλουν να συνεισφέρουν περαιτέρω σε σχέση με τα όσα συζητήσαμε σήμερα. Απλώ μια προθεσμία και το χρονοδιάγραμμα θα σα το δώσει ο πρόεδρο Σα παρακαλώ να έχετε την ευγενή καλοσύνη, αν έχετε περαιτέρω απόψεις, Άλλε προτάσει. Μέχρι τι 5 Δεκεμβρίου να τι υποβάλλετε. Γιατί έχουμε μετά τι τελικέ συναντήσει για να ετοιμαστεί το σχέδιο του κειμένου με τους σκιώδει εισηγητέ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο ώστε μετά να παρουσιαστεί το σχέδιο έκθεση. Σα ευχαριστώ ειλικρινώς. Ήταν πολύ χρήσιμο για μένα η σημερινή ημέρα και αγγίξαμε και πτυχές που στην προηγούμενη ακρόαση δεν τις είχαμε καν σκεφτεί. Εδώ λοιπόν έχουμε μια εικόνα πανοραμική των προτύπων, 360 μοιρών. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε κοινέ θέσει. Well, like Σας ευχαριστώ, κύριε Κόμη, που αναλάβατε τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης μαζί με τον Κώστα από τη Γραμματεία βρίσκεται δίπλα μου και τους συναδέλφους. Ε, κλείνοντας την ακρόαση να σας αναφέρω το χρονοδιάγραμμά μας για το πώς θα προχωρήσουμε όπως η Πιλάρα. Θα συντάξει τον κατάλογο με τις τροποποιήσεις αφού συζητήσει με τους σκιώδεις συζητές. και η κυρία Κοζίσνη, που πολύ γνωρίζεται από την έκθεση για τη στρατηγική θα συμμετάσχει ε, ενεργά εδώ. Υπάρχει λοιπόν ε, με την κυρία Μάντερ, την κυρία Ρούλα, την κυρία Σάλντερ Μόζε, την κυρία Γκυγιόμ. Ε, θα υπάρξει εξακολούθηση τη ειδική γνώση που υπήρχε και στην προηγούμενη φάση και μετά η κυρία Κόμη θα μα στείλει την, το σχέδιο εκθεσή τη ω τα Χριστούγεννα, 22 Δεκεμβρίου. Χριστουγεννιάτικο δώρο για όλου μα. Θα τα συζητήσουμε στις 24-25 Ιανουαρίου. Έπειτα προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ως ε, ε, ε τις 7 Φεβρουαρίου, 28 και 29 θα τα εξετάσουμε ξανά στην Επιτροπή, 20 και 21 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και γύρω στο Μάιο στην Ολομέλεια. Εδώ ήδη έχουμε ξεκινήσει τις ε, συζητήσεις με την δανική κυβέρνηση που θα έχει τότε την Προεδρία και τα γνωρίζει όλα αυτά και η Πολωνική Προεδρία. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερω η Δανέζικη κυβέρνηση να επιτελεστεί πρόοδο εδώ. Και υπάρχει και ομάδα εργασία στο Συμβούλιο που εργάζεται παράλληλα με εμά. Ε, νομίζω λοιπόν το ντοσιά αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την όλη στρατηγική ανάπτυξη τη ε, Ευρώπη για το 2020 και για την ε, πράξη της ενιαίας αγοράς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η διεθνή αγορά καλύπτει πλέον πάρα πολλά θέματα. Τους πολίτες, την ασφάλεια των καταναλωτών, ε, τους εργαζομένους ε, και τις εταιρείες, τα πάντα. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους ιδιαίτερως. Με συγχωρείτε που σας βιάζω κάπως. Παρ' όλα αυτά μην ξεχνάμε ότι περάσαμε και στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ όσους μας άκουσαν και θα υπάρξει και στα αρχεία του site μας το ε, η ακρόαση αυτή, καθώς και αντίτυπα, χάρτινα αντίτυπα όλων των παρουσιάσεων που έγιναν, τα, μπορούμε, τα οποία μπορούμε να σας στείλουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν για τέλος όλους τους συμμετέχοντες. Κυρίσω τη λήξη της ακρόασης. Θα ξανασυνέλθουμε ως Επιτροπή στις 3 για δύο σημεία στο τακτικό μας πρόγραμμα εργασιών. Για τα οχήματα του γεωργικού και δοσοκομικού τομέα και την, ε, ε, το, το, το, το στην Ευρωπαϊκή